Um, Καλημέρα σας, συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη που έχει τεθεί από τους συντονιστές της ΛΥΠΕ κατόπιν του ψηφίσματος που θετήθηκε από το Κοινοβούλιο πέρσι τον Ιούλιο και ζητούσε από την Κομισιόν ε, να δώσει κατευθυντήριες γραμμές στα κράτη-μέλη για την αποφυγή της ποινικοποίησης της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, για την, σχετικά με την ε, οδηγία υποβοήθησης. Έχουμε λοιπόν ε, μια σχετική μελέτη και μπορούμε με τη μελέτη αυτή να υποστηρίξουμε τη συζήτησή μας ε, για την οδηγία υποβοήθησης. Το πρόβλημα είναι ότι η Κομισιόν μέχρι τώρα είπε ότι δεν σκοπεύει να προβεί στην κατάρτιση τέτοιων κατευθυντηρίων γραμμών στις 8 Μαρτίου είχαμε μία συνάντηση με ΜΚΟ, κάποιες ήσασταν και εσείς, ε, ε, ΜΚΟ που υλοποιούν επιχειρήσεις ε, έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο και νομίζω ότι όλοι αντιμετωπίσαμε την πραγματικότητα ότι κάποια κράτη-μέλη όχι μόνο αποδίδουν κατηγορίες σε άτομα που προσπαθούν να σώσουν τη ζωή άλλων ε, και υπάρχει και κατάσχεση πλοίων, αλλά χρησιμοποιούνται πολιτικά αυτά τα περιστατικά ή ως μέθοδος αποτροπής. Και νομίζω ότι όσοι ήσασταν εκεί στη συνεδρίαση αυτή καταλάβατε όλες τις συνέπειες. Τώρα εδώ συζητάμε το θέμα της οδηγίας ε, υποβοήθησης και είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή στο θέμα αυτό. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε και τα νέα ότι θα συνεχιστεί η επιχείρηση Σοφία χωρίς πλοία, δηλαδή δεν ε, θα είναι διαθέσιμες πλέον ε, οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης. Έτσι λοιπόν το κρίσιμο ερώτημα Τώρα, το ποιο θα υλοποιεί αυτές τις δραστηριότητε έρευνα και διάσωση ε, αντί της επιχείρηση Σοφία είναι αυτό που τίθεται. Αυτά όλα τα πολύ σοβαρά ζητήματα λαμβάνουν χώρα και θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ολοκληρώναμε τη θητεία χωρίς ε, να παρακολουθούμε και το θέμα αυτό έτσι λοιπόν, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων, ε, σήμερα έχουμε καλέσει μία εκπρόσωπο από μία ΜΚΟ που προφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πρόκειται για μια μαρτυρία της Μιλένα Ζάζοβιτς, είναι πρόεδρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Are You με Y γράφεται, και παρέχει αρρωγή στους πρόσφυγες που περνούν στην Κροατία. Καταρχήν θα ακούσουμε κάποιες παρεμβάσεις ε, και από την ε, Ευρωπαϊκή, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοροφικής και Εκτοφυλακής και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την οδηγία υποβοήθησης για το που βρισκόμαστε και γιατί η Κομισιόν μέχρι τώρα έχει αρνηθεί να καταρτήσει κατευθυντήριε γραμμέ για τα κράτη-μέλη για την οδηγία υποβοήθηση. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το που βρισκόμαστε σε σχέση με την οδηγία υποβοήθησης και θα θέσουμε απευθείας ε, μια ερώτηση στην Κομισιόν ε, που θα απαντηθεί από τον Μάικλ Σότερ. Γιατί λοιπόν δεν τα κάνετε αυτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα αποτελέσματα της κοινή ε, μεταναστευτικής μας προσέγγισης ε, για τη μετανάστευση είναι σαφή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει υποστήριξη και προστασία σε εκατομμύρια ανθρώπους, ε, σώζοντας πάρα πολλές ζωές στη θάλασσα, χιλιάδες ζωές στη θάλασσα και βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης. Επίσης, θέλει να προστατεύσει την παράτυπη μετανάστευση μέσω σημαντικού αγώνα καταπολέμησης ε, του δικτύου των διακινητών. Και πρέπει να συνεχιστεί αυτό το έργο γιατί είναι ασταθής η κατάσταση και οι διακινητές ε, συνεχώς αναζητούν νέες ευκαιρίες. Και καθώς ε, η εμπορία ανθρώπων ε, παραμένει χαμηλού κινδύνου ε, επιχείρηση και ιδιαίτερα κερδοφόρος, η οποία προσελκύει επαγγελματικές κλιματικές ομάδες. Το 2018 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιδιακίνησης Ανθρώπων στη Europol έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο, όπως και στο παρελθόν. Είχαμε, είχε πάνω από 100 τέτοιες υποθέσεις για διακίνηση ανθρώπων. Θα ήθελα να το αναφέρω αυτό γιατί σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνει η χώρα η σημερινή συζήτηση. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι η ποινικοποίηση της πραγματικής ανθρωπιστικής βοήθειας θα πρέπει να αποφευχθεί. Αυτή είναι η θέση της Κομισιόν, σαφέστατα. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποβοήθηση της παράνομης εισόδιέλευσης και διαμονής ε, δεν ε, απαιτεί από τα κράτη-μέλη να ποινικοποιούν μια τέτοια βοήθεια. Δεν είναι ο στόχος της νομοθεσίας αυτός. Και για να είμαστε σαφείς, η νομοθεσία παρέχει στα κράτη-μέλη ρητά μέσα να μην επιβάλλουν τέτοιες κυρώσεις. Όμως ε, φυσικά η Κομισιόν κατανοεί τις ανησυχίες σε αυτόν τον τομέα και το στενό ενδιαφέρον το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί το ζήτημα. Όντως, έχει αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, ε, δυνατότητα που υπάρχει να ποινικοποιηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια και γι' αυτό κάναμε μία αξιολόγηση της δέσμης μέτρων ε, το 2018. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν ε, για αυτή την αξιολόγηση κατά την ανάλυση κομισιών δεν επιτρέπουν ε, να έχουμε μία ξεκάθαρη εικόνα στο ότι υπάρχει επαναλαμβανόμενη καταδίκη και απόδοση κατηγορών κατά ατόμων και οργανώσεων που παρέχουν βοήθεια σε πρόσφυγες στα κράτη-μέλη ότι υπάρχει έλλειψη στοιχείων που να δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση και προς ε, την ανάγκη για νομοθετική αλλαγή. Όμως, αν ε, σκεφτούμε το πόσο μεγάλες είναι οι ανησυχίε σε αυτό το αντιλαμβανόμενο κίνδυνο ποινικοποίηση και τη σημασία του θέματος, φυσικά για τις συνεχιζόμενες εξελίξεις, ε, η Κομισιόν έχει δεσμευτεί για να συνομιλήσει με την κοινωνία των πολιτών και τα ενδιαφερόμενα μέρη για να συλλέξει περισσότερα στοιχεία και να ξεκινήσει ένα διάλογο για την εφαρμογή των εφιστάμενων κανόνων. Γι' αυτό έχουμε συνομιλήσει με κρυσόπους τη κοινωνία των πολιτών και με τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Μάιο του 2018 είχαμε μια ειδική συνάντηση στις Βρυξέλλες με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους οργανισμούς και ακολούθησε συζήτηση με τη Eurojust και τους εθνικούς εισαγγελείς πέρσι. Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τις επαφές αυτές με μία νέα συνάντηση φέτος την Άνοιξη για να εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα οποιοδήποτε αντίκτυπο σε ε, μέλη της κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης. Επίσης ε, και για το περιεχόμενο για το συγκεκριμένο project ε, ε, που έχει εφαρμόσει η Κομισιόν ε, μεταξύ των ε, αναπτυγμένων δικτύων των ενδιαφερομένων μερών για τη μετανάστευση που χρηματοδοτείται από την Κομισιόν από το πρόγραμμα Ορίζοντα 2020. Ο κύριο στόχο μα είναι να δημιουργήσουμε, να διατηρήσουμε ένα συνεχή διάλογο και ανταλλαγή με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την κατάσταση επιτόπου και σε σχέση με το πώ εξελίσσεται. Και πιο γενικά, Θέλω να υπογραμμίσω ότι δεσμεύεται η Κομισιόν να υποστηρίξει ισχυρέ ανεξάρτητε πλουραλιστικέ κοινωνίε των πολιτών στα κράτη-μέλη. Εντό των αρμοδιοτήτων που μας δίνει η συνθήκη η Κομισιόν θα συνεχίσει να διασφαλίσει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θεμελιώδη ελευθερία. σύμφωνα με το εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο και θα διατηρήσει το ρόλο και τη λειτουργία των οργανώσεων τη κοινωνία των πολιτών που προωθούν και διαφυλάσσουν τι ευρωπαϊκέ αξίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να πω ότι η Κομισιόν έχει παρακολουθήσει την κατάσταση και που το επιτρέπουν οι συνθήκες και βάσει συγκεκριμένη ανάλυσης. Παραδείγματο χάρη, όταν είχαμε διαδικασία, έχουμε διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ουγγαρίας σε ό,τι αφορά την νομοθεσία της που ποινικοποιεί δραστηριότητες που υποστηρίζουν ε, τους ετούντες ε, άσυλο και, περι, και περιορίζουν ε, την δυνατότητα ε, κατάθεση αίτηση ασύλου. Ανυπομονώ για τη συζήτηση που θα έχουμε σήμερα και σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Okay, thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχατε την ευκαιρία να τη διαβάσετε τη μελέτη μας αυτή. Μάλιστα. Ε, άλλος εδώ παρόν όχι. Για ποιο λόγο ε, το ε, λέγω. Διότι ακούσαμε να μας λέτε για τα στοιχεία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμής. Τι στοιχεία είναι αυτά. ποινικοποίηση των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών. Για μας ποιο είναι το ζήτημα. Ένα από τα όσα ανέκυψαν από τις συζητήσεις μας ήταν ε, η αποτρεπτική αυτή δράση και επίδραση ε, από μεμονωμένες διώξεις, μπορεί να μην είναι συστηματική. Και η μελέτη έδειξε ότι αυτό έχει μια ευρύτερη συνέπεια. Όταν μια μήκη όπου δραστηριοποιείται φέρει πέν στη Μεσόγειο ή κάποιες άλλες εταιρείε και οι ΜΚΟ που ασχολούνται με παροχή συμβουλών και υποστήριξη διώκονται ε, αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα που αποτρέπει πολλούς από το να βοηθήσουν. Και γι' αυτό ρωτώ, υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές, θα ρωτήσουν και άλλοι φαντάζομαι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει σοβαρά ότι υπάρχουν ε, έτσι αποχρώσεις ενδείξεις γιατί άμα έχουμε μια ολόκληρη λίστα με διώξει και εισαγγελίε, θα πρέπει να έχουμε κατευθυντήριε γραμμέ. Και για να βγει ε, αυτή η οδηγία, πρέπει να κατανοήσουμε πραγματικά το πόσο έτσι, έχει μουδιάσει η κοινότητα ε, των ανθρωπιστικών οργανώσεων από τις διώξεις αυτές και τη στάζει. Αυτή ήταν η δική μου ερώτηση. Φαντάζομαι θα έχουν και άλλοι συνάδελφοι ερωτήσεις. Ποιος έχει τώρα σειρά. Η Μπίργκετ Σίπελ Α, μάλλον πρέπει να ακούσουμε όλους τους ομιλητές πριν να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί ήθελα να την ανακρίνω εγώ και εγώ ήμουνα και ξέχασα τους υπόλοιπους ομιλητές. Η κυρία Σίπελ χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Um, Αλλά δεν θα τις ξεχάσουμε τις ερωτήσεις μας ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, Λοιπόν, η Άννα Κριστίνα ε, Ζόρζε τώρα ε, θα πάρει το λόγο. Είστε διευθύντρια στην αρμόδια επιχείρηση ε, της Ευρωπαϊκής Σύνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Παρακαλώ, πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλή σας μέρα και από πλευρά μου. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να σας ευχαριστήσω ε, για την πρόσκληση στο Frontex ε, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα που είναι τόσο περίπλοκο και τόσο σημαντικό. Στα πλαίσια της εντολής του, ο Frontex βοηθάει τις εθνικές αρχές ε, στην υλοποίηση της ε, οδηγίας ε, διευκόλυνσης με πολλούς τρόπους. Συχνά ε, οι αξιωματούχοι της Frontex είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με τα θύματα. Τα τελευταία χρόνια σώσαμε πάνω από 310.000 ανθρώπους και μόλις πέρυσι 37.000 μετανάστες σώθηκαν με τη βοήθεια του Frontex. Από την άλλη, μαζί με εθνικούς εταίρους όπως η Ευρωπόλ και Ευρωπαϊκούς, η Eurojust και η επιχείρηση Σοφία. Ε, ο οργανισμός μας διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταπολέμηση της διακίνησης μεταναστών. Ε, στόχος μας ε, είναι οι διακινητές και οι λαθρέμποροι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των μεταναστών. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση ε, της συμπόνιας και της βοήθειας προς τους μετανάστες με την καταπολέμηση των διακινητών. Όλα αυτά αναφέρονται διεξοδικά στον κανονισμό του Frontex για τον τρόπο λειτουργίας τους. Ορισμένες επιχειρήσεις διάσωσης επίσης είναι σημαντικό στοιχείο των επιχειρησιακών σχεδίων σε σχέση με τις επιχειρήσεις στη θάλασσα. Είναι σαφείς οι διαδικασίες που ισχύουν. Όλες οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όπου ενέχεται ο Frontex είναι υπό τον έλεγχο και ε, την ιεραρχία του κράτους μέλους που ε, μας υποδέχεται. Μετά ε, την ε, αποβίβαση ε, ελέγχει και ε, καταγράφει ο Frontex τους μετανάστες μαζί με τις αρμόδιες αρχές της χώρας άφηξης. Ο οργανισμός στη συνέχεια παραπέμπει τους μετανάστες στις αρμόδιες αρχές για την υποστήριξη που θα τους παρασχεθεί εκείνοι που θέλουν να ζητήσουν άσυλο παραπέμπονται στι υπηρεσίε ασύλου. Ενδεχόμενα θύματα τράφιγγιν παραπέμπονται στην αστυνομία που μπορεί ε, στη συνέχεια να του παραπέμψει σε διεθνείς και εθνικές ΜΚΟ για ε, υποστήριξη. Οι συνόδευτοι ανήλικοι παραπέμπονται στι αρχές προστασίας ανηλίκων, ενώ οι έγκυε ε, σε γιατρό για ιατρική εξέταση οι διεθνείς οργανισμοί όπως είναι η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία ε, του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και η Διεθνής Υπηρεσία Μετανάστευσης συμμετέχουν ε, όπως και πολλές διεθνείς και χώρες ΜΚΟ μεταξύ αυτών το Save the Children και ο Ερυθρός Σταυρός. Ωστόσο, ο Frontex μέσω των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης δεν έχει ως ρόλο να ε, ασχολείται με όσους φτάνουν. Από το 2011 ε, βοηθάει τα κράτη-μέλη και τις τρίτες χώρες για τη δημιουργία δυνατοτήτων με ε, εκπαίδευση προσωπικού για την καταπολέμηση του τράφικη και την προστασία των ανηλίκων στα σύνορα. Έχουμε αφιερώσει ένα ολόκληρο έργο για να βοηθούμε του συνοριοφύλακε, να προστατεύουν τους ανηλίκους ε, που είναι θύματα διακινητών. Η έρευνα και η διάσωση είναι σημαντικό στοιχείο της ολοκληρωμένης διαχείρισης φύλαξης των ε, ε, συνόρων, Frontex συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις αρμόδιες αρχές. Η συνεργασία αυτή γίνεται στα πλαίσια γενικών αρχών ε, του ευρωπαϊκού δικαίου όπως είναι η ε, εξουσίας, η επικουρικότητα και η ε, έντιμη και επίσης τη συνεργασία. Έχουμε διαρθρωμένο διάλογο μόνιμο με τις ΜΚΟ μέσω του Συμβουλευτικού μας Φόρουμ. Ως Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Frontex συμμετέχει στην πολιτική συζήτηση για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη διευκόλυνση. Η μεταφορά της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία βεβαίως είναι στα χέρια των κρατών μελών. Και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη της κάθε χώρας είναι εκείνη που θα αποφασίσει αν η διευκόλυνση έχει λάβει χώρα σε κάποιο συγκεκριμένο επεισόδιο. Τέλος, ε, θα ήθελα ωστόσο να υπογραμμίσω το γεγονός ότι όλοι μας και η Frontex και τα κράτη-μέλη και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και η ΜΚΟ έχουμε κοινό στόχο να βοηθούμε τα θύματα ε, κατά την άφηξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να συνεργαστούμε για να μειώσουμε τα επόμενα χρόνια τον αριθμό των θυμάτων αυτών. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα η Μιλένα από την ΜΚΟ Άριο Σύριος με ύψιλο από τη Συρία. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λέγομαι Μιλένα Ζάζοβιτς και είμαι πρόεδρος της Αργίου Σύριους, μία ΜΚΟ που, που έχει έδρα στην Κροατία και παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια, εφαρμόζει προγράμματα ένταξης και παρακολουθεί τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς επανειλημμένα ε, αναφέρουμε παράνομες επαναπροωθήσεις ε, που γίνονται από τους αστυνομικούς της Κροατίας. Έχουμε ε, επιβεβαιωθεί τα πορίσματά μας από την Υπεταρμοστία και άλλους διεθνείς οργανισμούς που έχουν δημοσιεύσει μαρτυρίες εκατοντάδων προσφύγων που, που αναφέρουν ότι παράνομα έχουν αποθηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε καταγράψει το 2018 ε, πάρα πολλές ε, αποθήσει και κανένας δεν θεωρήθηκε υπεύθυνο στην Κροατία. Ε, η Ματίνα Χουσεΐνη ήταν μία, ένα κοριτσάκι έξι χρονών που αποθήθηκε τον Νοέμβριο του 2017 και κατόπιν πέθανε. Μας περιέγραψαν ότι η οικογένειά της είχε οικετέψει για να μείνει και να ζητήσει άσυλο Όμω όμως οι αστυνομικοί τη διέταξαν να επιστρέψουν πίσω στη Σερβία και ε, μόλις ε, λίγα λεπτά αργότερα χτυπήθηκε από ένα τρένο το κοριτσάκι και πέθανε. Η Έργιο Σύριος ήταν η πρώτη που ενημέρωσε το κοινό για αυτή τη τραγωδία και έφερε το θέμα των αποθήσεων στα πρωτοσέλιδα των περισσότερων ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ε, όμως, αντί οι αρχές ε, και το Υπουργείο Εσωτερικών να απαντήσει για το ποιος ευθύνεται, αποφάσισε να επιβάλλει σιωπή ε, και η δική μας οργάνωση ήταν μία από αυτές που υπέστησαν τις συνέπειες. Ε, εγώ ε, θα ήθελα να σας δώσω τη μαρτυρία μου για το τι βιώνουμε εμείς ως παράδοξες συνέπειες του πλησίου. Λέω παράδοξες γιατί αυτή η οδηγία αποτυχαίνει για το σκοπό που έχει σχεδιαστεί. Ο σκοπός ε, ήταν να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση και να γίνει μια διάκριση ε, μεταξύ των παράνομων δραστηριοτήτων και της ανθρωπιστικής βοήθειας. Όμως ε, δημιουργεί κάποιο πλαίσιο όπου παράδοξα θίζουν οι παράνομες δραστηριότητες και στην πραγματικότητα αποτρέπεται η πραγματική βοήθεια του να ε, καταγγέλλεται η παράνομη μετανάστευση στις αρχές και οι εθελοντές ε, έχουν συνέπειες ε, όταν προσπαθούν να συνδέσουν τους μετανάστες με τις αρχές για να ασκήσουν τα νόμα δικαιώματά τους. Επίσης, παράδοξο γιατί πνίγονται οι άνθρωποι ή κατάσχονται τα πλοία ε, και δικάζονται οι άνθρωποι για εγκλήματα που δεν έχουν διαπράξει. Γι' αυτό χρειαζόμαστε εννοημόμορφες κατευθυντήρες γραμμές για όλα τα κράτη-μέλη για το τι μπορεί να θεωρηθεί ή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ε, υποβοήθηση της παράνομης εισόδου. Έχουμε αντιμετωπίσει καταστάσεις ε, ε, που δεν αφορούν μόνο τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων στην Κροατία, αλλά παντού στην Ευρώπη. Εκπρόσωποι δεκάδων ΜΚΟ θα μπορούσαν να καθόνται εδώ στη θέση μου σήμερα. Ε, η Jürgen Entretet, μια άλλη ευρωπαϊκή ΜΚΟ που έχει σώσει πάνω από 4.000 ζωές το 2016 και το 2017, ποινικοποιήθηκε από τους ίδιους ανθρώπους που καλούνται να καθίσουν εδώ μαζί μας σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ. Και πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να είμαι ξαφέστατη. Οι δικοί μας εθελοντές ε, δεν υποβοηθούν την παράνομη διέλευση στην πραγματικότητα, αν δεν μπορεί να αποδείξει ένα άνθρωπο ότι είναι σε ευρωπαϊκή επικράτεια, όταν ε, ε, έρθει σε επαφή για βοήθεια, λίγη η συζήτηση. Γιατί διαφορετικά θα μπορούσε να θεωρηθεί αυτό ενθάρρυνση. Κανένα δεν θυμάται την υπόθεση του κοριτσιού που πέθανε ε, λίγα λεπτά μετά την απόθεσή τη το Νοέμβριο του 2017. Ε, στα 20 Μαρτίου 2018 στη μέση τη νύχτα, ενώ είχαμε χιονοθύελα, πάλι η οικογένεια της μικρής ε, Ματίνα ήρθε σε επαφή μαζί μας και είπαν ότι ήταν πάλι στην Κροατία και ήταν τρομοκρατημένη για την πιθανότητα μιας ακόμη απόθεσης. Είχαμε 14 ανθρώπους στην ομάδα, 11 παιδιά και το μικρότερο ήταν μόνο ενός έτους και μα συγκέτευαν να του βοηθήσουν να ρυθμίσουν το νομικό, τους καθεστώς στην Κροατία. Του εξηγήσαμε ότι το μόνο που μπορούμε νομικά να κάνουμε ήταν ε, να επικοινωνήσουμε με την αστυνομία και να την ενημερώσουμε για την περιουσία της οικογένειας στην Κροατία και για το, ε, ε, το αίτημά τους ασύλου. Επιπρόσθετα σε αυτό, ε, ζητήσαμε από έναν θελοντή να πάει στη συνοριακή περιοχή και να ενημερώσει την τοπική αστυνομία για την πληροφορία που είχαμε για μια οικογένεια προσφύγων με 11 παιδιά που ε, ήταν μέσα στο κρύο ε, στην κροατική πλευρά. Ενημερώσαμε και το Υπουργείο Εσωτερικών για την παρουσία της οικογένειας και το γεγονός ότι ο θελοντής θα πήγαινε ε, στο σημείο ελέγχου για να αποφευχθεί παρεξήγηση και πριν από αυτό δύο φορές αποθήθηκε η οικογένεια. Έτσι λοιπόν πιστεύαμε ότι η παρουσία του εθελοντή μας ήταν ο μόνος παράγοντας που θα απέφευγε την τρίτη απόθεση της οικογένειας εκείνη τη νύχτα και φαίνεται ότι το να έχουν επανέλθει στην κρατία και να μπορούν να καταθέσουν για το θάνατο του κοριτσιού ε, θύμωσε κάποιον στο Υπουργείο. Δύο εβδομάδες μετά το Υπουργείο ε, απήγγειλε κατηγορίες κατά ενός μέλου μα ότι είχε υποβοηθήσει την παράνομη εισόδου και επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ και ποινή φυλάκιση. Ε, και μόνο το πρόστιμο θα μα έκλεινε για πάντα. Είναι αδύνατον ένα άνθρωπο να πληρώσει κάτι τέτοιο στο δικαστήριο. Αποδείξαμε ότι η οικογένεια ήδη βρισκόταν στην Κροατία όταν είχε έρθει σε επαφή μαζί μα. Επομένω, δεν υπήρχε διέλευση συνόρου. Το αναγνώρισε ο δικαστή ότι δεν είχε άμεση επικοινωνία θελοντή με την οικογένεια, μόνο με του αστυνομικού και ότι δεν είχε καμία πρόθεση συμφέρον να υποβοηθήσει παράνομη δραστηριότητα. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε ένοχος ε, για αμέλεια και το δικαστήριο είπε ότι θα έπρεπε ε, να σκεφτεί ότι ίσω η οικογένεια δεν ήταν στην Κροατία, ακόμη και αν ήταν, ε, και ε, μα το είχαν επιβεβαιώσει γιατί μα έστειλαν την τοποθεσία του με το GPS. Αυτή η ακροβατσία επέτρεψε στο Υπουργείο Εσωτερικών να μα απαξιώσει στα μάτια του κοινού, συνδέοντα τη δουλειά μα με παράνομη δραστηριότητα και δεν χρειάστηκε να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσει για παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποθήσει. Να όμως δεν σταμάτησαν ε, εκεί. Το Υπουργείο επίσης είχε ξεκινήσει την ε, δραστηριότητα δυσφήμισης κατά της οικογένειας του κοριτσιού και των δικηγόρων τους ε, η οικογένεια τέθηκε υποκράτηση και της αρνήθηκαν πρόσβαση σε δικηγόρο και ο συνήγορος του πολίτη της Κροατής είπε ότι σχετικές πληροφορίες ε, για την υπόθεση αυτή, ακόμη και εικόνες από κάμερα, είχαν διαγραφεί από τους αστυνομικούς και το Υπουργείο έκανε τα πάντα για να σαμποτάρει την έρευνα. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι πρόσφυγε είχαν σε επαφή με τη δική μα ΜΚΟ. Κάποιοι κάλεσαν στα γραφεία μα ε, στο Ζάγκρεπ, κάποιοι έστειλαν τι αποθεσίε GPS για να, για να δείξουν ότι είναι στην κρατία και να ζητήσουν νομική υποστήριξη. Όλοι ζητούσαν βοήθεια στο να ρυθμίσουν ε, το νομικό του καθεστώ στην Κροατία, στο να έρθουν σε επαφή με την αστυνομία, όχι να διαφύγουν. Αλλά φοβούνταν τι αποθήσει ε, αν έρχονταν σε επαφή με την αστυνομία μόνοι του. Κάποιοι, όπως η οικογένεια της μικρής Ινάς, είχαν βιώσει στο παρελθόν τις αποθήσεις. Για όλους κάναμε τα ίδια, τους ε, οδηγήσαμε στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσουν άσυλο. Και κατόπιν οι εθελοντέ μα πήγαν στο ίδιο αστυνομικό τμήμα για να ελέγξουν αν είχαν γίνει σεβαστά τα δικαιώματά του. Όμω σε τέτοιε περιπτώσει οι εθελοντέ συχνά κρατούνταν χωρί εξήγηση στο αστυνομικό τμήμα για πάνω από 8 ή 10 ώρε και η αστυνομία τους απειλούσε λέγοντας ότι θα τους απήγγειλαν κατηγορίες αν συνέχισαν να παρακολουθούν τις διαδικασίες ε, χορήγηση Σύλλου και είχαμε και μια συνέντευξη τύπου για να θίξουμε αυτό το θέμα μαζί και με άλλες ΜΚΟ που ήταν στο στόχαστρο και πήγαν οι αστυνομικοί ε, στα σπίτια των ανθρώπων που πρόκειται να μιλήσουν ε, στην συνέντευξη τύπου και κλήθηκαν όλοι σε ανάκριση ακριβώς την ίδια ώρα που είχαμε κανονίσει τη συνέντευξη τύπου. Αυτό προκειμένου να κάνουν τις ΜΚΟ να σιωπάσουν. Ε, τέτοιες ε, διαδικασίες ε, δυσφήμισης και δίωξης γίνονται όλο ένα και περισσότερο απέναντι στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα. Γι' αυτό ζητάμε κατευθυντήριες γραμμές κοινέ για όλα τα κρατημέλη για το τι μπορεί να θεωρηθεί ή όχι ως υποβοήθηση παράνομης εισόδου διέλευσης και διαμονής λαμβάνουμε υπόψη ε, την κατάσταση και ε, συγκεκριμένα παραδείγματα ποινικοποίηση που σας παρουσίασα. Αν η Κομισιόν ε, δεν ξεκαθαρίσει τις οδηγίες, μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά των ΜΚΟ και πολιτών που τηρούν τον νόμο. Χωρί ανθρωπιστική βοήθεια και διάσωση στη θάλασσα, θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο στάφος η Μεσόγειο. Χωρί κανένα να παρακολουθεί στην πρόσβαση στι διαδικασίε ασύλου, χιλιάδε νέα θύματα θα ε, αποθούνταν εκτό Ευρώπη στα χέρια των διακινητών. Για μένα ως Ευρωπαίο πολίτη είναι απαράδεκτο αυτό και ελπίζω να είναι απαράδεκτο για όλου στην αίθουσα σήμερα. Για να καταλήξω, τα Ηνωμένα Έθνη για καλούς λόγου έχουν ε, ε, μια διακήρυξη για την προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα και η Κομισιόν πρέπει να προστατεύσει του υπερσπαστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κάνουν τη δουλειά του χωρί να φοβούνται την ποινικοποίηση. Αντί να δώσει ξεκάθαρε οδηγίε στα κράτη-μέλη για το τι κάνουν ε, με τους νεροφύλακες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, πρέπει να αναγνωρίσουν την κατάσταση, να αποτρέψουν νέες τραγωδίες και αν δεν μπορείτε να το κάνετε να μου το πείτε. Να πείτε τι θα κάνατε αν ήσασταν στη δική μου θέση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να εγγυθώ την νομική ασφάλεια στους εθελοντές μας, αν και τα κάνουν όλα με το γράμμα του νόμου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και πάμε μέσω στους συναδέλφους η Μπέρκη Τσίπελ πρώτη στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το εξή είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Θα πρέπει να καταπολεμούμε του εγκληματίε όπου και να βρίσκονται αυτοί. Μπορείτε όμω να μα δώσετε κάποια αριθμητικά στοιχεία για τι δραστηριότητε ε, διακινητών αυξήθηκαν ε, οι αριθμοί αυτοί αντίστοιχα και ταυτόχρονα ε, με τις δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης που δυσκολεύουν ε, την έλευση ε, των μεταναστών. Βγάζουμε, χτίζουμε φράχτες παντού. Στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, στο Καλέ, στη Θέοτα, στη Μελίγια και μετά ερχόμαστε και απορούμε. Μα πώς δεν μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη και καταφεύγουν σε διακινητές. Αφού δεν μπορούν να έρθουν. Δηλαδή προσπαθούμε να αποτρέψουμε την είσοδο κάποιων ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απλώς και μόνο επειδή χρησιμοποιούν την ε, βοήθεια των διακινητών. πιστεύετε ότι δεν έχουν λόγο αυτοί να ζητήσουν άσυλο. Προσπαθούμε να ποινικοποιήσουμε τους ανθρώπους ε, που βοηθούν κάποιους άλλους ανθρώπους που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να πεθάνουν ή να πνιγούν στη Μεσόγειο. Κατάσχουμε τα πλοία, ποινικοποιούμε τον κόσμο όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά και αλλού από ό,τι ακούμε. Είναι λύση αυτό το θέμα, αυτό που θέλουμε, ε, τι είναι να δυσκολεύουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, αν κάποιο καταλάβει ότι μπορεί να ε, το επιβληθεί ποινή φυλάξη μέχρι και 20 ετών, ποιο θα πάει να, να βοηθήσει μετά εκείνον που κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Δεν μιλούμε για ποινικοποίηση. Ε, αποτρέπουμε και εμποδίζουμε τους ανθρώπους να βοηθούν. Μα το να βοηθά του ανθρώπου και να σώζει ανθρώπου δεν είναι απλώ ευρωπαϊκή, ε, διεθνή ή ανθρωπιστική υποχρέωση. Είναι τελείως απαράδεκτα και παράνομα αυτά που κάνουν οι Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Έχει περιέλθει η γνώση σα. τι γίνεται με τους λεγόμενους παράτυπους μετανάστες στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι πολλοί παραμένουν στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι πολλοί εργάζονται στην Ευρώπη. Και ορισμένοι δεν καταγράφονται ποτέ. Εσείς κυνηγάτε και ελέγχετε και τους εργοδότες που εκμεταλλεύονται και απασχολούν παράνομα παράτυπους μετανάστες. Πολλά είναι τα ερωτηματικά και νομίζω είναι πραγματικά λυπηρό η Ήπειρός μας να λέει πάντα για να δικηρύσει ότι είναι Ήπειρος των δικαιωμάτων της δημοκρατίας και των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων και μετά κάνουμε τα μάτια. Και συνεργαζόμαστε και με τη Λιβική ε, ε, ε, ακτοφυλακή. Και θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, εάν η ε, ε, Λιβική ακτοφυλακή εμποδίζει τους μετανάστες να έρθουν στην Ευρώπη και τους επιστρέφουν στις ακτές, ε, μετά τι γίνεται. Ε, μας λέτε ότι τους ελέγχετε. Πού τους ελέγχετε. Ελέγχετε την ακτοφυλακή στα σκάφη. Μετά τι γίνεται στους καταβλισμούς. Ε, γιατί υπάρχουν καταγγελίες για βίες επιθέσεις, για βασανιστήρια κτλ και βίαιε αποθήσει που παράνομε είναι και αυτέ. Και θα ήθελα πραγματικά να ξέρω τι κάνει η Frontex και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριμένα. Υποστηρίζουμε τις ΜΚΟ που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά που όλο και περισσότερο δεν κάνουν τα κράτη-μέλη μας. Σταματάει η επιχείρηση Σοφία τώρα. Και τι γίνεται με την επιτήρηση της Μεσογείου με πλοία ή με ρομπότ. Ωραία, για να μετράμε τους νεκρούς και τους πνιγμένους. Τι άλλο θα κάνουμε. Και ποια είναι τα επόμενα βήματα και πώς μπορούμε να αποφύγουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή να γίνεται όλο και περισσότερο μια ένωση όπου ε, δεν είναι πια σεβαστές οι αξίες. Η, Ανα... η Μπάρμπαρα Σπινέλη, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, και για τους τρεις ομιλητές για τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Δεν θέλω να πω καταρχήν ότι το πρόβλημα δεν ε, είναι εδώ η αγωνία του Κοινοβουλίου, αλλά είναι η αγωνία των ανθρώπων που είναι στα κέντρα κράτησης, ε, στη, στο λιβικό έδαφος. Και ασχολούμαστε με αυτό γιατί η Μεσόγειος έχει αδειάσει από πλοία παροχής βοήθειας, γιατί η επιχείρηση Σοφία δεν ασχολείται πλέον, δεν έχει πλέον πλοία, αλλά μόνο αναγνωριστικά αεροσκάφη και προσωπικό για κατάρτιση της Λιβικής Οκτωφυλακής και γιατί οι ΜΚΟ έχουν εκδιωχθεί από τη Μεσόγειο. Εσείς μας είπατε επίσης ότι λείπουν αποδείξεις ποινικοποίησης ε, των μελών των ΜΚΟ. Έχουμε πάρα πολλές αποδείξεις και εσείς τις έχετε. Δεν ξέρω τι περιμένετε ακόμα. Στο πλαίσιο αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μιλένα Σταγιόβιτς για την δραστηριότητά της και για τις αποδείξεις που μας παρουσιάζει σε σχέση με την πολιτική των αποθήσεων που ασκεί η Κροατία. προς τη Βοσνία και τη Σερβία. Θα ήθελα επίσης να ξέρω σχετικά με το θάνατο του κοριτσιού από το Αφγανιστάν. Έχει πάει αυτή η υπόθεση ε, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Να ήθελα να μου πείτε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Και τέλος, θέλω να απευθυνθώ στην Άννα Κριστίνα από τη Frontex. για να μιλήσω για δικήματα. Για κατηγορίες που πολλαπλασιάζονται κατά τον ΜΚΟ με νέα είδη αδικημάτων. Όπως ε, παραδείγματο χάρη έχουμε το θέμα της διακίνησης που είναι παλιό. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος αδικήματος στο οποίο συζητείται πολύ στην ετηλική κυβέρνηση της ε, θαλάσσιας πειρατείας. Το εμπορικό πλοίο που έφτασε πρόσφατα στη Μάλτα Οι άνθρωποι εκεί κατηγορήθηκαν ότι διευκόλυναν μορφή θαλάσσιας πειρατείας γιατί οι μετανάστες που διασώθηκαν αντί να οδηγηθούν στη Λιβύη απείλησαν να πέσουν στη θάλασσα και άλλαξαν την πορεία του πλοίου. Κατηγορήθηκαν γι' αυτό, όμως δεν είναι αλήθεια. Απλώς απειλήσαν ότι θα ξαναπέσουν στη θάλασσα. Ένα άλλο είδος αδικήματος, πραγματικά πρωτότυπο, είναι το εξής, οι δράσεις της έρευνας και διάσωσης απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνες που γίνονται στην Ιταλία. Γιατί μιλάμε για γιότ και όχι για σκάφη παροχής βοηθείας. Είναι απίστευτη η ποσότητα των αδικημάτων που εφευρίσκουν για να εξαλείψουν από τη Μεσόγειο όλες τις ΜΚΟ αφού κατήργησαν και την επιχείρηση Σοφία. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μόνο η Λιβική εκτοφυλακή δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο. Και τέλος, μια ερώτηση στην Άννα Κριστίνα Γιώργη από τη Frontex. Εσείς ξέρετε ότι υπήρξε τις προηγούμενες μέρες μια επιστολή από τη Διευθύντρια της ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΧΟΜ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου νομιμοποιούνται οι ακτοφυλακές της Λιβύης. Πρόκειται για μια επιστολή που συμπεριέλαβε η Ιταλική κυβέρνηση σε μια οδηγία για κλείσιμο των Ιταλικών λιμένων. Αυτή η επιστολή ε, Στάλι στο Φαμπρίζ Λετζέρι. Αυτό που σας ρωτώ είναι το εξής. Να σας ζητώ να μας δώσετε το γράμμα που έγραψε ο Λετζέρι στην Κομισιόν γιατί πιθανότατα εξέπρασε αφιβολίες ή διατύπωσε ερωτήσεις στις οποίες η Κομισιόν απάντησε με μια επιστολή που φαίνεται να έχει γραφεί από τον Υπουργό Σαλβίνη. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ. Έχουμε και άλλα θέματα. Θα σας παρακαλούσα να είστε λίγο πιο σύντομοι. Η Άννα Γκόμες, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Ε, ε, είναι ανέκδοτο η Λιβική ακτοφυλακή. Εμείς την έχουμε εφεύρει. Όποιος γνωρίζει τη Λιβύη και πώς λειτουργεί η Λιβύη, η Λιβική ακτοφυλακή είναι μια πολιτοφυλακή που έχει αλλάξει όνομα. Και οι άνθρωποι ε, και λαθρέμποροι είναι και βασανιστές και λεφτά βγάζουν από τους μετανάστες και με διάφορες μαφίες συνεργάζονται ανά την Ευρώπη. Είναι εξωφρενικό που οι ευρωπαϊκές αρχές εξακολουθούν να μιλούν για λιβική ακτοφυλακή παραγνωρίζοντας ή αγνοώντας αυτή την πραγματικότητα. <coughs> με βγάζει από τα ρούχα μου πραγματικά. Γιατί καταλαβαίνω ότι Πού είναι το ανθρωπιστικό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά παραβιάζονται κατάφορα από εκείνους που ειναι το ανθρωπιστικο δικαιο το διεθνες δικαιο το διεθνες δικαιο της θαλασσας ολα αυτα παραβιαζονται καταφορα απο εκεινου που ειναι στι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ε, ε, κυνηγάνε τις ΜΚΟ που σώζουν ζωές, είτε στη θάλασσα είτε στη στεριά και τους καταγγέλουν. Και μάλιστα και όσους καταγγέλουν και καταπολεμούν τις αποθήσεις αυτές, όπως μας εξήγησε ε, η κυρία από την Κροατία την οποία πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω για το έργο που κάνουν. Τι κάνουν λοιπόν εκεί. Κάνουν πολύ καλή δουλειά, την ηθική δουλειά, την ανθρωπιστική, τη σωστή δουλειά των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εκείνοι προσπαθούν που να τους ε, ποινικοποιήσουν είναι φασίστες. Και αν δεν το βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι κάνει τέλο πάντων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ε, συγγνώμη κύριε Σούτερα, αλλά αυτά που μα παρουσιάσατε, α, θα πρέπει λέει να αποφεύγεται η ποινικοποίηση. Α το καλό. Ε, τι είναι αυτή η απάντηση με υπεκφυγέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίθεται ότι είναι θεματοφύλακας των ε, συνθήκων που θα πρέπει να στριμώχνουν τα κράτη-μέλη ε, να κάνουν αποθήσει και ποινικοποιούν τι ΜΚΟ. Αυτοί είναι οι εγκληματίε. Οι κυβερνήσει, σαν φασιστική κυβέρνηση του Σαλβίνη ή αυτό που κάνουν εκεί πέρα στην Κροατία αυτά που κάνουν και άλλες κυβερνήσεις. Αυτές θα πρέπει να κατηγορούνται και να ποινικοποιούνται γιατί δεν εφαρμόζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας λοιπά Και κατά τα άλλα, αυτοί είναι επίσης εκείνοι που επιτρέπουν στους διακινητές να λειτουργούν και να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί ακριβώς επειδή δεν ανοίγουμε ασφαλείς δρόμους ε, ε, για ε, τούντες άσυλο και μετανάστες, δίνουν δουλειά στους διακινητές. Δεν έχει άλλη εναλλακτική λύση ο κόσμος και νόμιμη οδό παρά να βάλει τη ζωή του στα χέρια των λαθρεμπόρων. Αυτοί θα πρέπει να πενικοποιούνται Και εγώ ως Πορτογαλίδα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τη δουλειά που κάνουν οι Πορτογάλοι στο Frontex και σώζουν και ζωές. Και δεν θα δεχόμουν ποτέ να πάει Πορτογάλος στο Frontex αν η πρώτη του υποχρέωση δεν ήταν να σώζει ζωές. Αυτή είναι η πρώτη υποχρέωση όλων μας και πραγματικά είμαι έξω φρενών που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς να το πω τώρα, ακολουθεί αυτή την τρομακτική γραμμή που μόλις μας παρουσιάσατε. Και επειδή φεύγω από το κοινοβούλιο και ελπίζω σύντομα να πάω κι εγώ στη Μεσόγειο να σώσω ζωές με τις ΜΚΙΟ. Πρόεδρο, ε, αυτά που είπε ο κύριο ε, Σπινέλη σχετικά με την επιστολή, η κυρία Σπινέλη με συγχωρείτε, ε, Είναι μια επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Frontex 18 Μαρτίου και ε, επειδή δεν έχουμε αυτή την επιστολή, με πάση περιπτώσει αναφέρεται ε, σχετικά με την ε, ακτοφυλακή και την περίπτωση της Λιβύης. Θα αυτά περίπου αναφέρει η επιστολή. Θα δω κατά πόσο μπορούμε να δούμε αυτή την επιστολή, γιατί υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα. Αλλά θέλω να σας πω ότι θα το θίξω το θέμα όταν θα έρθει αργότερα ο Επίτροπος ή Μάλεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω το εξής. Ε, το πρώτο συστημικό πρόβλημα είναι εδώ το γεγονός ότι το να διασχίσει κανείς ε, παράνομα τα σύνορα, αυτό δεν είναι το μόνο που μπορεί να κάνει κανείς. τη στιγμή που δεν υπάρχουν ε, νόμιμες δυνατότητες, είναι ένα συστημικό πρόβλημα που σημαίνει ότι όσοι διευκολύνουν σε εισαγωγικά, κατ' ουσίαν σώζουν ζωές. Ε, πώς αλλιώς να έρθουν οι άνθρωποι. Όταν ε, διευκολύνει κανείς που έτσι κι αλλιώς είναι παράνομο, ναι, το κάνεις αυτό γιατί σώζει ζωές. Περί αυτού πρόκειται και γι' αυτό αυτή η οδηγία είναι ε, λάθος από την αρχή γιατί δεν υπάρχουν ε, ασφαλείς ε, τρόποι διέλευσης. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι αρκετά προκλητικό το να ακούει κανείς την Κομισιόν και την Frontex. Η Κομισιόν λέει η ποινικοποίηση της καθαρά ανθρωπιστικής βοήθειας θα έπρεπε να αποφεύγεται. Τι σημαίνει αυτό το θα έπρεπε να απαγορεύεται διαρροπάλου. Ε, σε τελική ανάλυση ε, όταν ακούμε τέτοια πράγματα και ακούμε ε, τους εθελοντές που μπαίνουν, τους βάζουν στη φυλακή, που τους επιβάλλονται πρόστιμα που δεν μπορούν να πληρώσουν, σε τελική ανάλυση τι είδου Ευρώπη εσείς υπερασπίζεστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, νομίζω ότι είναι συνένοχος ε, και ως εκ τούτου ε, θεωρώ ότι το να βάζει κανείς τη ζωή ανθρώπων σε κίνδυνο αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ε, και που μας είπατε την ιστορία της Μιλένα και της οικογένειάς της ε, γιατί με τον τρόπο αυτό έχουμε και ένα στοιχείο πραγματικότητας μέσα σε αυτή την αίθουσα κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην ε, απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Frontex. Και θέλω επίσης να πω το εξή. Έχετε ένα έγγραφο και το είπατε και στην παρουσίασή σας ότι έχουμε 7.000 ε, παράνομες επιστροφές, ε, παναπροωθήσεις. Αυτό θα έπρεπε να εξοργήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Frontex για την παραβίαση του ε, διεθνούς δικαίου. Έχουμε ΜΚΟ και ως εκ τούτου ε, καταλαβαίνετε ότι με τον τρόπο αυτό παραβιάζουν το διεθνές ε, και το ενωσιακό δίκαιο. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε και σε αυτή την αίθουσα και εκτός αυτής. Μερικοί από εμά έχουμε συντάξει μια επιστολή και τα αναφέρουμε όλα αυτά, τις 7.000 επαναπροωθήσεις, ε, η χρηματοδότηση της κουρατείας ε, και αυτό τίθεται και γι' αυτό και εμείς ζητάμε ε, άμεση δράση γιατί κάπως πρέπει να λυθεί το όλο θέμα το ερώτημα που έβαλε είναι πώς ακριβώς ε, μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Και κατά τα άλλα θέλω να ακούσω από σένα Μιλένα να μας πεις ε, τι ε, γιατί ακούω τι δουλειά κάνεις, άκουσα το έτοιμά σου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας πείτε τι είδους υποστήριξη χρειάζεστε, ε, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι ΜΚΟ, αλλά θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς χρειάζεστε από εμάς. Γιατί κατ' ουσίαν παραβιάζεται το δίκαιο, αλλά παραβιάζονται και βασικές ανθρωπιστικές αρχές. Ε, ως εκ τούτου, εγώ θα ήθελα να γνωρίζω τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για να επιδείξουμε αλληλεγγύη στη δουλειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, μιλητές που είναι εδώ σήμερα και ευχαριστώ και την ε, Μιλένα και την Αργιού Σύριους. Γνωρίζω την ιστορία της και ευχαριστώ που μας καταθέτει αυτή την ξεκάθαρη και σημαντική μαρτυρία για το τι συμβαίνει δυστυχώς σε όλη την Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι παράλογη η συζήτηση αυτή, αυτή η ποινικοποίηση των ΜΚΟ, που ε, ουσιαστικά απλώ καλύπτουν μια τεράστια θεσμική ε, απουσία. Και δεν μιλάω μόνο για την ε, Μεσογειακή Οδό. Πολλοί συνάδελφοι έχουμε ζητήσει πραγματική ευρωπαϊκή αποστολή έρευνα και διάσωση στη Μεσόγειο αν ήμασταν συνεπείς για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων που θέσαμε, ε, ιδρύοντας την Ένωση θα έπρεπε να κάνουμε αυτό και να σώζουμε τις ζωές στη θάλασσα. Και για την Βαλκανική Οδό που σε πολλούς αρέσει να λένε ότι έχει κλείσει, θα ήθελα να υπενθυμίσω την κατάσταση που έχουμε στα σύνορα Βοσνίας Ερζεγοβίνης και Κροατίας, όπου χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε απελπισμένες, απάνθρωπες συνθήκες, χωρίς καμία πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, σε νομική αρρωγή. Επομένως, πράγματι πρέπει να αναρωτηθούμε αν βλέπετε τι συμβαίνει και η απάντηση δεν ε, μπορεί παρά να είναι ναι. Τα γνωρίζετε όλα απόλυτα. Γιατί υπάρχουν ε, το χάρη και η Βοσνία έχει λάβει πολλά εκατομμύρια ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για να προσφέρει ελάχιστες συνθήκες αξιοπρέπειας υποδοχής στους ετούντες άσυλο και δεν κατανοούμε πώς η Κομισιόν παρακολουθεί την πραγματική χρήση αυτών των πόρων, των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Εγώ συνεχώς λαμβάνω παραπάνω υλικό, τεκμηριωμένο, βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν ποιε είναι οι συστηματικέ παραβιάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων από τι αρχέ τη Κροατία και σε σχέση με την παραβίαση της αρχής της ε, μη ε, συλλογικής ε, επαναπροώθησης. Είχαμε και κοινοβουλευτική ε, περώτηση με 20 συναδέλφους πώς η Κομισιόν σκόπευε να διερευνήσει τις συστηματικές καταγγελίες ε, για τις παραβιάσεις. Ε, μιλάμε για κλοπές και παρενοχλήσεις των ανθρώπων από τις κρατικές αρχές. Χρειάστηκαν πέντε μήνες για να έχουμε απάντηση από την Κομισιόν. Γιατί χρειάστηκαν πέντε μήνες. Και επίσης ρωτήσαμε αν η Frontex ήταν παρούσα στα σύνορα αυτά για να μπορεί να παρακολουθήσει παρακολουθεί τι συμβαίνει. Ορίστε, στην ε, καθυστερημένη απάντηση της Κομισιόν υπήρχε δέσμευση να επαληθεύσει τις σοβαρές κατηγορίες κατά κρατικών αρχών και θα ήθελα να μου πείτε τι κάνετε. Η ποινικοποίηση μπροστά στα μάτια όλων δεν είναι μόνο στην Αριού ε, Σύριο, στο Σπιτερίβο, στην Εβέντα, στην Προακτίβα, στην Open Arms, στη Sea-Watch και σε άλλες κυβερνητικές οργανώσεις θα έλεγα ότι αυτή η ποινικοποίηση θέλει να εκφοβήσει και αυτό είναι απαράδεκτο. Τώρα για την οδηγία περί υποβοήθησης θα έπρεπε να αλλάξουμε και να καταστήσουμε υποχρεωτική τη ρήτρα για την ανθρωπιστική βοήθεια αν και με πόνο το λέω η ρήτρα είναι υποχρεωτική στην Ιταλία δυστυχώς δεν βλέπουμε τα αποτελέσματα και αυτή η συνεχής ποινικοποίηση όχι μόνο από την πλευρά της κυβέρνησης ε, αλλά και από ένα μέρος των δικαστικών αρχών συνεχίζει να υφίσταται και φαίνεται να ασκούν διώξεις ε, κατά οποιοδήποτε είδους αδικήματος αν και έτσι περισσότερες περιπτώσεις είναι άκαρπες οι διώξεις αυτές θα ήθελα να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτή τη θητεία με κάπως πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Υπάρχει ένα παράδοξο νομικό εδώ, ε, το ότι ε, η Κομισιόν ε, να μην θεωρείται ότι η Λιβύη είναι ασφαλής λιμένας. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να στέλνουμε ευρωπαϊκούς πόρους στη Λιβυκή Ακτοφυλακή που παραβιάζει συνεχώς τα θεμελιώδη δικαιώματα και ξέρουμε ότι ξαναστέλνει του ε, ανθρώπου ε, στις ε, φυλακές της Λιβύης που είναι πραγματική κόλαση. Θέλουμε ότι μας αξίζει, θεωρούμε ότι μας αξίζουν πιο ξεκάθαρε απαντήσει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Να, καλή τύχη. Ο κύριος Γιούρεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι αν Υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα εδώ, η κοινωνική σκοπιμότητα. Αυτό που πρέπει να μας απασχολεί δεν είναι η νομοθεσία. Γιατί αυτό είναι ο λαϊκισμός που υποτίθεται ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε. Αυτή είναι μια απαρχιωμένη αντίληψη για την πολιτική. Για να αντιμετωπίσουμε τους αντιπάλους μας και αν θεωρούμε ότι εμείς έχουμε δίκιο, θα πρέπει πάντα να τηρούμε το δίκαιο. Το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού και μιλώ για ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα λοιπά. Τώρα έφυγε η κυρία Αναγκόμες, έχει αποχωρήσει, αλλά μόλις ε, κατηγόρησε διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι είναι φασιστικές. Είναι βαριά κουβέντα αυτή και πολύ ενδεικτική. Διότι κατηγόρησε και την κροατική κυβέρνηση του κυρίου Πλάνκοβιτς, που ήταν πρώην συνάδελφός μας. Οι χώρες μας ε, είναι δημοκρατικές και υπάρχει και το άρθρο 7 στη συνθήκη και κανείς δεν έχει θεωρηθεί ε, ένοχος ως μη δημοκράτης. Όλα τα υπόλοιπα είναι γνώμες, προσωπικές και τίποτα άλλο, προσωπικές απόψεις που μπορεί ο καθένας να έχει τις δικές του. Ε, ε, άρα, θα πρέπει να αντιδράσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, σε τέτοιες επιθετικές ε, δηλώσεις. Και υποθέτω ότι ο, Κλοντ Μωράες δεν πρόκειται να αντιδράσει, διότι από ό,τι φαίνεται ε, η πλειοψηφία στην Επιτροπή μας εδώ κυβερνάει τη μειοψηφία. Αλλά επικαλούμε το άρθρο 11 του κανονισμού δεν ε, ε, μπορούμε να ανεχθούμε αυτή τη δήλωση της κυρίας Γκόμες, αλλιώς δεν τηρούμε τον ίδιο μας ε, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πραγματικά είναι φαύλος κύκλος αυτό. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και δύσκολα και πολλαπλασιάζονται συνεχώς. τα περιστατικά με τους μετανάστες. Και καμιά φορά είναι δύσκολο να παράσχει κανείς ανθρωπιστική βοήθεια. Και είναι δύσκολο να αντιδράσεις, ακόμα και αν έχεις ε, ανθρωπιστικά κινήτρα. Εγώ είμαι υπέρ του κράτους δικαίου φυσικά, αλλά και υπέρ του κράτους του κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Χόλμα, η τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ ε, που μπορώ να μιλήσω έστω και για δύο λεπτά. Εγώ προσωπικά πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι από τους ε, σοσιαλδημοκράτες, ε, το να απευθύνει κανείς ε, συλλήβδιν αιτιάσεις κατά της κροατικής κυβέρνησης ή οποιασδήποτε άλλη κυβέρνηση, αυτό δεν είναι σωστό. Και εγώ ξέρω τι συμβαίνει στην Κροατία και γνωρίζω ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Γιατί υπάρχουν χώρες οι οποίες απλά προωθούν τις επαναπροωθήσεις, η Ιταλία παραδείγματος χάρη, επαναπροωθούν τους ανθρώπους σε άλλες χώρες οι οποίοι ε, πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και χαίρομαι πάρα πολύ, ε, λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι ε, δεν μπορεί κανείς να επαναπροωθήσει από ανθρώπους από τρίτες χώρες σε άλλες χώρες. Δηλαδή αυτοί που βρίσκονται στη Σερβία και που η ε, SD θα ήθελε να παραμείνουν εκεί ε, αυτοί, ε, εφόσον παραμένουν, αυτό είναι δική τους ευθύνη. Εάν μπορούσε να παρέμει η Frontex, τα πράγματα θα γινόντουσαν με κάποιους κανόνες ε, και μόνο με βάση νομικές αποφάσεις. Γι' αυτό λοιπόν την απόφαση που θα λάβουμε τη θεωρώ λανθασμένη, γιατί διότι δεν θα συμβάλλουμε έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να έχουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτοί δεν ετούνται άσυλο και δεν μπορεί κανείς να τους σε βοηθήσει. Δεν μπορεί να τους βοηθήσει να τα πράξουν όλα αυτά με βάση κανόνες. Και κάτι άλλο. Ίσως ε, θα έπρεπε να προσφέρουμε κάποια βοήθεια στην κυβέρνηση της Κροατίας γιατί ε, και όπως και σε άλλες περιπτώσεις, ε, το όλο θέμα αυτή τη στιγμή δεν εξαρτάται από κομματική πολιτική. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη για τις ε, αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου, οφείλουμε με τη Frontex και με άλλους να βοηθήσουμε έτσι ώστε να απαλύνουμε την κατάσταση, να την αποκλιμακώσουμε, να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τους ανθρώπους, γιατί η κατεύθυνση δεν μπορεί να είναι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να είναι και επιστροφή στην πατρίδα, ανάλογα με το αν έχει το δικαίωμα να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Γιατί το δόγμα όλοι να μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν ε, ταυτίζεται ταυτίζει με τους νόμους μας και εμείς έχουμε κάποιους νόμους και οδηγίες και δεν μπορούμε τώρα αυθαίρετα να αποφασίζουμε ότι όποιος μόνος το αποφασίζει ότι δικαιούται άσυλο ή ότι είναι πρόσφυγας να μένει εδώ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι και οι ΜΚΟ πρέπει να τηρούν τους απαραίτητους ε, κανόνες. Εγώ είμαι κάθετα κατά της ποινικοποίηση, αλλά εκεί όπου οι ΜΚΟ πιστεύουν ότι πρέπει να προχωρήσουν πιο πολύ, νομίζω ότι εκεί πρέπει να αντιμετωπίζουν ε, το κράτος, όπου πραγματικά βοηθάνε, γιατί βοηθάνε τους ανθρώπους και εμείς στη Γερμανία έχουμε πάρα πολλούς που βοηθάνε. Αυτοί πρέπει να στηρίζονται οικονομικά έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τη βοήθειά τους στους ανθρώπους που βρίσκονται στη χώρα μας. Η βοήθεια να ε, δίδεται από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι η επιχειρηματολογία μας ε, θα πρέπει να είναι λιγάκι διαφοροποιημένη, γιατί οι συλλήβδιν κατηγορίες, όπως σας είπα, δεν βοηθούν, βοηθούν μόνο τους λαϊκιστές και αλλιώς κανέναν άλλο. Πρόεδρος, δεν έχουμε πια πολύ χρόνο, αλλά θα ήθελα να ζητήσω από τους τρεις συναδέλφους να τοποθετηθούν στα ερωτήματα που ετέθησαν, να μην κάνουν νέες ομιλίες. Και για την Επιτροπή θέλω να πω ότι αν έχετε την καλοσύνη να εστιάσετε σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Δηλαδή, ε, εγώ θεωρώ ότι είναι παράλογο γιατί υπάρχουν αρκετές αποχρώσεις ενδείξεις και αυτό που ενδιαφέρει είναι το τι γίνεται με τις ΜΚΟ. Ε, υπάρχουν παρεμβάσεις ε, στα σύνορα, στη Μεσόγειο, αλλά νομίζω ότι αυτές οι περιπτώσεις έχουν ασκήσει πολύ μεγάλη επιρροή είναι απόλυτα δικαιολογημένο το αίτημα του Κοινοβουλίου. Βεβαίως δύσκολο και για εσά, γιατί έχετε να κάνετε με διαφορετικά κράτη-μέλη, αλλά η απάντηση που δώσατε στην αρχή ε, πραγματικά μας ε, ε, φοβίζει λιγάκι. Ως εκ τούτου, ίσως μπορείτε να προσπαθήσετε να μας εξηγήσετε περί τίνος ακριβώς πρόκειται πριν ολοκληρωθεί η θητεία να μας πείτε τι είναι εκείνο που σας εμποδίζει να κάνετε κάτι άλλο. Κατά τα άλλα αυτό έχει ε, προετοιμαστεί από την Επιτροπή Αναφορών και όχι από τη δική μας Επιτροπή. Και αυτά που λένε οι ΜΚΟ ε, δεν είναι ότι προάγουν την παράνομη μετανάστευση, απλά θέλουν ε, μια ξεκάθαρη θέση για να μην ποινικοποιούνται. Πριν ολοκληρωθεί η θητεία, Θέλω να σας πω, επαναλαμβάνουμε, δεν ενισχύουμε τη μετανάστευση, απλά επιθυμούμε μία ξεκάθαρη θέση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Νομίζω αυτά η Κομισιόν τα γνωρίζει. Να μην καταλήξουμε στο να ποινικοποιούνται οι ΜΚΟ. Δίκιο έχει η κυρία Χόλμα, το πράγμα είναι περίπλοκο στα κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές και εμείς αυτό ζητάμε από εσά να τοποθετηθείτε στις κατευθυντήριες γραμμές. Και όσον αφορά τη Frontex, όταν θα έρθει ο κύριος Αβραμόπουλος θα του δείξουμε το θέμα της επιστολής. Θα ήθελα παρακαλώ να απαντήσετε όσο πιο καθαρά γίνεται, ξεκινώντας μέσα ε, νομίζω ότι αυτό το οποίο προκύπτει είναι πάρα πολύ περίπλοκο όσον αφορά την ε, αλληλεπίδραση με το ποινικό δίκαιο. Αλλά δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλείνει τα μάτια της. Μου είπατε να μην κάνω ομιλία, αλλά και εγώ έχω να πω πολλά πράγματα, γιατί ελέγχθησαν πολλά βαριά ε, που δεν είναι και απόλυτα αλήθεια. Κοιτάξτε, η Κομισιόν δουλεύει πολύ σκληρά όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές. Εμείς δουλεύουμε σκληρά σε αυτό. Έχουμε κάνει αξιολόγηση, σοβαρή αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι εδώ μιλάμε για το ποινικό δίκαιο. Είναι κάτι το πάρα πολύ ευαίσθητο για όλα τα κράτη-μέλη. Εμείς ε, δεν παρεμβαίνουμε στο εθνικό ποινικό δίκαιο του κάθε κράτους μέλους, αλλά μην δημιουργείτε την εντύπωση ότι η Κομισιόν κλείνει την πόρτα. Όχι. Το εξετάζουμε το θέμα. Έχουμε διάλογο. Είναι σημαντικό για μας να διατηρηθεί ο διάλογος. Άκουσα τι είπαν οι συνάδελφοι και αυτό και άλλα στοιχεία θα τα λάβουμε υπόψη μας. Ε, θα τα εξετάσουμε ε, θα εξετάσουμε όλες τις μελέτες και όπως σας είπα αυτή είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Ε, προβλέπεται μία συνάντηση ε, και στη συνάντηση αυτή θα τα εξετάσουμε όλα με περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Κομισιόν δεσμεύεται και αξιολογεί ιδιαίτερα την θαμάσια δουλειά των ε, οργανώσεων ε, ε, της κοινωνίας των πολιτών. Θέλουμε να είμαστε ενημερωμένοι για τις συνθήκες, τα ακούσαμε αυτά σήμερα το πρωί και όπως είπα και προηγουμένως, σε περιπτώσεις που κρίνεται σκόπιμο, εμείς εκεί πραγματικά έχουμε παρέμβει, έχουμε δρομολογήσει διαδικασίες επί παραβάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και δρά αποφασιστικά. Γι' αυτό να ξεφύγετε λιγάκι από αυτή την άποψη που έχετε ότι η Κομισιόν δεν κάνει τη δουλειά της. Όχι, η Κομισιόν την κάνει τη δουλειά της και την κάνει με βάση αποδεικτικά στοιχεία. Μα τα έχετε, λέει ο Πρόεδρος, τα αποδεικτικά στοιχεία. Κοιτάξτε, λέει ο πρόεδρο, εμεί ε, δεν θέλουμε να φύγει η Επιτροπή που να έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ε, κατανοεί βέβαια την πίεση στα κράτη-μέλη, αλλά τώρα ε, η Κομισιόν ακολουθεί μια διαφορετική διαδρομή γιατί λέτε ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Μα συγγνώμη, η Επιτροπή Αναφορών έχει προετοιμάσει αυτή την υπόθεση και είναι και αρκετά εκτεταμένη το να λέει κανείς ε, ότι όλα αυτά ε, υπάγονται στο ποινικό δίκαιο, αυτό είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Γιατί υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές ε, οι οποίες για όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν έτσι ώστε να μην ποινικοποιούνται οι ΜΚΟ. Αυτή είναι μια κλασική περίπτωση για την Κομισιόν. Αν η απάντηση είναι ότι αυτό δεν αρέσει στα κράτη-μέλη, εντάξει τη δεχόμαστε, αλλά κατά τα άλλα δεν μπορεί κανεί να λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, ότι ότι είναι αυτά όλα θέμα ποινικού δικαίου, εντάσσονται στο ποινικό δίκαιο. Εγώ σας είπα, μέχρι το τέλος τη θητεία θέλουμε να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Ε, γιατί από ό,τι φαίνεται φοβάμαι δεν μπορούμε να βασιστούμε στο ότι η Επιτροπή ε, θα σημειώσει πρώτο. Ε, εσείς μου βάζετε ε, λόγια στο στόμα, ότι εγώ είπα ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Εγώ είπα ικανοποιητικά επαρκή, επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Απαρκή αποδεικτικά στοιχεία νομίζω ότι υπάρχουν. Η Frontex θέλετε να τοποθετηθείτε παρακαλώ στο θέμα της επιστολής. Δεν μπορώ να απαντήσω για το θέμα της επιστολής ε, που αναφέρθηκε. Αν αυτή είναι η ερώτηση που είχατε για μένα, δεν μπορώ να απαντήσω. Θα το θίξουμε με την Κομισιόν. Αν θέλετε όμως σε συντομία να απαντήσετε. Ναι, θα απαντήσω στις ερωτήσεις ε, που τέθηκαν ε, σε ό,τι αφορά την περίπτωση του κοριτσιού, ενώ ήταν υποκράτηση οικογένεια, τρεις φορές έπρεπε να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ε, διατάξει την Κροατία, να απελευθερώσει την οικογένεια από την κράτηση και να μπορεί να έρθει σε επαφή με τον δικηγόρο. Ε, ξεκινήσαμε την υπόθεση εκ μέρους της οικογένειας της Ματίνα, καθώς ε, ήταν άγνωστος δράστης, όμως απέριψε η δικαστική αρχή την υπόθεση λόγω της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων και κατόπιν αποφασίσαμε να στείλουμε την υπόθεση σε υψηλότερα δικαστικά όργανα και ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη τελικά θα απονεμηθεί. Σε ό,τι αφορά τη δική μας υπόθεση. Φοβόμαστε ότι μπορεί να περιμένουμε για χρόνια να αποφανθεί το ανατό δικαστήριο και ε, στο πρωτοδικείο συνεχώς απεξινόταν η δουλειά μας σε ό,τι αφορά το τι χρειαζόμαστε. Μπορεί να χρειαζόμαστε 43.000 ευρώ αλλά ελπίζουμε ότι τελικά δεν θα χρειαστεί, γιατί ελπίζουμε ότι υπάρχει το κράτος δικαίου στην Κροατία. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο τι χρειάζονται οι αιτούντες άσυλο στην πραγματικότητα, πραγματική δυνατότητα να ζητήσουν διεθνή προστασία χωρί να αποθούνται ή να ξυλοκοπούνται. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε τα επιχείρηματα του Υπουργείου τη Κροατία, όπου αναφέρεται το άρθρο 13 του Συνοριακού Κώδικα Σέγγεν για να δικαιολογήσει τι αποθήσει, ενώ γνωρίζει το άρθρο 14 που λέει ότι πρέπει να αποφεύγεται αυτή η πρακτική. Μέχρι να επιληθεί λοιπόν αυτό η ΜΚΟ θα πρέπει να συνεχίζουν να υποστηρίζουν τους πρόσφυγες ε, στο να ρυθμίσουν το νομικό τους καθεστώς χωρίς να φοβούνται την ποινικοποίηση. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν ε, ναι, θα πρέπει να λάβει μια πιο κάθετη θέση για το θέμα αυτό και να ορίσει καλύτερα τους κανόνες γιατί στη δική μας περίπτωση βλέπετε ότι η κροτική κυβέρνηση χρησιμοποιεί κάποιες άρρωστες συστάσεις κατά τον ΜΚΟ. Εμείς απλώς ε, ζητούμε για το σεβασμό του νόμου και από τις δύο πλευρές. Ωραία, ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές και ευχαριστώ για τους συναδέλφους που ήταν παρόντες και συμμετείχαν στη συζήτηση. Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 9. Αν θέλουν οι συνάδελφοι να συμμετέχουν να έρθουν εδώ, έχουμε καθυστερήσει λίγο. Θα παρουσιάσω λοιπόν το σημείο όσο έρχονται οι συνάδελφοι. Πρόκειται για την, ε, τον έλεγχο καταλληλότητας ε, που ξεκίνησε η Κομισιόν στο τέλος του 2016 αφού ανακοίνωσε τον Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση στο μέτρο του 2015 υποτίθεται ότι έπρεπε να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2018 Είχαμε αρκετά στοιχεία όπως ε, το νομοθεσία για την μπλε κάρτα για άλλα ζητήματα, αλλά είχαμε και κάποιες μελέτες σε σχέση με το κόστο της μης Ευρώπης ε, στο θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Έτσι λοιπόν είναι ένα πολύ δύσκολο τομέα αυτός, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ιδιαίτερη κινητικότητα για την νομιμή μετανάστευση και στο Κοινοβούλιο που δεν μπορούμε καν να καταλήξουμε σε πρώτη ανάγνωση για την μπλε κάρτα, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να προδεύσει επειδή έχει τον όρο μετανάστευση εντός. Είμαστε λοιπόν σε πολύ κακή κατάσταση, σε δύσκολη θέση. Δεν έφταει η Κομισιόν εδώ. Ε, η Κομισιόν τα πάμε δυστυχώς κάποιες από τις ομάδες μας εδώ στο Κοινοβούλιο ε, μπλοκάρουν. Έτσι λοιπόν είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση για την αναθεώρηση της μπλε κάρτας η πρώτη ανάγνωση. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το κάνουμε αυτό. Πρόκειται για έλεγχο καταλληλότητα, ε, για την ομετράστευση. Κανένα δεν είναι κατάλληλο και αν θέλετε μπορούμε να το κλείσουμε εδώ. Αν έχετε καλύτερα πράγματα να κάνετε, δεν ξέρω. Μπορούμε απλώ να ζητήσουμε από τι ομάδε ε, που δεν θέλουν ε, την πλεκάρτα στην πρώτη ανάγνωση να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ή θέλετε να πείτε κάτι. Θα υπάρχει τελικά καθόλου νόμο μετανάστευση στην επόμενη θητεία. Δεν είμαι σίγουρη. Τώρα δεν φταίει η Κομισιόν, δεν θα σα ασκήσουμε κριτική γι' αυτό βλέπω ποιο φταίει, αλλά ίσως μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα λίγο περαιτέρω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ουσιαστικά αντιμετωπίζει με έναν ελεύθερο τρόπο την νόμιμη μετανάστευση. Καταρχήν, ε, λοιπόν, ε, να ακούσουμε εσάς κυριετηριών και κατόπιν θα ακούσουμε την παρουσίαση των που συζητούσαν οι συνάδελφοι για το κόστος της μη νόμιμης μετανάστευσης. Πού βρισκόμαστε λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την μπλε κάρτα ίσως, να μας πείτε τις σκέψη σας. Uh, um, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ε, θέλω να σας πω σε σχέση με την εισαγωγή σας ότι και σήμερα έχουμε νόμιμη μετανάστευση ε, ε από την ανθρωπιστική σκοπιά ε, που είναι η μετεγκατάσταση και εφαρμόζεται. Έχουμε και πιλωτικά προγράμματα που πριν από λίγες εβδομάδες αναφέρθηκαν και έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και έχουμε και την γαλάζια κάρτα ε, που αναφέρατε και χαίρομαι πάρα πολύ που και σας είμαι ευγνώμων που είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επίτροπη ε, δεν ευθύνεται για την αποτυχία αυτού του εγχειρήματος. Μάλλον το Συμβούλιο που το βλέπει κάπως επιπόλαια και ελαφρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει η γαλάζια κάρτα που λειτουργεί. Και όχι το Κοινοβούλιο, λέει ο Πρόεδρος τη Επιτροπής. Ναι, ναι, το ξέρουμε, δεν φταίει και το Κοινοβούλιο. Είναι σαφή τα πράγματα αυτά. Αλλά σε σχέση με αυτό το πλαίσιο, ποιο είναι το θέμα θελήσαμε να ελέγξουμε κατά πόσο η πολιτική που έχουμε για την νόμιμη μετανάστευση και το κεκτημένο, το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, είναι κατάλληλο για το σκοπό που έχει δημιουργηθεί. Και θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ταυτόχρονα είναι αναγκαιότητα και πραγματικότητα η μετανάστευση, αλλά και περίπλοκο φαινόμενο πολύ. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο ε, ζήτησαν να γίνουν οι μελέτες αυτές και τώρα έχουμε αρκετά στοιχεία και βάσει αυτών μπορούμε να κάνουμε τους σχεδιασμούς μας, τους προγραμματισμούς μας και να οικοδομήσουμε τη μελλοντική μας πολιτική. Εντάσσω και τις δύο μελέτες στο ευρύτερο πολιτικό και γενικότερο πλαίσιο ε, λόγω της λεγόμενης μεταναστευτικής κρίσης και της κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα, η πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια εστιάστηκε πάρα πολύ στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και στη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων και την αποτελεσματική διαχείριση ε, της έλευσης και αύξηση των ανθρώπων που ζητούν προστασία ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπήρξε μια ευρύτατη πολιτική συνένεση ανά την Ευρώπη ότι θα πρέπει να μειώσουμε όσο ε, αυτό είναι δυνατό την παράνομη μετανάστευση, αλλά δεν μπορούμε να σταματούμε εκεί. Ε, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν φτάνει αυτό θα πρέπει να διαχειριστούμε γενικότερα τη μετανάστευση πολύ πέρα από την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και ε, τα θέματα της αντιμετώπισης των επιγουσών καταστάσεων. Είναι τρεις πυλώνες. Ανθρωπιστική ε, ανθρωπιστικοί λόγοι που είναι η μετακατάσταση. Ε, επίσης, νόμιμη μετανάστευση χρειαζόμαστε για τις αγορές εργασίας μας. Αλλά και ο τρίτος πυλώνας είναι να υπάρχουν νόμιμες οδοί ε, προς την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες, έτσι ώστε να προσφέρουμε μία οδό στους μετανάστες. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη προώθησε την νόμιμη μετανάστευση ε, στο ε, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα το αντίστοιχο και το θεματολόγιο το 2015 στην αντίστοιχη ανακοίνωση και του περασμένου Σεπτεμβρίου και στην τελευταία έκθεση προόδου, την πολύ πρόσφατη του Μαρτίου 2019. Ποια είναι λοιπόν τα αποτέλεσματα του ελέγχου καταλληλότητας που κάναμε. Είναι σημαντικό να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική νόμιμης μετανάστευσης, γενικότερα ε, στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Υπάρχουν και θετικά στοιχεία βάσει ε, του σημερινού κεκτημένου και θα ήθελα να σας δώσω δύο παραδείγματα Πρώτον, αυξάνεται το επίπεδο των δικαιωμάτων και η προστασία της οικογενειακής ζωής για τους ε, νομίμως διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλού υπήρξαν πιο περιορισμένες επιδράσεις, ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά την προσέλκυση των ταλέντων και των δεξιοτήτων που χρειαζόμαστε για την αγορά εργασίας. Αναφερθήκατε και εσείς αυτό, Πρόεδρε. Και μετά υπάρχουν και κάποια οριζόντια κρίσιμα θέματα, το νομικό πλαίσιο που είναι κατακαιρματισμένο και έχει και πολλά ελλείμματα. Υπάρχουν και προβλήματα εφαρμογής σε ό,τι αφορά τη μεταφορά της οδηγίας για την νόμιμη μετανάστευση. Η συνέχεια βεβαίως ε, αφορά την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το επόμενο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Αλλά τώρα το θέμα είναι οι ουσιαστικές ε, συζητήσεις για να εξαχθούν τα σωστά πολιτικά συμπεράσματα. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Πρώτον, θέλουμε πιο εναρμονισμένη και αποτελεσματική προσέγγιση για να προσελκύονται εργαζόμενοι υψηλών προσόντων. Ε, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και τα κοινά και να υπάρχει ε, τρόπος υποβολής ε, ενδιαφέροντος. Οι συνάδελφοι που θα ακολουθήσουν θα μπουν σε λεπτομέρειες για τα μοντέλα αυτά, τα οποία ε, ήταν αρκετά επιτυχή στον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Στην Ευρώπη έχουμε ε, μοντέλα ε, που βασίζονται στη ζήτηση. Δηλαδή για να έρθει κάποιος νόμιμα μετανάστης ε, πρέπει να έχει συγκεκριμένη προσφορά η θέση εργασίας. Ενώ οι άλλες χώρες έχουν μια προεπιλογή και στη συνέχεια βρίσκουν τους ειδικού από την προεπιλογή αυτή. Ε, τα συστήματα λοιπόν των τρίτων χωρών δεν είναι ένα προς ένα εύκολο να μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιγραφούν. Αλλά Στη Σουηδία και την Πολωνία υπάρχουν ήδη καλές εμπειρίες. Ε, αυτά τα στοιχεία της μελέτης ε, θα μας οδηγήσουν και σε συμπεράσματα. Τελειώνω εγώ λέγοντας το εξής. Όλα τα θεσμικά όργανα και οι ενεχόμενοι που συμμετείχαν στη διαβούλευση για τον έλεγχο καταλληλότητας συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών ετώνησαν ότι ένα κοινό ε, νομικό πλαίσιο έχει ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία. Αυτό είναι με ένα ελπιδοφόρο, αλλά θα δούμε στις λεπτομέρειες τι σημαίνει και υπάρχει και ανάγκη ε, να έχουμε μια πιο μακροχρόνια, μια πρόθεσμη προοπτική για τη μετανάστευση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα παραμελήσουμε τις σημερινές ανάγκες. Δεύτερον, στο μέλλον χρειάζεται να επεκταθεί και να διευρυνθεί το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Αυτό είναι ζήτημα των επομένων μηνών τα ευρήματα της μελέτης μας ε, είναι χρήσιμα. Ε, χρειάζεται δουλειά από όλους, το Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε η κοινή μας πολιτική για την νόμιμη μετανάστευση είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα και τις προκλήσεις των οικονομιών και των κοινωνιών μας. Περιμένουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον τις απόψεις σας και την επόμενη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ε, τελευταίο σχόλιο, Πρόεδρε. Τώρα μπορεί κανείς να δει το ποτήρι μισό γεμάτο ή μισό άδειο. Είναι θέμα ερμηνείας. Πάντως κάτι έχει μέσα το ποτήρι. Και τα επόμενα χρόνια, τις επόμενους μήνες, την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο θα πρέπει να φροντίσουμε να το γεμίσουμε το ποτήρι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει καν ποτήρι. Κανείς δεν βάζει τίποτα σε αυτό το ποτήρι. Δεν υπάρχει ποτήρι. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε νόμιμη μετανάστευση. Το θέμα μας είναι η επαναπρόθεση. Ε, μερικοί λένε δεν υπάρχει καν νόμιμη μετανάστευση. Εν πάση εσείς ε, πρέπει να κάνετε τη δουλειά σας. Ε, εμείς πιστεύαμε ότι τα κράτη-μέλη που συνεχίζουν και λένε ότι πρέπει να υπάρχει κάποια νόμιμη οδός έτσι ώστε να μην υπάρχει τόσο εκτεταμένη τόσο εκτεταμένη παράνομη μετανάστευση. Τα κράτη-μέλη και οι λαϊκιστικές δυνάμεις, τα κοινοβούλια, θέλουν να θεωρήσουν το έγγραφο περί δεξιοτήτων αυτό που λέμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ίσως να αναθεωρήσει τι απόψει. να είναι λίγο πιο ρεαλιστική. Δεν μπορούμε να έχουμε νόμιμέ οδούς, ε, γιατί δεν μπορούμε και καν να αναθεωρήσουμε το θέμα, το φάκελο με, τα, ε, με τις υψηλές και ουσιαστικές δεξιότητες. Φαρισαϊσμός υπάρχει. Δεν μπορούμε να βρούμε νόμιμες οδούς για να αποτρέψουμε την παράνομη μετανάστευση. Εγώ δεν είμαι και ιδιαίτερα αισιόδοξο, αλλά και πάλι βέβαια αυτό ε, δεν είναι το πρόβλημα της Κομισιόν ε, σχετικά με τη μετεγκατάσταση. Η μετεγκατάσταση δεν εντάσσεται στο θέμα της ε, νόμιμης μετανάστευσης. Τώρα, να δούμε το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης Ο Πίτε Βαν Μπαλεχόη και οι συνάδελφός του ε, θα ε, μας παρουσιάσουν το επόμενο θέμα. Θα παρουσιάσουν μία μελέτη και νομίζω η Ελίνα θα ε, παρουσιάσει το θέμα αυτό. Thank you very much and can we move to the second Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσει κανείς ε, την παρέμβασή του. Εν πάση θα κάνω ό,τι μπορώ. Ε, θα παρουσιάσω το Μη Ευρώπη ε, κάτω από το πρίσμα της μετανάστευσης σήμερα και βλέπουμε ότι έχουμε εδώ και ένα από τους συντάκτες αυτής της ε, μελέτης. Πριν περάσουμε στο θέμα της ε, νόμιμης μετανάστευσης, ε, θέλω να πω ότι αυτό εντάσσεται σε ένα αίτημα που στείλατε σε εμά και στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ήθελα λοιπόν να δράξω την ευκαιρία για να διευκρινίσω το γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Και νομίζω ότι αυτό αναφέρθηκε ήδη σε μια έκθεση του 1983 που συντάχθηκε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκεί αναφέρεται η μη Ευρώπη. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα τα φαινόμενα επιτείνονται και ίσως τότε αυτό να ήταν έτσι μια προφητική δήλωση. Το κλειδί για για την έκθεση αυτή, ε, όπως θα αναφερθεί και στην επόμενη ενημέρωση, είναι να δούμε λιγάκι τα θέματα της ελευθερίας, της δικαιοσύνης. Αυτό που λείπει είναι ότι δεν υπάρχει εφαρμογή, δεν εφαρμόζονται οι διεθνείς κανόνες και οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και επίσης ε, δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται σεβαστό το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε σήμερα κάποια παραδείγματα. Αυτές οι ελλείψεις έχουν επιπτώσεις σε ατομικό επίπεδο δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ασκήσει και να διεκδικήσει κανείς τα ατομικά του δικαιώματα, αλλά υπάρχουν και οικονομικές επιπτώσεις. 180 δις ευρώ είναι το αποτέλεσμα, είναι ο λογαριασμός. Ας δούμε τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε οι κοινωνίες να είναι πιο ασφαλείς και πιο ελεύθερες. Υπάρχουν αρκετές επιλογές ε, που θα μπορούσε να επιλέξει ο νομοθέτης που περιλαμβάνουν περαιτέρω ε, προσπάθειες ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημιουργία των νόμιμων οδών για τους μετανάστες να μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ολοκλήρωση του πλαισίου των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που προκύπτει λοιπόν από όλο αυτό το πρόγραμμα είναι ότι όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα υπάρχουν τρεις σημαντικές διαστάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, όταν μιλάμε για μετανάστε, πρέπει να δει κανείς τι μεταναστευτικέ και βλέπουμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις ε, σωρεύονται σε αυτές τις ε, μεταναστευτικές οδούς. Αυτή είναι μια εικόνα που έχει σχέση με την πολιτική ασύλου που σας παρουσίασα στις αρχές του έτους. Και εκεί φαίνεται ε, τις αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες σωρεύονται για το μεμονωμένο ενδιαφερόμενο. Ένα άλλο ενδιαφέρον πόρισμα από αυτή την έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις στα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ότι έχουμε άμεσες και έμεσες επιπτώσεις οι οποίες επίσης ε, ε, επιδεινώνονται στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Δηλαδή, ε, δεν ε, ψάχνουμε αμέσω το υλικό και το άϊλο κόστο, αλλά βλέπουμε και το τι προκύπτει για το συγκεκριμένο άνθρωπο σε επίπεδο παιδεία, απασχόληση, αλλά και τη ε, σωματική και τη πνευματική του υγεία, λόγω του ότι ακριβώ δεν υπάρχει συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ βλέπουμε έναν πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται όλες οι αρνητικές επιπτώσεις, ε, ε, κυρίως όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι έχουμε αυτή τη γραμμή που βλέπετε με τις κουκίδες γύρω από το πλαίσιο ε, και εκεί φαίνεται η έλλειψη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι η διαφθορά έχει κόστος, αλλά σίγουρα αυτή δεν είναι και η σφαιρική εικόνα. Πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες για να διαπιστώσουμε το τι χάνουμε που δεν έχουμε εγγυήσεις για τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ότι ορισμένοι τομείς επηρεάζουν με μονομένες ομάδες ε, που είναι μικρότερες από άλλες όπως η ΛΟΑΤΚΕ και άλλες ε, περιπτώσεις όπου διαπιστώνουμε ότι πρέπει να πράξουν περισσότερες ε, έρευνες. Η αυτοπροστασία ε, η αυτοδιάθεση είναι ένας τομέας όπου πρέπει να τον εξετάσουμε και βλέπουμε επίσης και το πορτοκαλί τετραγωνίδιο στο επάνω κομμάτι 22 δις ευρώ και επ' αυτού θα εστιάσω την προσοχή μου σύντομα. Τα βασικά πορίσματα αυτής της έκθεσης, την οποία θα επεξεργαστεί η συνάδελφός μου μετά από μένα, είναι ότι η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από 20 χρόνια ήταν να αντιμετωπίζονται ε, σωστά οι μετανάστες ε, χωρίς διακριτική μεταχείριση. Αυτό δεν εφαρμόζεται ε, δεν ισχύει. Υπάρχει λοιπόν και μια τομεακή προσέγγιση. Αυτά οι ελλείψεις και οι φραγμοί έχουν προκαλέσει απώλεια εισοδήματος και έχουν προκαλέσει επίσης και απώλεια εισόδων σε επίπεδο κοινότητας αλλά και η ε, ικανότητα των ανθρώπων αυτών να βρουν εργασία. Αυτό επίσης είναι ένα πρόβλημα. Αυτή η μελέτη καλύπτει μόνο, μόνο τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται εδώ και διαπιστώνουμε τις αρνητικές επιπτώσεις σε αυτούς. Όσον αφορά λοιπόν το μέλλον, ο συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ε, διάφορες δυνατότητες. Καταρχήν να υπάρχει καλύτερη εφαρμογή των κανόνων που υπάρχουν ε, και το τι πρέπει να λάβει υπόψη του το επόμενο κοινοβούλιο είναι να επεκταθεί η νομοθεσία και σε άλλους τομείς ή να υπάρχει και ένας δεσμευτικός ε, κώδικας ε, ε, που να καλύπτει όλες τις χώρες. Ανάλογα λοιπόν με την επιλογή που θα γίνει, 22 δις ευρώ, σας είπα, θα μπορούσαν να επιτυγχάνονται κάθε χρόνο. Αυτό θα είναι το όφελος και από αυτού μπορεί να συνεχίσει η Αλίνα. Παρακαλώ, η συνάδελφός μου. Thank you so much. Ευχαριστώ. Καταρχήν, ευχαριστώ και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που ζήτησε αυτή τη μελέτη και την ε, μονάδα του ΕΠΙΡΕΣ. Ήταν ε, μια συνεργατική προσπάθεια η μελέτη αυτή. Είχαμε διεπιστημονική έρευνα, εκεί συμμετέχαν, συμμετείχαν επιστήμονες, οικονομολόγοι, ε, πολιτικοί επιστήμονες το κόστος της ε, μη Ευρώπης ε, και η προσέγγιση μας καταρχήν ήθελε να εντοπίσει ε, νομικά κενά και πρακτικά εμπόδια στην σημερινό κεκτημένο για την μετανάστευση. Κατόπιν προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο στάτου, τον οικονομικό αντίκτυπο, τον αντίκτυπο σε επίπεδο ατόμων, σε ό,τι φορά την υγεία η μη Ευρώπη, η ανυπαρξία της Ευρώπης και θεωρώ ότι σε πάρα πολλούς τομείς και στον τομέα της μετανάστευσης ε, έχει ε, χαθεί το όνειρο είτε θα έχουμε μια πραγματική Ευρώπη ή δεν θα υπάρχει λύση. Ε, φοβάμαι ότι τα κράτη-μέλη δεν μετακινούνται. Αυτό λοιπόν πρέπει να ζητήσουμε γιατί αλλιώς θα χαθούμε σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς τομείς η Μπάρμπαρα. Θέλετε, Μπάρμπαρα, εσείς να πείτε κάτι παρακαλώ. Ε, ε, Κοιτάξτε, Εγώ είμαι σκιώδη συγγήτρια για την ε, μπλε κάρτα και θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδεικνύει ιδιαίτερο, ε, ιδιαίτερη αισιοδοξία όταν μιλά για το Συμβούλιο το οποίο θα έπρεπε να έχει κατανοήσει την ε, προστιθέμενη αξία που θα πρόκειται από την εναρμόνιση αυτών των νόμιμων οδών. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το Συμβούλιο, ξέρετε, τελικά δεν έχει καταλάβει τίποτα για όλα αυτά και το Συμβούλιο απλά ήθελε να ε, επιβάλλει την ε, αναπομπή της μπλε κάρτας, της blue card. Αυτή τη στιγμή όσον αφορά την μπλε κάρτα, έχουμε μία ε, κατάσταση. Ε, Μια κατάσταση που έχει προκύψει, που δεν λειτουργεί και νομίζω αυτά επιβεβαιώνονται πλήρως από το έγγραφο και την ε, μελέτη που παρουσιάστηκε προηγουμένως. Εάν λειτουργούσε, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είχε καταθέσει πρόταση αλλαγής. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα πρέπει ε, να κοιτάμε, να δούμε το ποτήρι αν θα είναι μισοάδιο ή μισογεμάτο, εγώ πιστεύω κάθε φορά που ένας πολιτικός χρησιμοποιεί αυτό το ποτήρι, το η πρόταση, εμένα με ζώνουν τα φίδια. Γιατί ε, αισθάνεται, ε, ή εγώ αισθάνομαι ότι ίσως υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί και να μην κατάλαβα ή να μην έχω συνειδητοποιήσει. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για απαντήσεις. Ε, σας είπα ότι δεν υπάρχει καν το ποτήρι, δεν υφίσταται το θέμα για τα μέτρα για την νόμιμη μετανάστευση. Θα ήθελα να δεχτώ και να πω με κάθε ειλικρίνεια ότι η όλη προσπάθεια είναι εμβαλωματική υπάρχει υψηλή ανεργία, υποτίθεται υπάρχουν ε, μέτρα προστασίας, ε, κατόπιν ε, υπάρχουν υποτίθεται οι δεξιότητες οι οποίες θα πρέπει να προβληθούν σε σχέση με τους μετανάστες. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν κάνει μελέτες. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και με ήπιες αναθεωρήσεις το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λειτουργούν λάθος. Συμφωνώ με την κυρία Σπινέλη ότι δεν μπορεί κανείς να είναι αισιόδοξο. Δεν είναι βέβαια απόλυτα η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όπως είπε η κυρία Σίπολ, οι άνθρωποι ε, δεν συνειδητοποιούν ότι το να μην υπάρχει Ευρώπη, η ανυπαρξία Ευρώπης, αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος. Εν πάση περιπτώσει, ε, δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ε, και είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε ε, τι θα γίνει με το επόμενο κοινοβούλιο, πώς, ποια θα είναι η σύστασή του, αλλά κάποιοι τουλάχιστον θα υπάρχουν και οι συνάδελφοί μας μας περιέγραψαν τι ακριβώς συμβαίνει. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την μελέτη που μας παρουσιάσατε και που μας δώσατε αυτό το fitness check. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους υπόλοιπους ε, συναδέλφους ε, από το, την Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεχίζουμε λοιπόν. Προχωρούμε στο θέμα της Eurojust και θα παρακαλούσα να έρθει στο πάνελ η Ερμόδη. Uh, λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε καθυστέρηση σχετική. Πάμε μέσα στο σημείο 10, που είναι η παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Eurojust από τον πρόεδρό της. Καλώς ορίσατε, Βλάτισλαβ. Πάντα χαιρόμαστε να υποδεχόμαστε τον πρόεδρο της Eurojust. Είχαμε πολλές συναντήσεις μαζί του και τουλάχιστον η Επιτροπή μας ξέρει πολύ καλά τι ε, δουλειά κάνετε, τι ανάγκες έχει ο οργανισμός, το προπολογισμό σας και τα λοιπά. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται για τη Eurojust και τις δραστηριότητές της, γιατί πραγματικά είναι αναγκαία και ξέρουμε ότι χρειάζεται προστασία ο ρόλος της και οι ανάγκες της ιδιαίτερες και αυτό φαίνεται σαφώς ε, κατά τα τέλη της ε, θητείας. Θα μας πείτε περισσότερα ότι είναι αιτήσια έκθεση που καλύπτει τα πεπραγμένα και τις δραστηριότητες ε, και μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνης. Θυμίζω στους συναδέλφους ότι το Δεκέμβριο είχαμε το νέο κανονισμό για τη Eurojust που θα τεθεί σε ισχύ, ελπίζουμε, για να δώσει περισσότερη επιχειρησιακή δυνατότητα στη Βλάντι στράφη σας δίνω το λόγο. Καλώς ορίσατε και παρακαλώ να μας παρουσιάσετε την ετήσια έκθεσή σας. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, Αγαπητά κύριε Μωράς, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε ε, την ετήσια έκθεσή μας για το 2018. Σε όλους σας. Για τελευταία φορά παρουσιάζω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ με τη συγκεκριμένη σύνθεση ε, αυτή την έκθεση. Και έχω κάθε λόγο να σας ευχαριστήσω, όπως είπε και ο Πρόεδρος, για την υποστήριξη που απολαύσαμε κατά τη διάρκεια της δικής σας θητείας. Δείξατε στην κοινοβουλευτική αυτή περίοδο ότι νοιάζεστε ε, ε, για την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους πολίτες, αλλά και για μας τους ίδιους τις αρχές ε, επιβολής του νόμου και τις δικαστικές. Εγώ σας ομιλώ ως εισαγγελέα. Οι εισαγγελείς διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αλυσίδα ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξασφαλίζουν ότι οι κακοποιοί ε, φυλακίζονται βάζει σε ισχυρά στοιχεία που έχουν ε, συγκεντρωθεί με νόμιμους τρόπους και πάντα με αρχές και ανθρώπινα δικαιώματα. Οι ε, εισαγγελίες είναι στην ίδια την καρδιά της αλυσίδας της ασφάλειας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είμαι ευγνώμων για όλη την υποστήριξή σας, την οποία επιδείξατε σαφέστατα και επιδείξατε ότι πραγματικά νοιάζεστε και για μας. Θέλω να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεσή μας. Στο πρώτο τμήμα θα μιλήσω λίγο για τρεις περιπτώσεις, τρεις υποθέσεις συγκεκριμένε, και αργότερα θα αναφερθώ σε κάποιες μελλοντικές προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει ο οργανισμός μου αλλά και το γενικό ποινικό σύστημα στην Ευρώπη θα ακούσετε, ενδεχομένως έχετε ακούσει την επιχείρηση Πολύνο που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα κοινή επιτυχία στην καταπολέμηση σοβαρού διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος. Η επιχείρηση αυτή, η υπόθεση συγκεκριμένη επιλέγει για την έκθεση γιατί δείχνει τι μπορούν να επιτυχάνουν οι χώρες όταν συνεργάζονται και όταν υποστηρίζονται από οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Europol και η Eurojust. Αυτή η υπόθεση ξεκίνησε το 2014 οι ε, Ολλανδικές αρχές ε, μας υπέστησαν την προσοχή ε, ότι εξέπλαιναν χρήμα μικρά εστιατόρια και καταστήματα που πουλούσαν παγωτά. Και σύντομα ανακάλυψαν ότι υπήρχαν διασυνδέσεις με τη Γερμανία και αποτάνθηκαν στους ομολόγους τους στη Γερμανία για να δουν τι γίνεται και εκεί. Και για να μην τα πολυλογώ, έγιναν πολλές εκεί συνεδριάσεις και οι δύο χώρες ανακάλυψαν ότι υπήρχαν και άλλες συνδέσεις με άλλες χώρες όπως η Ιταλία και το Βέλγιο. Και γι' αυτό επειδή ήταν πολλές ενεχόμενες χώρες ε, στη Eurojust ε, ασχοληθήκαμε αυτό το θέμα μαζί και με τη Europol. είχαμε συνεισφορές των κρατών μελών προς την Europol και χάρη σε αυτό προετοιμάσαμε και εκπονήσαμε μια αναλυτική έκθεση και καταλάβαμε καλύτερα την εικόνα της εγκληματική αυτής δραστηριότητας. Από τη Λατινική Αμερική λοιπόν εισήγαγαν ε, ναρκωτικά από την Αμβέρσα και το Ρότερνταμ από τους λιμένες αυτούς και στη συνέχεια τα πουλούσαν κυρίως στη Γερμανία ε, και τα ε, έσοδα κατέληγαν στις κάτω χώρες. με αυτή τη διασυνοριακή λειτουργία προσπαθούσαν να ε, ξεφύγουν από τις διοκτικές αρχές ε, και κάθε τμήμα της αλυσίδας φαινόταν σαν να ήταν ένα ξεχωριστό τμήμα και όχι ένας κρίκος μιας αλυσίδας και ενός δικτύου διασυνοριακού και διεθνούς. Γιατί νόμιζαν ότι οι διοκτικές αρχές κάθε χώρας θα δρούσαν ξεχωριστά. Ε, οι χώρες αυτές λοιπόν ε, σύστησαν μια ομάδα κοινή ερευνητική με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust ε, που ζήτησε και οικονομική υποστήριξη η ομάδα αυτή. Επί μια τριετία λοιπόν χρηματοδοτήθηκε και από ε, κοινοτικούς πόρους 180.000 ευρώ. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα που έδωσαν στους Ευρωπαίους φορολογουμένους, πολύ εντυπωσιακό. Δύο εκατομμύρια ε, προϊόντα ε, ε, εγκλήματος και τέσσερι, χρήματα και τέσσερις τόνοι κοκαΐνη ένα δις ευρώ αξία και 84 άτομα συνελήφθησαν. Αυτό πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακός δείκτης ε, απόδοσης και επίδοσης μάλλον. Και αυτή η υπόθεση μας λέει ότι ε, δεν θα πρέπει ποτέ να υποτιμούμε σχετικά μικρές διμερείς περιπτώσεις και υποθέσεις που μετά από πολλή δουλειά ε, φαίνεται ότι είναι και πολυμερείς με πολλές διακλαδώσεις και πλοκάμια και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Και ε, κάποιες υποθέσεις χρειάζονται χρόνια για να αναπτυχθούν, ενώ άλλες χρειάζονται ταχύτατη δράση. Ε, να σας παρουσιάσω ένα παράδειγμα ειδικής εκμετάλλευσης Τον Αύγουστο του 2018 κατηγορήθηκε μια Σουηδή ότι ε, συστηματικά κακοποιούσε σεξουαλικά τα ίδια της τα παιδιά. Και αφού ανακαλύφθηκαν ε, ε, κάποιες μαγνητοφωνήσεις στην Σουηδία, ζητήθηκε βοήθεια πρώτον για να εντοπίσουμε την υποπτή και μετά θα μπορούσαμε να ε, εκδώσουμε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης με τη μορφή και στις γλώσσες που χρειάζεται αυτό. Και αυτό ακριβώς ε, πράξαμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Διευκολύναμε την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος ε, σύλληψης και της ευρωπαϊκής έρευνας εντολής για να γίνονται κατοίκον έρευνες. Και χάρη στην καλή νομοθεσία που έχουμε, καταφέραμε να τη συλλάβουμε και χάρη στην ε, βοήθεια των κοινωνικών υπηρεσιών που πήγαν τα παιδιά σε ένα ασφαλές μέρος, αποκαταστήσαμε και πάλι τη δικαιοσύνη. Και δεν θα ήταν πλήρης η αναφορά μου σε διάφορες υποθέσεις αν δεν αναφερόμουν στον, στην ε, την τρομοκρατία που είναι τόσο σημαντικό θέμα ε, για τα κράτη-μέλη και την Ευρώπη και πόση μεγάλη σημασία δίδεται. Πέρυσι ε, αντιμετωπίσαμε περίπου 200 περιπτώσεις τρομοκρατίας ε, που σημαίνει αύξηση και πάλι σε σύγκριση με την προπερασμένη χρονιά. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι το 2018, αλλά είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της αποτελεσματικής ε, και ουσιαστικής απόκρισης της δικαιοσύνης σε κάποιες απειλές για τις, ασφι... Ε, τις ασφάλειες. Πριν από μια μισή εβδομάδα μόλις ε, δώσαμε την υποστήριξή μας στις Ουγγρικές και Βελγικές αρχές. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Ένας σύρος συνελήφθη στην Ουγγαρία, ο οποίος ήταν ύποπτος ενεργούς συμμετοχής ε, στο φόνο 22 προσώπων. Απευθύνθηκαν σε εμά και εμείς εξασφαλίσαμε τις πληροφορίες με το σωστό τρόπο προς τις αρμόδιες αρχές και με βάση αυτές τις πληροφορίες ε, καταφέραμε να συλλάβουμε τον ύποπτο αυτό και να ε, φυλακιστεί και να μπορέσει να αρχίσει η διαδικασία παράδοσης. Την ίδια μέρα είχαμε και άλλες επιθέσεις στο Μαλί, στην Πορκίνα Φάσο και στην ε, ακτή Ελεφαντοστού το 2015 και 2016 με 74 νεκρούς και πολλούς ακόμα τραυματίες. Γιατί αναφέρω αυτή την υπόθεση, για τον εξής λόγο, διότι στην τρομοκρατία βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή μετακίνηση από το διμερές επίπεδο και τη διμερή διάσταση όλο και περισσότερο έχουμε διεθνή. Όλο και περισσότερες χώρες συμμετέχουν ε, στις έρευνες και ε, όλο και πιο εξέχοντα ρόλο διαδραματίζουν τρίτες χώρες πλέον. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και πρόθυμοι για τη συνεργασία με χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθούμε να οικοδομήσουμε γερούς δεσμούς με κάποιες περιφέρειες, όπως προκειμένου είναι η Δυτική Αφρική. Ανταλλαγή λοιπόν πληροφοριών, ανταλλαγή υποδεικτικών στοιχείων, όλο και περισσότερο αποκτούν σημασία ε, σε τέτοιες υποθέσεις. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζουμε και την πρωτοβουλία 7 κρατών μελών για να συσταθεί ένα μητρό αντιμετώπιση της τρομοκρατίας δικαστικού τύπου στη Eurojust για να ανοιχνεύουμε σχέσεις που έχουν διάφορες υποθέσεις μεταξύ τους. Αυτό ε, σε σχέση με τις ε, διάφορες συγκεκριμένες υποθέσεις. Τι γίνεται τώρα με τις μελλοντικές προκλήσεις. Τρεις είναι αυτές. Η πρώτη, η ψηφιοποίηση και οι τεχνολογίες, η συνεργασία με τρίτες χώρες και ο αγώνας για να διατηρήσουμε το σημερινό επίπεδο υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει η Eurojust στα κράτη-μέλη. Η ψηφιοποίηση είναι όλο και περισσότερο πρόβλημα. Ε, γιατί σε αυτόν τον όλο και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο ε, πολλοί εισαγγελεί είναι ακόμα ε, αναγκασμένοι να δρουν κάπως απομονωμένοι. Τα εθνικά συστήματα δεν έχουν σχεδιαστεί για να συνεργάζονται και να μοιράζονται πληροφορίες και αποδεικτικά στοιχεία με ε, εταίρους στην Αλοδαπή. Για το λόγο αυτό η Eurojust προτείνει ένα νέο όραμα προς την κατεύθυνση αυτή και το Δεκέμβριο προτείναμε ε, ε, ένα νέο project που λέγεται ψηφιακή δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό, πολύ απλά, διότι αυτή τη στιγμή η Eurojust λαμβάνει πληροφορίες με διάφορους μορφότυπους από διάφορους διάβλους και σε διαφορετικές γλώσσες. Και υπάρχουν λοιπόν δεδομένα στα εθνικά συστήματα τα οποία χρειάζεται ε, να ε, εισάγονται με το χέρι. Τα δεδομένα χρειάζεται να μεταφράζονται στα κράτη-μέλη ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απαιτούνται πολλές ε, προσπάθειες εκατέρωθεν για να ανταποκρινόμαστε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Τα κράτη-μέλη καλωσόρισαν αυτή την πρωτοβουλία της Eurojust και πρέπει να σας πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που θα συνεχίσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάλυση αυτών των θεμάτων και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε κάτι το χειροπιαστό στο εγγύης μέλλον. Ανέφερα ότι είναι απαραίτητο να συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρες σε θέματα τρομοκρατίας όσον αφορά την τρομοκρατία, πλέον το έγκλημα ε, επεκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει διεθνή διάσταση, ως εκ τούτου ε, αντίστοιχη πρέπει να είναι και η αντίδραση. Όσον αφορά τα στατιστικά δεδομένα, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν όλες και περισσότερες επιπτώσεις σε σχέση με τρίτες χώρες. Πέρσι είχαμε 1.300 περίπου περιπτώσεις που αφορούσαν χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να διευκολυνθεί λοιπόν η συνεργασία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θέλησαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της ε, Λατινικής Αμερικής. Το τελευταίο πρόβλημα, τα χρήματα και οι πόροι. Ε, στο μέλλον θέλουμε να διατηρηθεί το επίπεδο υπηρεσιών το οποίο προσφέρουμε αυτή τη στιγμή. Πέρυσι 3.300 περιπτώσεις άνοιξαν στη Eurojust και αυτά είναι η προαιρετική παραπομπή από κράτη-μέλη προς την Eurojust. Αυτό αντιστοιχεί σε μια αύξηση της τάξης του 22% και άλλες 3.400 ε, περιπτώσεις είναι παλιές περιπτώσεις που εκκρεμούν ε, σε γενικές λοιπόν γραμμές. Ε, στηρίζουμε τα κράτη-μέλη σε περισσότερες από 6.500 περιπτώσεις. Και αυτό το κάνουμε με έναν αρκετά περιορισμένο ε, προϋπολογισμό 38,6 εκατομμύρια. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός μας και μπορώ να σας ε, παραπέμψω στην ε, τελευταία σας έκθεση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Εκεί αναφέρεται ότι θα πρέπει να εστιάσετε σε δραστηριότητες που φέρνουν προς θέμενη αξία χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες απόδοσης. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα για αυτό το θέμα. Τώρα, όσον αφορά την μελλοντική προοπτική και το θέμα το χρηματοδοτικό, βλέπετε στη διαφάνεια τα στοιχεία ε, και θέλω να σας πω ότι αντιμετωπίζουμε οικονομικά προβλήματα. Αυτό βέβαια ενοχλεί γιατί υπάρχουν άλλες ε, αρχές εφαρμογής του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παίρνουν περισσότερα χρήματα. 33% θα πάρει στον επόμενο προπλογισμό περισσότερα Europol. Και μπορώ να σας φέρω και, αναφέρω και άλλα παραδείγματα, αλλά μπορείτε και να τα βρείτε στην ε, σελίδα 37 της ετήσιας έκθεσης. Και ο λόγος που τα αναφέρω όλα αυτά είναι πάρα πολύ απλός. Εκείνο το οποίο θέλω να σας επισημάνω εδώ είναι ότι η βασική συνταγή για επιτυχία στο θέμα της δικαστικής συνεργασίας η βασική συνταγή είναι ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και αυτή η μαγική λέξη το μαζί πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην αστυνομία και παρα, παραμελώντας την ε, δικαστική εξουσία, αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, το θέμα είναι στα χέρια σας ε, και εγώ, ολοκληρώντας, θέλω να πω ότι η Eurojust οργανώνει ε, μια ειδική εκδήλωση για όλους ε, τους υποψήφιους ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μπορείτε να μας επισκεφτείτε όλοι, θα είναι ανοιχτέ οι θύρες. 2 Μαΐου λοιπόν μπορείτε να έρθετε σε εμά για να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες μας. Θα έχουμε ανοιχτέ τις πόρτες μας σε όλους τους υποψήφιους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αν δεν σας πειράζει, σε τρεις να δώσω το λόγο αλλά αν θέλετε να μιλήσετε περισσότεροι ε, θα πρέπει όλοι να μιλάνε ένα λεπτό από ό,τι βλέπω δεν είναι δυνατόν θα έρθει μετά ο Επίτροπος και εκεί θα υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις ε, γιατί ε, θα είναι και η τελευταία του επίσκεψη εμάς ένα λεπτό γίνεται λέτε όχι αλλά εν πάση ένα λεπτό να μιλήσετε παρακαλώ ή δυνατόν Σας ευχαριστώ Πρόεδρε σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Υποστηρίζω το ρόλο της Eurojust. Πιστεύω ότι η Eurojust κάνει τη διαφορά και ιδίω αν σκεφτούμε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε το διεθνές οργανωμένο έγκλημα το οποίο διαπερνά τις κοινωνίες μας και ε, ουσιαστικά ε, στοχεύει στο ε, να παραπλανήσει ακόμη και τις κυβερνήσεις μας. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα της τρομοκρατίας, ότι οι άνθρωποι αυτοί δρούν για τρομοκρατικούς σκοπούς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιος είναι ο ρόλος της Eurojust, τι μπορεί να κάνει η Eurojust για να προστατεύσει τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Σύντομα θα περάσουμε η οδηγία για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και έχετε μα κατά νου την περίπτωση του Χουιπίντο, ο οποίος ήταν πηγή για αυτά τα football leagues. Έχει τώρα ε, συλληφθεί στην Πορτογαλία μετά από την έκδοσή του. Ακριβώς αυτά ε, αυτό το σκάνδαλο για το ποδόσφαιρο είναι ε, παράδειγμα μια φιωσικής οργάνωσης που διαπερνά το ποδόσφαιρο σε όλη την Ευρώπη. Ο ρόλος της Eurojust θα είναι πάρα πολύ σημαντικός και ήθελα να αναφερθείτε σε αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις στην Πορτογαλία για το ρόλο της Eurojust. Εντάξει, το κατάλαβα, λέει ο πρόεδρος, να είστε σύντομοι. <laughs> Γιατί θα έρθει ο Επίτροπος και θα έχουμε ένα εκατομμύριο ερωτήσεις και δεν έχουμε χρόνο. Νάταλη. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την ε, παρουσίαση. Εγώ υποστηρίζω το ρόλο του οργανισμού είναι εντελώς ε, απαραίτητος ε, και φαίνεται από τα όσα μας είπε ο Πρόεδρος, η δράση είναι ολοένα και πιο διασυνοριακή και διεθνική και φυσικά υπάρχουν και οι διακλαδώσεις. Η Eurojust έχει προσθεμένη αξία σε ό,τι αφορά τη δικαστική συνεργασία. Τρεις ερωτήσεις έχω να σας ε, θέσω. Μιλήσαμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ήταν και πιο σημαντική στιγμή ε, της παρουσίασής σας στην Επιτροπή Καταπολέμησης Τρομοκρατίες. Εμείς παρουσιάσαμε κάποιες συστάσεις που επιμένουν στο ρόλο του οργανισμού και υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Europol με μια ιδέα επιτακτικής συνεργασίας για να υποστηριχτούν οι δράσεις για την αποτελεσματική ανείχνευση των δραστών και των μελλοντικών τρομοκρατικών επιθέσεων. Αυτό το μνημόνιο που υπογράφει μεταξύ Eurojust και Europol και το χαιρετίζω ε, υπάρχει αυτό το μνημόνιο. Θέλω να μου πείτε ποιε είναι οι τα συγκεκριμένα στάδια για να ενισχυθεί συνεργασία. Πώς έχει εξελιχθεί η ανταλλαγή πληροφοριών. Μιλήσατε για την πρόκληση της ψηφιοποίηση και ε, ότι πολλές φορές ε, δρούν μεμονωμένα οι αρχές στα κράτη-μέλη. θα υπάρχει συστηματική ανταλλαγή. Και προτελευταία ερώτηση, σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Ε, η συνεργασία αυτή πώς ε, οργανώνεται συγκεκριμένα με την εισαγγελία και για την μεταρρύθμιση της Eurojust. Ήμουν εισηγήτρια και το περασμένο Οκτώβριο θετήσαμε τη σχετική νομοθεσία. Πού βρισκόμαστε με την εφαρμογή. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσινίτσι και κατόπιν κυρία Βερζιά και τέλος. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Χαμράν ε, για την παρουσίασή του. Εγώ ως ε, Ιταλίδα δικαστής ε, πάντοτε πίστευα στην ανταλλαγή πληροφοριών και στη δικαστική συνεργασία και στο δίκτυο συνεργασίας που είναι απολύτως απαραίτητο για την καταπολάμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Πάντοτε λοιπόν το υποστήριζε και η Eurojust ε, είχε σημαντική δουλειά. Πάρα πολλές ερωτήσεις θα είχα, θα προσπαθώ όμως ε, να πω δύο πράγματα. Καταρχήν, εσείς αναφερθήκατε στην υπόθεση Πολύνο και υπογραμμίσατε την ύπαρξη οργανωμένου εγκλήματος ενός ε, μαφιόζικου δικτύου, είπατε. Εσείς θεωρείτε ότι στη σημερινή νομοθεσία είναι κατάλληλα τα μέσα που έχουμε για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα, ε, για να λάβουμε υπόψη και τη διαφοροποίηση της νομοθεσίας μεταξύ των κρατών μελών, πώς θα έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος προς αυτή την κατεύθυνση και να έχουμε, πρέπει να χάρη, ένα κοινό ορισμό για την ε, εγκληματική οργάνωση. Και θέλω κάτι να ρωτήσει. Από τον προηγούμενο Οκτώβριο ανανεώθηκε η Σύμβαση του Παλέρμο και ε, εκεί έχουν προσχωρήσει 189 κράτη. Υπό το φως της αναγκαιότητας να ενισχυθεί η συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών, η Σύμβαση του Παλέρμο όπου έχει προσχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο μέσο και πώς θα μπορούσαμε να την αξιοποιήσουμε. Και τέλος μια συγκεκριμένη ερώτηση και κλείνω. Υπάρχει ένα θέμα επί του οποίου δεν έχουν γίνει πολλά ακόμη, αλλά κάτι θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε παρόλη την ε, πτωτική τάση του μεταναστευτικού και αναφέρουμε στη διακίνηση μεταναστών, στο πώς θα καταπολεμήσουμε τη διακίνηση των μεταναστών. Νομίζω ότι πολλά περισσότερα πρέπει να κάνουμε. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας και σας ευχαριστώ εκ νέου για την παρουσία σας εδώ και για την εξαιρετική δουλειά που κάνει η Eurojust στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Σας ευχαριστώ. Μαρή Κριστίν, παρακαλώ. Σύντομα γιατί περιμένει Επίτροπος. Σας παρακαλώ, Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Η Eurojust ε, προβαίνει σε διεθνή δικαστική συνεργασία. Εδώ είμαστε λίγο δύσπιστοι όταν ε, μιλάμε για διεθνή δικαστική συνεργασία δυνάμει ε, των χωρών με τις οποίες αυτή η συνεργασία υλοποιείται. Και γι' αυτό εξεπλάγει να διαβάσω τη σελίδα 30 της εκθεσής σας ότι η Eurojust ε, έχει συνεργαστεί με τη Λιβύη, τη μόνη χώρα που αναφέρεται στην έκθεση, στην Μεσόγειο, στην περιοχή της Μεσογείου. Όλοι ξέρουμε εδώ ότι δεν υπάρχει δικαστικό σύστημα στη Λιβύη. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε σε τι συνίσταται η συνεργασία μεταξύ Eurojust και Λιβύης και ιδίως σε τι συνίσταται υποθέσεις ε, επί των οποίων συνεργάζεται η Eurojust με τη Λιβύη σε ό,τι αφορά τη διακίνηση μεταναστών. Υπάρχει κάτι που μας εκπλήσει λοιπόν όταν ε, βλέπουμε τη λιβική πραγματικότητα και στην περίπτωση που δεν μπορεί να μας δώσει απαντήσεις ε, ο προσκεκλημένος μας θα έλεγα να θέσουμε την ερώτηση αυτή γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και αν μπορείτε σήμερα όλα, αν δεν μπορείτε σήμερα να μα τα απαντήσετε όλα, παρακαλώ να έλθετε σε επαφή με τα μέλη, όπω είπε η Μαρία Κριστίνε. Να είστε σύντομο, παρακαλώ. Πολύ ωραία, θα κάνω ό,τι μπορώ. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλες αυτές τις ερωτήσεις που ετέθησαν, για το ενδιαφέρον που επιδείξατε. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, την προστασία των καταγγελόντων ε, και την περίπτωση Ρουί Πίντο. Κοιτάξτε, η Eurojust ε, στηρίζει τα κράτη-μέλη ε, και η προστασία των καταγγελόντων είναι ένα θέμα πολιτικό, είναι ένα θέμα περισσότερο που αφορά στα εθνικά κοινοβούλια. Εκεί να καλούνται να δημιουργήσουν όλες τις προϋποθέσεις για να προστατεύονται οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Σε αυτή την περίπτωση, θέλω να σας πω, του Ρουιπίντο ήταν ε, καταγγέλνουν σε μια άλλη περίπτωση, αλλά παραδόθηκε από την Ουγγαρία στην Πορτογαλία για μια άλλη περίπτωση, όχι για εκείνη ε, για την οποία συνεργαζόταν με τις αρχές της αστυνομίας και τις δικαστικές αρχές. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, ε, στο ρόλο της Europol και στο μέλλον της ε, συνεργασίας ανάμεσα στη Eurojust, τη Europol, την ανταλλαγή πληροφοριών. Ξέρετε, εδώ επιθυμούμε και στόχος μας είναι να έχουμε μια συστηματική ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών ανάμεσα σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό είναι ήδη και νομικό αίτημα, είναι απέτηση που εκφράζεται μέσα από διάφορα εργαλεία ε, υπάρχει τράπεζα δεδομένων. Ε, γι' αυτό λοιπόν η πρόσβαση αυτή, hit no access, ε, είναι εφικτή και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αρκετά χρήματα για να ε, ικανοποιήσουμε αυτό το νομικό αίτημα. Γιατί το πρόβλημα είναι βασικά καθαρά οικονομικό. Όσον αφορά την περίπτωση Πολίνο, Πράγματι είναι απολύτως απαραίτητο να εναρμονιστούν οι νομοθεσίες και όσον αφορά την εναρμόνιση σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα έχουμε πετύχει πάρα πολλά. Νομίζω λοιπόν ότι στα κράτη-μέλη έχει επιτευχθεί συμφωνία ότι αντί να εστιάσουμε σε νομοθετικές εξελίξεις θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στην ανταλλαγή πληροφοριών. Αν θέλετε αυτό είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει για την παράνομη μετανάστευση. Εκεί στηρίζουμε τις χώρες οποτεδήποτε μας το ζητάνε και αυτό ίσως και να έχει σχέση με την ανταλλαγή ή αν θέλετε και με τον συντονισμό των πληροφοριών ε, σε γενικές γραμμές, πάντως υπάρχει το πλαίσιο. Βεβαίως ε, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τον ε, αριθμό των περιπτώσεων που φτάνουν σε μας. Αυτό είναι γεγονός. Και τέλος, ε, μια άλλη τελευταία ερώτηση έχει σχέση ε, με τη συνεργασία με τη Λιβύη. Δηλαδή, τι είδους ε, συνεργασία έχουμε με τη Λιβύη. Ξέρετε, αυτή η συνεργασία είναι τόσο στρατηγικής όσο και επιχειρησιακής φύσεως και έχει εκφραστεί επανειλημμένα το αίτημα να βοηθήσουμε τη Λιβύη σε περιπτώσεις παράνομης ε, μετανάστευσης. Σε στρατηγικούς τομείς ε, θέλουμε να υπάρχει μια ε, σταθερή συνεργασία και γι' αυτό στηρίζουμε το πρόγραμμα Euromed Δικαιοσύνη. Εκεί η Λιβύη έχει προσχωρήσει στο πρόγραμμα αυτό και η μεγάλη πρόκληση σε σχέση με τη Λιβύη είναι να βρει εκεί κανείς τις κατάλληλες, τις αρμόδιες αρχές για να συνεργαστεί μαζί τους. Ο πρόεδρος. Μαρία Κριστίν ε, Βεξιά, δεν έχουμε χρόνο. Θα σας απαντήσει γραπτό. Σας άκουσε. Το είπα στην αρχή και ε, συμφώνησε. Ευχαριστώ πολύ. Σημειώνουμε τα δημοσιονομικά και σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να έρθετε λίγο πιο κοντά. Ε, θεωρητικά, όχι, πολιτικά, δεν το εννοώ έτσι. Um, okay. Um, um, λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Συνήθως, συνήθω, 11.30 έχει πάει η ώρα. Χωρί εισαγωγέ, θέλω να πω ότι είναι η τελευταία φορά που έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Επίτροπο. Προφανέ τελειώνει η θητεία, αλλά έπρεπε να το πω σε περίπτωση που δεν το ξέρατε. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, βέβαια. Όχι. Πώς να το πω τώρα. Σκεφτείτε προσεκτικά ποια είναι τα κρίσιμα θέματα που θέλετε να ρωτήσετε τον κύριο Επίτροπο την τελευταία φορά που τον ε, βλέπουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Πέντε χρόνια. Πώς περάσαν έτσι. Δεν ξέρω, εμεί τα νιώθουμε σαν 25 χρόνια. Εσεί στην Κομισιόν ένα αιώνα για το θέμα αυτό, το συγκεκριμένο. Τώρα στην Επιτροπή Γεωργίας μπορεί να ήταν ε, δύο χρόνια για μας και τέσσερα για σας. Αλλά για τα δικά μας θέματα μπορεί να μας έχουν φανεί και 25 χρόνια. Έχω χάσει το μέτρημα, λέει ο Επίτροπος. Νομίζω χθες, λες και ήταν χθες που ήρθα για πρώτη φορά. Ναι, έτσι το βλέπετε εσείς. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Νιώθω σαν να έχουν περάσει 25 χρόνια, τουλάχιστον. Δεν πιστεύω ότι ήταν μέσα σε πέντε χρόνια τόσο έντονα αυτά που ζήσαμε. Λοιπόν, ήταν πάρα πολλά τα θέματα, δεν θέλω να τα παριθμίσω. Σε εσά ο λόγο, Επίτροπε, για να μα πείτε ό,τι θέλετε στην τελευταία σα εμφάνιση εδώ, πριν τελειώσει η θητεία μα, στην Επιτροπή Ελευθεριών. Ευχαριστώ πολύ και την ομάδα σα και όλου και τη Σοφία και όλου του συνεργάτε, σε περίπτωση που δεν έχουμε στο τέλο χρόνο να αναφερθούμε σε αυτό. Άρα έχετε ζήσει περισσότερα χρόνια από μένα. Τουλάχιστον αυτό νιώθω, λέει ο κύριο Μωράε. Ευχαριστώ, αγαπητέ Κλοντ, αγαπητέ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Πραγματικά είναι η τελευταία φορά που έρχομαι εδώ, τα τελευταία 4,5 χρόνια. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που έχουμε να τα ξαναπούμε πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται για να έρθω σήμερα. Πριν από πέντε σχεδόν χρόνια, όπως είπε προηγουμένως ο Κλοντ, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2014 είχαμε την πρώτη μας ανταλλαγή απόψεων. Δεν ήταν απλή ανταλλαγή απόψεων, ήταν κάτι περισσότερο. Αισθάνθηκα πραγματικά ότι έδινε εξετάσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την εμπιστοσύνη ε, ε, που εναποθέσετε στο πρόσωπό μου και είναι το σημαντικότερο ε, στη σχέση μας. Για την εμπιστοσύνη τότε στην ακρόαση επιβεβαίωσης αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας. Χάρη στην ισχυρή συνεργασία μας επιτύχαμε πολλά και στα θέματα της μετανάστευσης και της ασφάλειας παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίσαμε τεράστιες προκλήσεις τις οποίες όλοι γνωρίζουμε μια πρωτοφανής ε, μεταναστευτική ροή, ένα ρεύμα και μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων. Ε, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, ούτε συμφωνούσαμε πάντα για όλα. Το 2014 μου είχαν πει ότι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ είναι η πιο δύσκολη επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά κάποιο τρόπο είναι σωστό αυτό. Εσεί είστε η Επιτροπή εκείνη που ασχολείται με τα θέματα που βλέπουμε σήμερα να καθορίζουν ε, τις συζητήσεις για τις ευρωπαϊκές εκλογές. Μετανάστευση και ασφάλεια είναι θέματα κατεξοχήν πολιτικά, εξορισμού πολιτικά τα οποία τα κράτη-μέλη για πολύ καιρό θεωρούσαν ότι αξίζουν μόνο εθνικές λύσεις. Θα πρέπει κανείς να αναγνωρίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν έβλεπε πέρα από τα σιλό και θεωρούσε ότι ε, χρειαζόντουσαν μακροπρόθεσμες συνολικές ε, στρατηγικές. Σίγουρα είναι απαιτητική η Επιτροπή σας και καλά κάνει και δίκιο έχει. Εγώ ανέκαθεν ε, ένιωθα την υποστήριξή σας στην ανάπτυξη αυτών των συνολικών πολιτικών για τις οποίες πάντα ήταν έμπνευση η θεώρηση του Κοινοβουλίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για το δικό σας έργο. Όλοι συνεισφέρατε στο να καταλήξουν σημαντικά νομοθετήματα σε χρόνο ρεκόρ και ε, πολλές φορές με παράλληλες εργασίες για διάφορα θέματα. Παράδειγμα, το πιο πρόσφατο, την περασμένη εβδομάδα, μόλις σε 7 μήνες καταφέραμε να συμφωνήσουμε για να ενισχύσουμε ε, με 10.000 ε, υπαλλήλους το Frontex και να δώσουμε και ισχυρές και πραγματικές εξουσίες για να υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη, ανταποκρινόμενοι στο λόγο μας και στις υποσχέσεις μας. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω το σύνολο της Επιτροπής σας και ιδιαίτερα τη Ρομπέρτα Μετζόλα και την ομάδα της και τους και για τις προσπάθειές σας αυτές προσβλέπω στην ε, ψηφοφορία σήμερα για να επιβεβαιώσετε το συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολλά επιτεύγματα και έχουμε χαράξει ένα χάρτη πολιτικής για τα επόμενα έτη και για την πολιτική της μετανάστευσης και για την πολιτική ασφαλείας. Θα ήθελα όμως να ξεκαθαρίσω ότι απομένουν ακόμα πάρα πολλά να γίνουν ε, συγκεκριμένα να εφαρμοστούν πλήρω όλα τα νομοθετικά κείμενα που έχουν εγκριθεί. Οι κοινέ μας προσπάθειες επικεντρώθηκαν στο να βρούμε ε, τις καλύτερες και βιώσιμες δυνατές λύσεις βάσει των αρχών της ευθύνη και της αλληλεγγύη, που είναι πραγματικά στην καρδιά των ευρωπαϊκών μας αξιών. Και εσεί είστε οι βασικοί υπερασπιστές των αξιών αυτών. Προτείναμε και άμεσες λύσεις και πιο μακροπρόθεσμες για τη μετανάστευση ε, σε όλες τις πτυχές, εσωτερικές και εξωτερικές, με ένα πάρα πολύ ειδικό στόχο. Συγκεκριμένα, να απαντούμε εγκαίρως και αποτελεσματικά στις κρίσεις. Μια προσέγγιση ισορροπημένη που κάλυπτε όλες τις πτυχές της μετανάστευσης να σώσουμε ζωές. Πάνω από 700.000 ζωές σώθηκαν στη Μεσόγειο από το 2015. Υποστήριξη των κρατών της πρώτης γραμμής στην υποδοχή ε, των μεταναστών με το σωστό τρόπο. Από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε τα κράτη-μέλη όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Μάλτα υποστηρίζοντας ε, με επιτόπου βοήθεια οικονομική, επιχειρησιακή και ε, πόρους. Κάναμε τη μετεκατάσταση και την επανεκατάσταση πραγματικότητα. Πάνω από 34.000 άνθρωποι που χρειάζονταν διεθνή προστασία μετεκαταστάθηκαν από την Ελλάδα και την Ιταλία. Και πάνω από 50.000 ε, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βρήκαν μια νέα αιστεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 μειώνουμε τα κίνητρα για την ε, παράνομη μετανάστευση ε, με συντονισμό και με διάλυση ε, δικτύων λάθροδιακινητών. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων μας εξασφαλίζοντας ότι οι καλόπιστοι ταξιδιώτες δεν παρεμποδίζονται στη μετακίνησή τους. Και βεβαίως με μια πολύ ισχυρή κοινή πολιτική ασύλου ε, για την νόμιμη μετανάστευση και ένταξη στην κοινωνία. Σε αυτά τα θέματα θα επανέλθω στη συνέχεια. Αυτό που μπορώ να σας πω τώρα είναι ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Σήμερα έχουν υποχωρήσει σε επίπεδα πριν της κρίσης και χαμηλότερα οι αφήξεις. 100.000 150.000 ήταν οι αυξήσει. 90% χαμηλότερε από το 2015, το 2018. Το 2019 εξακολουθεί η μείωση. Η ε, δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας οδήγησε ε, σε ήπια μείωση, ειδικά ε, στην Ανατολική Μεσόδιο και την αντίστοιχη οδό. Με τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία ε, στηρίζουμε ε, την υποδοχή τους εκεί. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των κοινών δράσεων των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα ουσιαστικό στοιχείο της πολιτικής μας για τη μετανάστευση ήταν η ενίσχυση των ομίμων οδών για να αποθαρρυνθεί ε, η χρήση παρανόμων οδών και να σπάσει το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών. Και δημιουργούμε τις βάσεις για μια μετανάστευση νόμιμη που να βασίζεται στις ανάγκες της αγοράς. Δυστυχώς έχει αποτελματωθεί το ζήτημα της γαλάζιας κάρτας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Κλοντ Μωράης για τις προσπάθειές του. Υποστηρίζεται πλήρως τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει η ελκυστική Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Είμαι βέβαιο ότι και το επόμενο κοινοβούλιο θα διατηρήσει το υψηλό επίπεδο φιλοδοξία για την νόμιμη μετανάστευση. Μόλι σα παρουσιάστηκε ε, ε, ο έλεγχο καταλληλότητα για την νόμιμη μετανάστευση. Πραγματικά οι κανόνε μας είναι κατάλληλοι για το σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί. Βεβαίω βελτιώσει πάντα χωρούν και μπορούμε να ε, κανονίσουμε καλύτερα τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όσους έρχονται εδώ για σπουδές, εργασία ή για οικογενειακούς λόγους. Και αυτό μάλιστα είναι προς το συμφέρον όλων μας. Ένα κεντρικό ε, σημείο της πολιτικής μας ήταν πάντα οι διεθνείς συνεργασίες και συνέργειες. Χαίρομαι πολύ που έχουμε πολλά πιλωτικά προγράμματα για την εργασιακή μετανάστευση με χώρες εταίρους ε, σημαντικές και αυτό έρχεται να συμπληρωθεί και από το πλαίσιο εταιρική σχέση για τη μετανάστευση ε, που ε, εγγράφεται σε όλες τις συμφωνίες μας με τις ε, χώρες αυτές. Έρχομαι σε ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα των τελευταίων ετών να υπάρξει πραγματική αλλαγή για τη μετανάστευση με μια κοινή πολιτική και ένα κοινό μάλλον ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που ενέκρινε τη θέση του και για τα επτά νομοθετήματα που είναι τμήμα αυτής της συνολικής μεταρρύθμισης. Σε ευχαριστώ και για την προθυμία σας συνεργασία με το Συμβούλιο για τις διαπραγματεύσεις όλων μας των προτάσεων, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα σύστημα ασύλου κατάλληλο να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του μέλλοντος. Γνωρίζω ότι είναι ε, κοινή μας η ε, αποφασιστικότητα, αλλά και ε, η δυσφορία. Χρειάζεται να κάνουμε προσπάθειες. Εγώ θα έχω αυτό το θέμα ψηλά στις προτεραιότητές μου μέχρι το τέλος της θητείας μου. Θα συνεχίσω να εργάζομαι με τα κράτη-μέλη για να σημειώσουμε πρόοδο του επόμενου μήνε, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε με το επόμενο κοινοβούλιο ως μέρος αυτής της συνολικής πολιτικής. Επίσης, ε, λυπάμαι που δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε τους τρίμερες διαλόγους για την οδηγία περί επιστροφών πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Βάζουμε τη δυνατά μας να παρέμβουμε το συντομότερο δυνατόν για να αποτρέψουμε την παράτιμη μετανάστευση και να καταπολεμήσουμε τις αιτίε. Όμως, ε, στην περίπτωση που ένα άτομο μένει παράτυπα ε, σε ευρωπαϊκή επικράτεια θα πρέπει να επιστραφεί. Αυτό είναι κλειδί για την αξιοπιστία οποιασδήποτε ισορροπημένη πολιτική για τη μετανάστευση και για να διασφαλίσουμε την υποστήριξη των πολιτών μα. Τώρα, για να έρθω στι θεωρήσει. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσφατη συμφωνία για τον κώδικα θεωρήσεων. Ο Χουάν Φερνάντο Λόπε Αγγιλάρου, η και η ομάδα του, με του κοιόδης εισηγητέ. θα ήθελα να του ευχαριστήσω. Η νέα μα πολιτική για τι θεωρήσει ε, έχει διευκολύνει ε, τους πολίτες, πολίτες από τη Γεωργία και από άλλες χώρες μπορούν, και την Ουκρανία, μπορούν να ε, ταξιδέψουν τώρα χωρίς θεώρηση και αυτό ενδυναμώνει τους δεσμούς ε, μεταξύ των πολιτών. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ο χώρος Σέγγεν. Όπως επανειλημμένα έχουμε πει σε αυτή την αίθουσα, η Σέγγεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να είναι κάτι που δεν αλλάζει θα πρέπει να έχουμε σαφείς κανόνες για τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή. Η κυρία Φαγιών επιση είναι αποφασισμένη. Είμαι σιγουρο Το 2014, κατά τη διάρκεια τη ακρόασή μου, Σα ζήτησα να σκεφτούμε από κοινού το πώ θα δυναμώσουμε την ικανότητα ελέγχων στα σύνορά μα. Αυτό παραμένει μέρο ε, τη εργασία μα. Όπω έχω επαναλάβει η Ευρώπη ποτέ δεν θα είναι φρούριο, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ποιος περνά τα σύνορά μας. Τα εξωτερικά μας σύνορα είναι ο σύνδεσμος ε, μεταξύ ε, τη κοινή μα δουλειά για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Τώρα, χάρη σε αυτό το έργο, όλα τα άτομα στα εξωτερικά σύνορα υπόκεινται σε ελέγχου ε, μέσω προηγμένων συστημάτων πληροφοριών, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγεν, το ε, ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών ε, Έγκρισης Ταξιδίου και το σύστημα πρόσβασης. Εσείς έχετε παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις ορόσημας για τη διαλειτουργικότητα που θα συνδέσει όλα αυτά τα συστήματα. Είναι το τελευταίο επίτευγμα, το να σπάσουμε τα σιλό, το να κλείσουμε τα τυφλά σημεία. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας ε, στο βάκελο αυτό και κυρίως ευχαριστώ τους συζητητές Ελένης και Μελό και τους Κιώδης φυσικά. Τώρα, η αποτροπή τη ρίζοσπαστικοποίηση και η καταπολέμηση τη τρομοκρατία και offline και online ήταν στο επίκεντρο των πολιτικών μα. Για να διασφαλίσουμε ένα ασφαλέ επιγραμμικό περιβάλλον, προτείναμε νομοθεσία για να αφαιρέσουμε γρήγορα το δημοκρατικό περιεχόμενο επιγραμμικά. Τα πρόσφατε εξελίξει μα έδειξαν την σημασία του να αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Λυπάμαι που δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το φάκελο αυτό πριν από τις εκλογές. Είναι μια χαμένη ευκαιρία. Τώρα δεν θα αναφέρω μια μια την νομοθεσία που υιοθετήθηκε για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη σοβαρό έγκλημα και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, ναρκωτικά πολέμηση του τράφικινγκ. Είναι μη εξαντλητικό ο κατάλογος. Όλα αυτά τα ξέρουμε εδώ πολύ καλά. Αλλά θέλω να δράξω την ευκαιρία να σα ενημερώσω ότι έχουμε μία προκαταρκτή συμφωνία για τις διαπραγματεύσεις PNR με τον Καναδά σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Και θα σας ενημερώσουν οι συνεργάτες μου. Και Κάτι τελευταίο αλλά σημαντικό για τη χρηματοδότηση. Η Κομισιόν ε, πρότεινε να αυξηθεί η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για το 2021-2027 για τη μετανάστευση και το άσυλο, για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την ασφάλεια. Πρόκειται για ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα που θέλει να στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους φιλόδοξους ε, στόχους ε, με επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης. Πιστεύω ότι το επόμενο κοινοβούλιο θα διατηρήσει αυτό το υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, αυτέ είναι ορισμένε από τι συγκεκριμένε δράσει μα και επιτεύγματα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σα ευχαριστήσω όλου για την προσωπική σας δέσμευση, αποφασιστικότητα, για τα διαπραγματευτικά σα προσόντα δεξιότητε ε, και τι προσπαθίε. σα. Θα μπορούσα να αναφέρω ένα προ ένα του αλλά καταρχήν είστε πάρα πολλοί και δεύτερον οι εισηγητές δεν είναι οι μόνοι που έχουν συνεισφέρει στο να επιτευχθεί αυτή η τεράστια δουλειά. Υπήρξαν ε, και πάρα πολύ σημαντικές για κάθε φάκελο ομάδε σκιώδων εισηγητών και όλα τα μέλη αυτής της ε, Επιτροπής. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που συζητήσατε και ψηφίσατε αυτούς τους φακέλους. Επίσης, ευχαριστώ και τους βοηθούς σας, τους πολιτικούς σας συμβούλους και τη γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. καθώς είναι καθοριστικός ο ρόλος σε κάθε επιτυχία. Όπως σας είπα, θα θέλω να συνεχίσω το έργο για να ολοκληρώσουμε του φακελού που έχουμε ακόμα επιτάπητο. Ξέρω ότι ορισμένοι από εσά θα επιστρέψουν μετά τι εκλογέ και θα ήθελα να σα ε, καλωσορίσω εκ νέου για να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο μαζί. Λυπάμαι πολύ που κάποιοι αποφάσισαν να μην επιστρέψουν γιατί η εμπειρία σα είναι πολύτιμη και είμαι σίγουρο ότι θα τη χρησιμοποιήσετε στην υπηρεσία τη Ευρώπη, του κοινού μας οίκου. Είμαι σίγουρο ότι θα ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μα με πολλού από εσά και έχω κάτι σημαντικό, προσωπικά σημαντικό να πω στο τέλος που προέρχεται από την καρδιά μου. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Κλωτ Μωράη, τον πρόεδρο τη Επιτροπή. Ήταν μεγάλη μου τιμή και ήμουν τυχερό να συνεργαστώ με ένα πρόεδρο της Επιτροπής του Βεληνικού του. Κλοντ, είσαι ένας ε, από τους ε, καλύτερους πολιτικούς στην Ευρώπη. Είσαι αποτελεσματικός, δεσμευμένος και έμπειρο νομοθέτης. Όταν θα λάβει η χώρα το Brexit, θα... η Ευρώπη θα τις λείψει της Ευρώπης και της επιτροπή αυτής θα τις λείψει. Και προσωπικά θα μου λείψει να εργάζομαι μαζί σου με αυτόν τον δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Σε ευχαριστώ που ήσουν ε, πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Σε ευχαριστώ για την υποστήριξή σου και για τη φιλία σου. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είχαμε μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα, ακόμα δεν έχουμε και το Brexit. Ίσως λοιπόν να είμαι εγώ ένας από εκείνους που θα επανέλθει ε, δεν μπορώ να κάνω καμία επιλογή, στην ε, χώρα μου επικρατεί μια αναστάτωση. Τέλος πάντων, ποτέ δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Πριν λοιπόν ε, περάσουμε ε, στα θέματα που αφορούν τα τελευταία πέντε χρόνια. Εσείς αναφερθήκατε πραγματικά χάρη στους και ηγητές. Βλέπετε το πόσο εξαντλημένο είναι το προσωπικό και τα μέλη μας. Πραγματικά αυτό είναι κάτι συνηθισμένο σε μας. Πολύ εξαντλημένοι όλοι. Γιατί είναι πάρα πολλέ οι νομοθετικέ διατάξει που περνάνε από αυτή την Επιτροπή. Όποιο είναι αντικειμενικό ε, ξέρει πολύ καλά ότι αυτό δεν συμβαίνει σε καμία άλλη Επιτροπή. Ένα τόσο τεράστιο νομοθετικό έργο. Κάποιο λοιπόν πρέπει να ασχοληθεί με αυτό και το κάνουν οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ. Δεν είναι αυτοί που ασχολούνται με τον προπολογισμό. Εχθέ στη συνεδρίαση για τον προπολογισμό πάρα πολλά δικά μα συζητήθηκαν και επιπλέον ε, και το άρθρο 7 παραδείγματος χάρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα άρθρο που έχει μεγάλη συναισθηματική φόρτιση για τα μέλη μας αλλά και για τους συνεργάτες. Πριν αρχίζουν πολύ να ρωτάνε για το τι κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε, θέλω να πω ότι η Επιτροπή αυτή ήταν μοναδική. Αναφερθήκατε ε, στα θέματα, στο Συμβούλιο, στο χρόνο, ασκήσατε κριτική. Ε, οι άνθρωποι αυτοί εδώ που βρίσκονται εδώ ασχολήθηκαν και με το PNR που είναι ένα ιστορικό θέμα που εξετάσαμε στην Επιτροπή μας. Ή έχουμε εδώ ανθρώπους που διαπραγματεύτηκαν τεράστια θέματα σχεδόν στο διάλειμμα τους το μεσημέρι. Εδώ είχαμε ένα σύμβουλο που ήταν έτοιμος να καταρρεύσει, εντάξει δεν τον αναφέρω για να μην τον ε, φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά να σας πω κάτι, αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε εμά. Τουλάχιστον πάνω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τα τελευταία πέντε χρόνια ε, έγινε καταπληκτική δουλειά και από εσά, Όλων αυτών τώρα λεχθέντων μπορείτε και εσείς ε, να κάνετε τα σχόλιά σας ε, για ό,τι επιθυμείτε. Βεβαίως και τα θέματα μας είναι πολιτικά και πολιτικά παραμένουν. Αρχίσω με την κυρία Χολμάιερ. Αν έχει την καλοσύνη ε, να είσαστε ακριβείς στα θέματά σας και λυπάμαι που ε, μακρηγόρησα. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα, ένα θερμό ευχαριστώ στον κύριο Επίτροπο, γιατί πραγματικά ήταν συνεχώς ε, πρόθυμος, ε, αδιάλειπτα πρόθυμος να έρχεται εδώ και να μας ε, απαντά στις ερωτήσεις μας. Επέδειξε και μεγάλο θάρρος. Τα θέματα δεν ήταν απλά, τα θέματα που χειρίστηκε. Είχαμε τα θέματα της ε, τρομοκρατίας, ε, του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, αυτά είναι θέματα με διεθνή διάσταση. Κατόπιν είχαμε το θέμα της μετανάστευσης των προσφύγων, το παράνομο εμπόριο ανθρώπινων όντων. Δεν είναι εύκολο να τα εξετάσει κανείς αυτά τα θέματα σε πέντε χρόνια. Μα 25 χρόνια δεν λύθηκαν αυτά τα θέματα. Δυστυχώς βέβαια σε κάποια θέματα υπάρχουν καθυστερήσεις. Γιατί αν δούμε το θέμα, το θέμα της χορήγησης ασύλου, εκεί υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Βέβαια υπάρχει και ο διχασμός στα κράτη-μέλη. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι στην επόμενη θητεία θα προχωρήσουμε περισσότερα θα επικρατήσει μεγαλύτερη συνένεση και συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Τουλάχιστον εγώ ε, δεν έχω παραιτηθεί από την ελπίδα. Ερωτήσεις τώρα συγκεκριμένα. Πρώτη ερώτηση. Αφορά τη νέα κατάσταση στη Frontex. Βλέπουμε ότι μεγαλώνει η Frontex τόσο όσον αφορά τις αρμοδιότητές της, όσο και όσον αφορά στο προσωπικό που θα απασχολεί. Κατόπιν τούτου, μιλάμε για περίπου 10.000 ε, συνεργάτες της Frontex, άνδρες και γυναίκες. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά και η δομή της Frontex. Εμένα λοιπόν αυτό με ενδιαφέρει, γιατί ξέρετε είναι κατελή διαφορετικό να έχω 500-600 ανθρώπους και κάποια στιγμή να φτάσω μέχρι και 10.000 μια τάξη μεγέθους ε, η οποία είναι ίσως ε, υπερβολική για έναν ε, τέτοιο εξωτερικό οργανισμό. Κανονικά τέτοιου είδους εξωτερικά γραφεία, εξωτερικοί οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν τέτοιες μεγάλες διαστάσεις. Με ενδιαφέρει λοιπόν στο μέλλον πώς θα είναι διαρθρωμένη Frontex, τι είδους δομή θα έχει. Αυτό ήταν το ένα ερώτημα, το πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο ερώτημα, το θέμα για τα εσωτερικά σύνορα. Εκεί είχαμε μία αποτυχία. Απέτυχε ο τριμερής διάλογος. Και ρωτώ, μήπως ε, στο μέλλον και από πλευράς κρατών μελών θα ήταν καλύτερα να δώσουν σημασία σε ευέλικτες ε, στιγμιές ή βραχυπρόθεσμες πράξεις. Γιατί σε τελική ανάλυση το όλο θέμα είναι διαχείριση κινδύνου. Αν πρόκειται για διεθνή εγκληματικότητα, ε, για μένα, ξέρετε, είναι το ίδιο σαν να γίνεται κάποιο έλεγχο μέσα στη Γερμανία, μέσα στη Γαλλία, μέσα στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η συνεργασία στα σύνορα για την αντιμετώπιση τη διεθνού εγκληματικότητα θα πρέπει να είναι κάτι αυτονόητο και όχι να αντιμετωπίζεται περιοριστικά. Γι' αυτό λοιπόν με ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκέφτεται να κάνει επί του θέματος αυτού. Πρόεδρος, αν έχει την καλοσύνη, δύο λεπτά ο καθένας ε, ε, να αναφέρετε τα βασικά σας θέματα, γιατί σήμερα όλοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Η Μπίργκιτ έχει το λόγο. Τώρα, ε, μετά από τρία λεπτά μίλησε η προαλήσασα, να δω εγώ τι θα κάνω. Μην ανησυχείτε. Θα αναφερθώ σε κάποιες εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Επίτροπος, ο οποίος είπε θέλουμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη στο να καλωσορίζουν τους ε, μετανάστες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να σας πω κάτι, εγώ δεν το πιστεύω πια. Δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη θα καλωσορίζουν μετανάστες. Ξέρετε κάτι, θα χαιρόντουσαν πάρα πολύ ε, και εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ τα κράτη-μέλη δεχόντουσαν ότι τέλος πάντων υπάρχει το θέμα της μετανάστευση, ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και δεν το βλέπουν το θέμα τελείως διαφορετικά. Εμένα με ενδιαφέρει και τι γίνεται με τα χρήματα. Πού πάνε τα λεφτά, στην Ουγγαρία ή ε, σε επαναπροωθήσεις στην Σάντα Μελία και αλλού. Κατανοώ βέβαια ότι ορισμένες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βρίσκονται ε, παγίδα όπως τα Βαλκάνια. Ξέρετε γιατί όμως, γιατί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι πρόθυμα να δεχτούν τους μετανάστες. Όσον αφορά την μπλε κάρτα, την επανεγκατάσταση ή μετεγκατάσταση και επαναπρόθεση, δεν είμαι πια αισιόδοξη. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν πολύ γρήγορα αποφάσεις όταν πρόκειται για τρομοκρατία και θέματα ασφάλειας, αλλά όταν πρόκειται για άλλα θέματα καθυστερούν, δεν αποφασίζουν. Και ξέρετε κάτι κύριε Επίτροπε, πριν έρθετε είχαμε πει σε ένα άλλο θέμα ότι η ανυπαρξία κοινή ευρωπαϊκής γραμμής τόσο όσον αφορά την νόμη μετανάστευση για πρόσφυγες όσο και όσον αφορά την νόμη μετανάστευση για ανθρώπους που αναζητούν μια καλύτερη ζωή αυτό είναι πρόβλημα γιατί κανείς εκτός αλλά ίσως και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν κατανοεί τις διάφορες δυνατότητες που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν για να να εισέλθει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με νόμιμο τρόπο. Να πω κάτι για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση με Τουρκία. Ξέρετε, αυτή δεν έγινε με τη συγκατάθεση και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγινε μόνο με τα κράτη-μέλη. Αυτή η συμφωνία δεν λειτουργεί. Στο μέλλον, λοιπόν, ελπίζω, αν θέλουμε να χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια, να γίνονται οι απαραίτητε συζητήσει και στου τρει ευρωπαϊκού θεσμού. Ή, αν θέλετε, τότε τα κράτη-μέλη να τα κάνουν μόνα του και να πληρώνουν κιόλα. Να πληρώνουν και να αναλαμβάνουν το βάρος αν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ναι, εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας έγινε πολλή δουλειά, κάναμε πάρα πολλά, εξακολουθούμε να προσβλέπουμε και σε άλλα στο μέλλον και εγώ το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα κατανοήσουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις και αν αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει στο μέλλον να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ε, τότε χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, περισσότερους κανόνε σε όλου του τομείς και θέλω να ελπίζω ότι το καλοκαίρι επιτέλους θα το καταλάβουν αυτό και τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ, Μπέρκετ. Η Ναταλή Γκρισμπέκ από τους Φιλελευθέρου έχει αποχωρήσει. Η Γιώτη της Αρχεντίνη. Α, όχι, έχουμε ECR. Ζητώ συγγνώμη. Χέλγα Στέβεν από τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Συγγνώμη, Χέλγα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμε Επίτροπε. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 2012 για μα κατά της Ιταλίας ήταν η υπόθεση, αποφάσισε ότι δεν μπορούν να γίνονται συλλογικές ε, απελάσεις και επιστροφές προς την τελευταία χώρα τράνσιτ. Αυτό σταμάτησε ως πρακτική και καταδικάστηκε η Ιταλία ε, διότι ε, παρακολουθούσε τα εξωτερικά σύνορα και τους έστειλε στη Λιβύη. Από τότε μπορούμε να μιλήσουμε για μια ευρωπαϊκή πολιτική ανοιχτών σύνορων όπως φτάνει σε ευρωπαϊκές ε, ακτές, προστατεύεται και παίρνει και χρήματα. Αυτό το έχουν καταλάβει πολλοί στην Αλοδαπή και το εκμεταλλεύονται οι λαθρέμποροι. Χάνονται λοιπόν ε, ανθρώπινες ζωές. Ε, η Τουρκία με τη συμφωνία της έχει αναλάβει την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων και μπορεί να μας εκβιάζει κιόλας. Και η Frontex ενισχύεται βέβαια, αλλά τι γίνεται ε, με την εφαρμογή όλων αυτών. Ε, δεν υπάρχει ισχυρή πολιτική για την προστασία των συνόρων. Συγκεκριμένη ερώτηση, κύριε Αφραμόπουλη. Σήμερα έχετε αναθέσει στις υπηρεσίες σας ε, να δουν τι γίνεται με τις επιχειρήσεις επιστροφών στη θάλασσα, όπως ίσχυαν πριν από το 2012 και τι γίνεται με την απόφαση ε, του δικαστηρίου που προανέφερα. Τι κάνατε συγκεκριμένα για να ε, αποφύγουμε ε, τις τρευλές συνέπειες αυτής της ακτιβιστικού τύπου απόφασης του δικαστηρίου που έχουμε τώρα μαζικές παράνομες διελεύσεις στα σύνορα. Και σε μια πρόσφατη πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρχε κάτι σχετικό. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαρχεντίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, για την επισκόπηση, για τις ευχαρισίε και πραγματικά αισθανόμαστε λίγο περίεργα τώρα που είναι η τελευταία συνεδρίαση. Ε, και συμφωνώ με τον Κλώτ Μωράες. Ε, δεν είναι λες και ήταν χθε, λες και ήταν πριν από 25 χρόνια. Αλλά ε, πολύ διαφορετικές είναι οι εκτιμήσεις που έχω εγώ για την παρελθούσα πενταετία. Ε, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίσαμε την μεταναστευτική κρίση. Ε, βασικά μια διαχείριση κάναμε, για να είμαστε ειλικρινείς. Μας ε, πληροφόρησαν για το fitness check, για τον έλεγχο καταλληλότητας για την νόμιμη μετανάστευση, που καταλήγει, λέει ότι είμαστε εντάξει και δεν χρειάζεται να αλλάξει νομοθεσία για να έρχονται περισσότεροι μετανάστες νόμιμα για λόγους εργασίας εννοώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τότε είμαι πραγματικά απογοητευμένη αν είναι αυτό το συμπέρασμα και η επιχειρηματολογία, αν θα φτάσουμε στην οδηγία επιστροφών που είμαι και εισηγήτρια. Τότε θα έλεγα ας μην αρχίσουμε καν να το συζητούμε, διότι δεν υπάρχει ανάγκη αναδιατύπωση της οδηγίας αυτής. Αυτό που χρειάζεται είναι τα κράτη-μέλη να την εφαρμόζουν. Και δεν μπορώ να συμφωνήσω ε, ότι είμαστε fit μετά από το fitness check αυτό. Γιατί τα κράτη-μέλη πρέπει να αλλάξουν τακτική και νοοτροπία. Για, ε, χρειάζονται νέα ε, νομοθεσία για να έρχονται νόμιμα. αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη είναι άτομα με χαμηλή μόρφωση και χαμηλή προσόντα που θα έχουν και χαμηλές αμοιβέ. για το PNR με τον Καναδά μιλήσατε για τη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Μήπως θα μπορούσατε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση. Είδαμε αυτή την επιστολή που έχει στείλει ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Διεύθυνσης ε, Home στο Διευθυντή του Frontex. Σήμερα το πρωί ζήτησε ένας συνάδελφος να δούμε αυτή την επιστολή για να ολοκληρωθεί η εικόνα ε, και γίνεται λόγος εκεί για τη συνεργασία Frontex με το κέντρο διάσωσης στη Λιβύη. Θα ήθελα να μάθω τι και πώς ισχύει εκεί. Το ρώτησα και χθε και η απάντηση του διευθυντού της Frontex ήταν ότι αν ένα αεροσκάφος της επιχείρησης Frontex δει ένα σκάφος που χρειάζεται βοήθεια ε, θα ενημερώνει τα διάφορα κέντρα και μεταξύ αυτό και το Λιβικό Κέντρο Διάσωσης. Βέβαια δεν υπάρχει επίσημη λέει, συνεργασία μεταξύ των Λιβικών αρχών και της Frontex. Αν όμως ενημερώνουμε και τη Λιβύη και την Τρίπολη, εγώ αυτό το θεωρώ συνεργασία και ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες. Ε, εκείνοι που διασώζονται από τους ε, Λίβιους επιστρέφουν στη Λιβύη και όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί. Θα μπορούσατε λίγο να μας διευκρινίσετε ποιο είναι το σημερινό καθεστώς σας παρακαλώ. Γιατί η Μεσόγειος αρχίζει να αδειάζει πάρα πολύ τώρα που κλείνει και η επιχείρηση Σοφία γιατί δεν έχει πια σκάφη και ε, η άλλη επιχείρηση είναι μόνο κοντά στις ευρωπαϊκές αρχές και αν ένα σκάφος της εμπορικής ναυτιλίας ε, θα αισθανόμουν πάρα πολύ ε, μόνο στην ε, Μεσόγειο. Δυστυχώ πρέπει να φύγω γιατί πρέπει να πάω να παρουσιάσω στην ΕΟΚΕ το θέμα μου. Είναι διάφοροι οι συναδελφοί που ήθελαν να θέσουν αυτό το θέμα σε σχέση με την επιστολή. μήπω η Κομισιόν θα μπορούσε να μα απαντήσει γι' αυτό. Και το άλλο θέμα αφορά το PNR, με συμφωνία με τον Καναδά θα έχουμε και μία συνάντηση στις 11 Απριλίου. Ίσως μπορούμε να περιμένουμε τότε για την απάντηση. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Έρνστ, παρακαλώ. Με ναι, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ και σένα, Κλοντ. Καλό είναι να συναντιόμαστε και ε, πραγματικά το αντέξαμε αυτό πολλές φορές παρόλο που διαφωνούμε και το γνωρίζει πολύ καλά ο κύριος Επίτροπος. Είναι γεγονός ότι είναι δύσκολη η Επιτροπή αυτή και καλά θα κάνει να παραμείνει δύσκολη. Αν κοιτάξει κανείς την τελευταία πενταετία οφείλει να ομολογήσει ότι σε ό,τι αφορά την πολιτική για τους πρόσφυγες και για τα κράτη-μέλη αποτύχαμε και στο ανθρωπιστικό σκέλος και στο σκέλος της ισορροπίας, εξισορρόπησης. Δεν πετύχαμε τίποτα. Εντάξει, προωθήσαμε το Frontex, θα το ψηφίσουμε αργότερα και το ξέρουμε. Από την άλλη όμως, σε αυτή την πενταετία, αν το δούμε σχετικά με την προηγούμενη πενταετία ή συγκριτικά με άλλες περιόδους και άλλες δεκαετίες, ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς θανάτους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο τώρα. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και με ανησυχεί και εμένα. Γιατί δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό. Ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, επί μία διετία σχεδόν να μας αφήνει μετέωρους σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα της Ένωσης που είναι η πολιτική ασύλου και μετανάστευσης. Αυτή η δέσμη για το άσυλο ε, γενικά να το παραγωνείς, να το κάνει στην άκρη. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά για το Frontex συμφωνίζουμε. Και μετά μπορεί να διαφωνήσουμε για το τι θα πληρώσουμε και πώς θα πληρωθεί. Ας είναι. Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει το ένα χωρίς το άλλο. Και για μένα είναι τελείως ασαφές για ποιο λόγο το πακέτο του ασύλου και γενικά δεν μπορεί να προχωρήσει. Γιατί δεν διαπραγματεύεστε μαζί μας. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε μια θετική απόφαση για το Δουβλίνο. Για να μην την χαρακτήσω και ιστορική, ας πούμε, αν θεωρήσουμε ότι ε, βοηθήσαμε ε, στη συμφωνία. Θα ήθελα να μας πείτε και για το Δουβλίνο κάποια πράγματα, σας παρακαλώ. Πού έχει κολλήσει, ε, είναι καινούργιοι λόγοι ή γνωστοί παλιοί. Και δύο μικρά ακόμα. Τα hot spot με ανησυχούν πάρα πολύ στην πατρίδα σας, κύριε Επιτροπέ. Είναι αφόρητες οι εικόνες που βλέπουμε από εκεί. Πρέπει να το αναφέρω. Για ποιο λόγο αρνείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φύγουν οι άνθρωποι από εκεί και να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα, να βρεθεί κάποια διαφορετική λύση. Τα νησιά έχουν ε, γεμίσει, αφόρητη είναι η κατάσταση. Ε, ε, δηλαδή και μόνο τις εικόνες να βλέπω εγώ παθαίνω. Πρέπει να ληφθεί μια απόφαση για να βελτιωθεί κάπως η κοινωνική κατάσταση, αν μη τι άλλο. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα τη γνώμη σας. Θεωρείτε θεμητό αυτό που γίνεται να προωθείτε η ποινικοποίηση των σκαφών διάσωσης από τη Μεσόγειο, που δεν λέγονται Frontex τα πλοία. Θέλω ε, πραγματικά να μου απαντήσετε, γιατί αυτό ενδιαφέρει και συγκινεί πολλούς ανθρώπους. Ο Πέτερ Νίντερμελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητώ συγγνώμη γιατί και εγώ πρέπει να φύγω για τη σάντση του προεδρίου. Πρώτα απ' όλα, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνατε τα τελευταία χρόνια. Εξεταστήκαμε, εξετάσαμε μαζί πάρα πολλά θέματα. Κάτι άλλο επιτρέψτε μου να πω. Εγώ είμαι ένας από τους ε, ευρωβουλευτές βουλευτές εκείνους οι οποίοι μετά τα πέντε χρόνια είναι πραγματικά απογοητευμένου. Γιατί το Κοινοβούλιο έκανε πάρα πολλά για να επιλύσει διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, όμως το Συμβούλιο δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Και πρέπει να πούμε με απόλυτη σαφήνεια ότι οι μετανάστες η μετανάστευση και οι πρόσφυγες έγινε πολιτικό θέμα σε πάρα πολλά κράτη-μέλη. Ε, τα κράτη-μέλη προσπαθούν να αντλήσουν από αυτό το θέμα πολιτικό κεφάλαιο ε, η μετανάστευση και οι πρόσφυγες προκαλούν ε, κηρύγματα μίσους. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για το μέλλον. Και το ερώτημα που θέλω να κάνω είναι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε κάποιο πρόγραμμα, σκέφτεστε κάτι. Πώς θα μπορέσετε να πείστε τα κράτη-μέλη να φτάσουν ε, σε επικοδομητικές λύσεις και όχι στο, στην υπόθαλψη, υποκίνηση ε, μίσους και στα κηρύγματα μίσους. Οποτεδήποτε λίγη γίνεται λόγος για μετανάστευση. Η κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για αυτή την τελευταία συνάντησή μας. Για μένα ε, είναι ευκαιρία η σημερινή για να ε, εκφράσω αμφιβολίες ε, που συνέχισαν να υπάρχουν τα τελευταία πέντε χρόνια. Πρόκειται για την συνέπεια και την ειλικρίνεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα μετανάστευσης. Και θα ήθελα να αναφερθώ στην επιστολή για την οποία έγινε λόγος ήδη πριν από μένα από την Διευθύντρια Παρασκευή Μίχου ε, την οποία έστειλε ε, στον ε, Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής. Μία επιστολή όπου ζητά την λειτουργία της ζώνης που έχει σχέση με τη Λιβύη. Γίνεται λόγος για την ακτοφυλακή της Λιβύης, την πολύ καλή δουλειά που κάνουν, ότι έχουν διασώσει άτομα και γίνεται λόγος για τη σωστή χρήση του προσωπικού στη Λιβύη, ότι είναι περισσότερο επαγγελματίες, ε, πιο χρήσιμοι. Παράλληλα λοιπόν με αυτή την επιστολή, η Νατάσα Μπερτό, εκπρόσωπος της Επιτροπής, μας είπε ότι η Λιβύη δεν είναι ασφαλής χώρα. Τώρα, ανάμεσα σε αυτή την επιστολή που σας ανέφερα και στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Προφανώς υπάρχει χάσμα. Προφανώς ε, αντιφάσκουν αυτές οι δύο τοποθετήσεις. Κατανοώ βέβαια ότι δεν είναι το ίδιο το να μιλάει κανείς ε, για ασφαλή ε, χώρα και για μια ζώνη ΣΑΡ, αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια οδηγία για τα κλειστά λιμάνια αυτή όμως η επιστολή της κυρίας Μιχού, Μιχού της κυρίας Παρασκευής Μιχού είναι μια ε, επιστολή που καταλήγει στο ότι το να επαναπροωθούνται άτομα στη Λιβύη αυτό είναι και νόμιμο και σκόπιμο. Σε μια παρεμφερή επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν θα τη διαβάσω τώρα, δεν υπάρχει ούτε μία λέξη που να αφορά στην κατάσταση των ε, μεταναστών ε, στους ε, καταβλισμούς. Καταλαβαίνετε πολύ καλά σε τι αναφέρομαι. Από το 16 τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλουν αυτή την κατάσταση και το έκαναν και τελευταία φορά τώρα το Μάρτι, πρόσφατα. Ως εκ τούτου, πώς είναι δυνατόν μία ζώνη ΣΑΡ για έρευνα και διάσωση ε, μπορεί να κρίνεται ικανοποιητική σε σχέση με τη Λιβύη. Από την άλλη όμως η Λιβύη να μην είναι ασφαλής χώρα. Τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να δημοσιοποιήσετε την επιστολή Φαμπρίς Λεζέρη που στάλει στην Επιτροπή μία επιστολή η οποία εκφράζει κάποιες ε, επιφυλάξεις και μια επιστολή στην οποία η κυρία Μίχου αποφάσισε να τοποθετηθεί με μια μακροσκελέστατη επιστολή. Ε, θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο πράγματι λάβατε αυτή την επιστολή από την κυρία Φαμπρίζ Λεζέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τσινίτσι. Ευχαριστώ Κλοντ. Εγώ θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Αβραμόπουλο για το έργο του όλα αυτά τα χρόνια που δεν ήταν και τόσο απλό και για το γεγονό ότι πάντοτε ερχόταν εδώ στην Επιτροπή μας σαν και είμαστε απαιτητικοί. Αλλά αυτό επειδή ασχολούμαστε με ιδιαίτερα ευαίσθητα και πολύπλοκα θύματα και ήταν και ιδιαίτερα επίκαιρα αυτά τα χρόνια. Τώρα, εγώ θα είχα πολλές ερωτήσεις ε, να σας θέσω αλλά θα ήθελα να πω ότι και εγώ έχω απογοητευτεί από τα αποτελέσματα τόσες δουλειά σε σχέση με το μεταναστευτικό. Δυστυχώς φάνηκε πλήρως το έλλειμμα αλληλεγγύης και ευθύνη από την πλευρά των ευρωπαϊκών χωρών. Και πραγματικά με προβληματίζει και σε σχέση με το πώς ε, θα διαμορφωθούν οι μελλοντικέ δράσει στο θέμα τη μετανάστευση. Μιλήσατε για συμφωνίε συνεργασία με τι τρίτε χώρε. Θέλω να σα ρωτήσω. Με ποιο τρόπο και μέσω ποιων διαδικασιών θα μπορέσουμε συγκεκριμένα να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες για να εγγυηθούμε πιο αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου, αλλά και κυρίως για να εγγυηθούμε την, ε, τον πλήρη και απόλυτο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κατόπιν. Μια ερώτηση που αναφέρεται σε ένα θέμα που ξέρετε ότι μου είναι πολύ οικείο, την προστασία των ανηλίκων και μιλώ εδώ για τους ε, ανήλικους μετανάστες. Εσείς... Μιλήσατε για τα θετικά αποτελέσματα της συμφωνίας με την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, Σύμφωνα με διάφορες πηγές, στα τρία χρόνια της συμφωνίας, εκατοντάδες ασυνόδευτοι ανήλικοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε μη αξιοπρεπείς συνθήκες ε, εκεί όπου τους έχουν υποδεκτεί. Και ήθελα να ρωτήσω πώς η Επιτροπή θα μπορέσει να υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στην περίπτωση αυτή, έτσι ώστε οι πιο ευάλωτοι μετανάστες, δηλαδή οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, να τοποθετηθούν σε κατάλληλε δομέ σύμφωνα με τι ανάγκε του και να έχουν και την απαραίτητη υποστήριξη. Αλλά σα ρωτώ και πιο γενικά. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διασφαλίσει στις χώρες πρώτη υποδοχή, την κατάλληλη υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο άφηξη των μεταναστών. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους πόρους, αλλά και στο είδος της πολιτικής που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί για να υποστηριχθούν οι χώρες πρώτης υποδοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Κύριε Επίτροπε. Συγγνώμη που εγκαταλείπει το κοινοβούλιο μετά από 15 χρόνια και το συζωγιό μου σε σχέση, η μου, σε σχέση με το τι έχει γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια στον τομέα αυτό είναι πολύ αρνητική. Θα ήθελα να δω την Κομισιόν να αποτελεί μεγαλύτερο θεματοφύλακα των συνθήκων και να θέτει τα κράτη-μέλη ενώπιον των ευθυνών τους. Και αυτό είναι απόλυτα σαφές στο ότι υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ καταπολέμησης ε, της τρομοκρατίας με το μεταναστευτικό. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια ρητορική μίσους που χρησιμοποιείται από τα κρατημέλη για να στιγματίσουν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Εξακολουθεί να υπάρχει φόβος στις κοινωνίες μας και πραγματικά αυτό έχει να κάνει με την καταστροφή της δημοκρατίας και των αξιών μας. Θα ήθελα η Κομισιόν να ήταν περισσότερο στην πρώτη γραμμή και να αντιμετωπίζει τα κράτη-μέλη. Σήμερα, μάλιστα, είδαμε κάποιον εκπροσωπή την Κομισιόν και συζητήσαμε το θέμα τη ποινικοποίηση των ΜΚΟ που σώζουν ζωέ στη Μεσόγειο. Και ήταν πολύ απογοητευτικό που είπε ο κύριο αυτό ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί η ποινικοποίηση το ΜΚΟ. Δεν είναι αυτό που περιμένουμε από την Κομισιόν, σα το λέω ειλικρινά. Ο κύριο Τζούρεκ. Ευχαριστώ πολύ. Το τέλος της θητείας ε, είναι μια εποχή ευχαριστειών αλλά και θεμελιωδών ερωτήσεων. Και μια θεμελιώδης ερώτηση είναι σε τι θα πρέπει να χρησιμεύσει η πολιτική στο μεταναστευτικό. Μερικές φορές ακούμε ότι θα πρέπει να χρησιμεύσει για να καλυφθούν τα δημογραφικά κενά στην αγορά εργασίας. Αυτό όμως ε, είναι και κοινικό. Γιατί εδώ θα πρέπει να θυμόμαστε και θέματα που έχουν να κάνουν και με τη γλώσσα. Η αγορά εργασίας αυτή καθ' αυτή δεν αρκεί ως δικαιολογία. Επίσης θα ήταν ε, κοινική δικαιολογία προς τις κυβερνήσεις μας. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα πρέπει να έχουμε νέες γενιές και αν ζούσαμε χωρί σύνορα, αυτό θα ήταν επίθεση στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί είναι τόσο φυσικό να έχει σύνορα, όπω είναι φυσικό να έχει σπίτι, να ελέγχει δηλαδή τον ε, ζωτικό σου χώρο και το να ελέγχει ε, τη ζωή σου είναι κάτι διαφορετικό. Και ακούσαμε δυστυχώ ε, σε αυτήν την επιτροπή ότι αν η μετανάστευση είναι ανθρώπινο δικαιώματα, τότε δεν υπάρχει και ο όρο παράνομη μετανάστευση. Όμως ε, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε με αυτή τη λογική καμία λογική πολιτική. Και κάτι ακόμα, ίσως σε έκτακτες περιπτώσεις ε, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας. Αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, αλλά ακόμη και έτσι δεν μπορούμε να προκαλούμε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, ε, γιατί μιλάμε μόνο για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Είναι κάτι συγκεκριμένο, κάτι ειδικό. αν ε, έχουμε σοβαρά μεταναστευτικά ζητήματα, μερικές ε, φορές είναι δύσκολο να ασχοληθούμε και με δύο περιπτώσεις που μπορεί να έχουμε σοβαρά ζητήματα και η πολιτική μας ε, δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Φαίνεται ότι θα πρέπει να εξυπηρετήσουμε το κοινό καλό, δηλαδή να φροντίζουμε το καλό του δικού μας έθνους και θα έπρεπε να είμαστε πολιτικά υπεύθυνοι. Κυρίες και κύριοι, ε, και εγώ είμαι στο τέλος της θητείας μου. Είμαι μέλος σε τρεις επιτροπές. Αυτή ήταν η τρίτη μου επιλογή, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όμως, νομίζω ότι πραγματικά εδώ έχουμε συζητήσει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και ευχαριστώ πολύ τον Κλώτ και όλους τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ. Δύο τελευταίοι μιλητές. Η κυρία Βερζιά και η κυρία Σλάιν. Σας παρακαλώ να είστε σύντομες ε, για να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Η Μαρή Κριστίν Βερζιά πρώτη παρακαλώ. Merci, Monsieur le Commissaire. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δεν ξέρω αν κάναμε καλή δουλειά Πάντως γεγονός είναι ότι από δουλειά δεν έλειπε η δουλειά. Είχα την ευτυχία να ζήσω δύο θητείες. Ε, ο απολογισμό δεν είναι καλός νομίζω. Αντίθετα με τα λεγόμενά σας, είναι σαφές ότι έχουμε ενισχύσει την Ευρώπη φρούριο, αλλά όχι για όλους. Έχουμε τα λόγια, έχουμε και τις πραγματικότητες. Όλο το σύστημα βασίζεται στους καλούς ε, μετανάστες και τους κακούς πρόσφυγες και όχι το αντίστροφο. Κάθε χρόνο έχουμε 2,5 εκατομμύρια μετανάστες που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 3 εκατομμύρια εκατό το 2017 η πρώτη εθνικότητα είναι οι Ουκρανοί, τους οποίους υποδέχονται οι Πολωνοί. Και αυτοί είναι οι καλοί οικονομικοί μετανάστες. Αυτά όλα μου φαίνονται πολύ κοινικά ακούγοντας διάφορα λεγόμενα. Σε ποιους κλείνουμε τις πόρτες τώρα και θα τις κλείνουμε όλο και πιο ερμητικά είναι οι πρόσφυγες. Αυτό που δεν λειτουργεί στην Ευρώπη είναι το καθεστώς ασύλου. Δεν υπάρχει καθεστώς ευρωπαϊκού ασύλου, ούτε πρόκειται να υπάρξει ευρωπαϊκό καθεστώς ασύλου όσο τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι θέλουν στο θέμα αυτό. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα. Ένα αριθμητικό στοιχείο να σας δώσω. 90% των ατόμων που δικαιούνται διεθνή προστασία και το τονίζω, διεθνή προστασία που δίνει τα κράτη-μέλη, αυτό δίνεται σε ανθρώπους που έρχονται στη Μεσόγειο ε, ε, με παράτυπα, ε, διασχίζοντας τη Μεσόγειο. Άρα υπάρχει πρόβλημα. Και γι' αυτό θέλαμε τις θεωρήσεις αυτές τις ανθρωπιστικές. Και όσα είδαμε τώρα με την επιχείρηση ε, τι ε, κανουμε UFORNAV βγάλαμε τα σκάφη για να μην έχουν ανταποκρίνονται στη διεθνή τους υποχρέωση αλλά έχουμε αεροσκάφη εγώ επίσης δεν θα είμαι υποψήφια και φεύγω έτσι με μια πικρία πρέπει να σας πω με μια πικρία διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν στο επίπεδο των προκλήσεων της παγκόσμιας κρίσης ε, γύρω από το προσφυγικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται, υποδέχεται ε, ένα πρόσφυγα ανά χίλιους κατοίκους και συνολικά 6% των προσφύγων παγκοσμίω. Κύριε Αβραμόπουλε, εγώ για αυτό το θέμα δεν μπορώ να σας δώσω συγχαρητήρια. Έλλη, παρακαλώ πάρα πολύ σύντομα. Κύριε Αγαπητέ Επίτροπε, δεν μπορώ να χάσω ίσως αυτή τη τελευταία ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία όλα αυτά τα έτη, αλλά και για να κάνω μια συνολική αποτίμηση. Ξεκίνησε η Κομισιόν ε, με πολύ ψηλή φιλοδοξία, με ευρωπαϊκό θεματολόγιο ε, για τη μετανάστευση που θα αντιμετώπιζε πλήρως το φαινόμενο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν συνεπής αυτό το χρόνια. Απλώς ε, σημείωνε τις διενέξεις μεταξύ των κράτων μελών και οι πολιτικές του Συμβουλίου και της Κομισιόν την τελευταία περίοδο επικεντρώθηκαν μόνο στην εξωτερική ανάθεση στη Μεσόγειο, στην Τουρκία, στη Βασνία και για την εσωτερική αλληλεγγύη ένα βήμα προς τα μπρος όπως και η κυρία Γκόμες εγώ θα ήθελα περισσότερο θάρρος από την πλευρά της Κομισιόν για να σέβεται περισσότερο τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις συνθήκες και ε, θα θέλαμε να συνεργαστείτε περισσότερο με το Κοινοβούλιο που έκανε το καθήκον του εγκρίνοντα όλα τα μέρη της μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Όμω κυρίως σας ρωτώ ποια θα είναι Ποιο θα είναι το πεπρωμένο του Δουβλίνου. Τα δύο τρίτα του Κοινοβουλίου έδωσαν ε, ισχυρό μήνυμα στι κυβερνήσει, εγκρίνοντα μια μεταρρύθμιση που ζητά σε όλε τι χώρε ε, να αναλάβουν τι ευθύνε του για την υποδοχή και ε, να αξιολογήσουν τι αιτήσει ασύλου. Γιατί στο Συμβούλιο Οι ίδιε πολιτικέ ομάδε και οι ίδιε εθνικότητε δεν μπόρεσαν να βρουν συμφωνία και πώ σκοπεύετε να δώσετε μια διαρθρωτική λύση στο θέμα των αφήξεων, αν πλέον δεν προωθήσετε την μεταρρύθμιση του Διβλίνου που είναι πραγματική υποκρισία και ο λόγος για τους οποίους κάποιε δειλέ κυβερνήσει μπλοκάνουν τα άτομα στη θάλασσα ακόμη και 20 ημέρε και μάλιστα και μέσα στα Χριστούγεννα. Μιλώ λοιπόν για temporary arrangement και πώ θα αιτιολογήσετε αυτό το νομικό παραδοξό ότι δεν αναγνωρίζετε ω ασφαλή λιμένα στη Λιβύη αλλά συνεχίζετε να υποστηρίζετε την Λιβική εκτεφυλακή που στέλνει τα άτομα σε αυτά τα κολαστήρια, στι φυλακέ. Πραγματικά εύχομαι να αλλάξετε πορεία. Πρόεδρος. Επίτροπε, ε, για τελευταία φορά λοιπόν σε αυτή τη θητεία μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Παρακαλώ. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και ακόμη και για τις επικρίσεις σας. Αλλά αναρωτιέμαι, κάποιοι ε, από εσά ε, ε, ξέρετε ποιος προσπάθησε και ποιος δεν βοηθούσε, ήμουν ξεκάθαρο στην αρχή. Χάρη σε εσάς κάναμε πολλά, σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα, αλλά κατανοώ και όλοι συμφωνούμε ότι δεν ε, δεχτήκαμε και τόση υποστήριξη, όχι από τα κρατημέλη, από κάποιες κυβερνήσεις των κρατών μελών. Δεν ήταν η κατάσταση πέντε χρόνια πριν όπως είναι σήμερα. Εν τω μεταξύ, πολιτικές αλλαγές σε πολλές χώρες οδήγησαν σε μια νέα στάση και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Να σας εξομολογηθώ κάτι. Όταν ήμουν εδώ πριν πέντε χρόνια, εγώ είχα την εντύπωση ως ε, υπουργός, ε, πρώην υπουργός, ότι ήταν ένα ισχυρό εκτελεστικό όργανο κομισιόν, όμως δεν ισχύει. Χάρη στη δική συνεργασία κάναμε κάτι, αλλά δεν υποστηριχτήκαμε και ιδιαίτερα από κάποιες κυβερνήσεις, κυρίως τα τελευταία δύο έτη. Έτσι λοιπόν, δεν είστε ικανοποιημένοι με τα όσα κάνατε. Παρακαλώ να είστε ειλικρινείς και να εκφράσετε τη δυσαρεσκιά σας σε αυτούς που την προκάλεσαν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σχεδόν σε όλα τα σχόλια, γιατί υπάρχουν κάποιοι κοινοί παρανομαστέ στι ερωτήσει που μου τέθηκαν. Όταν ε, υιοθετηθεί η ε, νομοθεσία για τη Frontex, η Ευρωπαϊκή Συνολική και Φυλακή, θα ξεκινήσει να λειτουργεί ο οργανισμός ε, για την κυρία Χολμαϊέρ, απαντώ, και θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει έτσι όπως αποφασίστηκε, ακόμη και αν θα χρειαστεί αναδιάρθρωση. Όμως ήταν μεγάλο επίτευγμα. Όπως είπα, λυπάμαι που οι διαπραγματεύσεις της ε, τροποποίησης του Συνοριακού Κώδικα Σέγγεν για την ε, προσωρινή επανεισαγωγή των ελέγχων στα σύνορα δεν υλοκρίθηκε από τη σημερινή θητεία του Κοινοβουλίου. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε δουλειά για το, για το φάκελο αυτό συγγνώμη, υπό τη Φιλανδική Προεδρία εν ώψη της ε, μελλοντικής επιβέωσης της θέσης του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση, όλες οι επιλογές παραμένουν ανοιχτέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά σύνορα, η Κομισιόν εκφράζει τη λύπη της που παρόλες τις προσπάθειες οι συνοριακοί έλεγχοι συνεχίζονται, εμένουν σε κάποια εσωτερικά σύνορα. Για να υπενθυμίσω η Κομισιόν ενθάρρυνε τα κράτη-μέλη να αναφερθούν ε, σε αναλογικούς ε, αστυνομικούς ελέγχους και συνεργασία ως ε, εναλλακτική λύση σε συνοριακού ελέγχου. Προτείναμε και αλλαγέ στου κανόνε για την προσωρινή επανεισαγωγή των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Η Κομισιόν θα συνεχίσει τις προσπάθειες να επανέλθει στη Σέγγεν όπως πριν, χωρίς να έχουμε εσωτερικούς ελέγχους. Όλες οι προσπαθίες μας για το μεταναστευτικό και για την ασφάλεια κατευθύνονται προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτήν την οδό. Κύριε Σίπελ. Ήταν ε, πολύ λογική η κριτική που κάνατε στα κρατημέλη. Το είπα και πριν. Αλλά όχι. Δεν θα δεχτώ να σταματήσω να προσπαθώ για μια πολιτική λύση. Πρέπει να ολοκληρώσουμε όλα τα τμήματα της πολιτικής μας και για τη μετανάστευση και για την ασφάλεια. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, κυρία Σιπέλ. Εδώ συμφωνούμε. Γιατί μην θα επανέλθω για περισσότερες πληροφορίες. Κυρία Στίβενς, για την Ευρωπαϊκή Φυλακή και Εκτοφυλακή. Θα διασφαλίσουμε ότι όλα γίνονται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό θα ενδυναμωθεί περαιτέρω με την νέα νομοθεσία. Κύριε Σερτζεντίνη. Αλλά δεν είναι εδώ. Και εγώ είπα ότι υπάρχουν τρόποι η νόμιμη μετανάστευση να βελτιωθεί για την PNR για τον Καναδά. Όπως είπα και το επιβεβαίωσε και ο Κλοντ, οι υπηρεσίε μου θα σας ενημερώσουν λεπτομερώς την επόμενη εβδομάδα κιόλα. Τώρα για την επιστολή. Αυτή η επιστολή δηλώνει το προφανές. Αποσαφηνίζει το επιχειρησιακό καθεστώς που ισχύει για τις επιχειρήσεις έρευνα και διάσωσης δυνάμει του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Είμαι σίγουρος ότι έχετε συζητήσει χθες τις λεπτομέρειες με τον εκτελεστικό διευθυντή του Frontex, τον κύριο Λετζέρη. Κύριε Έρνστ. Θα ήθελα ευχαρίστως να έχω μακρά πολιτική συζήτηση μαζί σας και τους συναδέλφους. Το Δουβλίνο θα πρέπει να υιοθετηθεί και Μετανάστευση και ασφάλεια δεν ε, θα πρέπει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης για μικροπολιτικούς σκοπούς. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση σε κάποια κεντρή υποδοχή, συμφωνώ με την απόψή σας ότι θα πρέπει η κατάσταση να σέβεται τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα ήθελα επίσης ε, να ευχαριστήσω τον Πίτερ για την εξαιρετική του δουλειά και για τη δέσμευσή του. Αλλά επίσης έφυγε. Κυρία Γκόμες, για τη ρητηρική μίσους και το στιγματισμό και το λογικισμό. Όλα αυτά όντως καταστρέφουν τη δημοκρατία και την υποσκάπτουν. Θα μας λείψει το πάθος σας, Και από την επόμενη θέση σα παρακαλώ να αγωνιστείτε για να δοθούν περισσότερε αρμοδιότητες στην Κομισιόν. Και κάτι σημαντικό που είπατε πολύ και η κυρία Τσινίτση. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην μεταναστευτική κρίση σε όλα τα επίπεδα. Η Κομισιόν επανειλημμένα υπενθύμησε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν σκοπεύει να ποινικοποιήσει την ανθρωπιστική βοήθεια. Η αξιολόγηση του πακέτου όσων υποβοηθούν που υιοθετήθηκε το 2017 από την Κομισιόν αποκάλυψε ότι υπάρχουν, έχει έλλειψη από των αποδείξεων για να νομοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, επίσης εντόπισε πιθανές βελτιώσεις, ιδίως ό,τι αφορά τη σαφήνεια της ε, ανθρωπιστικής ρήτρας εξαίρεσης ε, σε ό,τι αφορά την ε, μη ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Η Κομισιόν άρχισε να συζητά με προσώπους της κοινωνίας των πολιτών και με τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχαμε μια ειδική συνεδρία στο Μάιο του 2018 και συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τι οργανώσει κοινωνία των πολιτών ε, να μα κοινοποιούν οποιασδήποτε σχετικέ πληροφορίε. Κύριε Βερζιά. Όχι, δεν θα κλείσουμε τις πόρτες στους πρόσφυγες. Είμαστε ε, σε σχέση με την ε, επαναγκατάσταση. Σας δώσαμε αριθμητικά στοιχεία, αλλά όπως είπα ήδη, χρειάζεται να συμπληρώσουμε την πολιτική μας με την μεταρρύθμιση του ασύλου. Ακούω και είπα στην αρχή ότι άκουσα πάρα πολλές επικριτικές παρτηρήσεις που στρέφονται κυρίως κατά των κρατών μελών. Και πιστέψτε με, δεδομένης και της ε, πείρας που έχω συσσωρεύσει τα τελευταία χρόνια, Συμφωνώ με ορισμένε επικρίσει. Όμω να μην ξεχνάμε τι έχουμε πετύχει. Τι έχει επιτευχθεί από όλους μας και κυρίως μέσω της συνεργασίας Κομισιών και Κοινοβουλίου τα τελευταία χρόνια. Να μην ξεχνάμε πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση επιτόπου. Όλοι θυμόμαστε πώς ήταν ε, η κατάσταση πριν 4,5 χρόνια. Τώρα έχει αλλάξει. Σας ε, παρουσίασα πάρα πολλά στοιχεία και νούμερα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Ας μην ξεχνάμε ότι πολύ σοβαρή μεταναστευτική κρίση, κρίση ασφαλείας, ε, την χρησιμοποιήσαμε καταλητικά για να, χρησιμοποιήσουμε, για να θετήσουμε πολιτικές για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα και να διαχειριστεί οποιαδήποτε μελλοντική απειλή. Έτσι λοιπόν, στο μέλλον όλοι θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε μία κοινή ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Θα ήθελα να σας πω ότι όταν λέω ότι σας ευχαριστώ για τη συνεργασία μας, το εννοώ. Κατανοώ ότι υπάρχουν διάφορε ιδεολογικές προσεγγίσεις, όμως η πολιτική μας, η πολιτική μας βασίστηκε στο ρεαλισμό. Αν δεν είχαμε κάνει αυτά που ήδη πράξαμε, θα βρισκόμασταν ακόμη στην κατάσταση κρίσης, αλλά το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Αν οι προτάσεις μας είχαν υιοθετηθεί πλήρω και είχαν υποστηριχθεί από όλα τα κράτη-μέλη, η Ευρώπη θα ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη για το μέλλον. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, η μετανάστευση ήρθε για να μείνει για πολλά χρόνια. Και δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Και μάλιστα αυτό ήταν και ο σκοπό μα. Να εθετήσουμε μια μελλοντική, μια συγγνώμη στρατηγική που να μας προφυλάσει για το μέλλον. Ξέρω ότι η κατάσταση θα δυσκολέψει τα επόμενα χρόνια και δεν ξέρω το Κοινοβούλιο με τη νέα του μορφή αν θα είναι σε θέση να συνεργαστεί με τον ίδιο τρόπο σε ένα πνεύμα εμπιστοσύνη με τη νέα Κομισιόν. Έτσι λοιπόν, δέχομαι κάποιες από τις επικρίσεις σας στο ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα, όμως όσοι μας ε, έχουν ε, κατακρίνει θα μετανιώσουν στο μέλλον για το ότι αυτή η Κομισιόν δεν θα είναι εδώ. Θυμηθείτε τα λόγια μου, σας παρακαλώ, και βάλτε τη δυνατά σας για να υπερασπίσετε την πολιτική που όλοι και κυρίως να υπερασπίσετε τις αξίες και τις αρχές επάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η πολιτική μας. Ε, αυτή είναι η κοινή μας ευθύνη. Εμεί τα τελευταία πέντε χρόνια συνεργαστήκαμε σε ένα πνεύμα εμπιστοσύνη και η πολιτική μα βασιζόταν σε ελληνική και σε ευθύνη. Γιατί όλοι πιστεύουμε στι ίδιε αξίε και οι αξίες αυτές αυτή τη στιγμή διακυβεύονται και θα είναι ακόμη σε μεγαλύτερο κίνδυνο τα επόμενα έτη. Σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα και για όλα όσα κάνατε όλα αυτά τα έτη και ανυπομονώ να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί σα ε, όσο θα είστε εδώ για τους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Μπάρμπαρα Σπινέλη, ναι, ήθελα μόνο να πω ότι δεν πήρα απάντηση για το θέμα αν είναι ασφαλής χώρα η Λιβύη ε, για να αποβιβάζονται εκεί ή όχι. Ευχαριστώ. Θα σας πω. Πότε θα μου πείτε. Τώρα. Οκ. Okay. Ωραία. Πώς έχει η κατάσταση στη Λιβύη. Χάος, κυρία Σπινέλη μου. δεν έχουμε ισχυρή εταιρική σχέση με τη χώρα αυτή γιατί οι συνομιλητέ μας είναι πάρα πολύ αδύναμοι. Και χάρη στη βοήθεια της δικής σα χώρα, της Ιταλίας, καταφέραμε τουλάχιστον να συνεργαζόμαστε με την νόμιμη κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Η Λιβύη παραμένει ο παράδεισος των διακινητών και των λαθρεμπόρων και οι εικόνες που έρχονται από εκεί είναι όνειδος για όλους μας. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε εκείνο που της αναλογούσε. Συνεργαστήκαμε με πολύ αξιοπρεπή τρόπο με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Έχουμε επιτόπου δικούς μας άνθρωπες. Έχουμε εκπαιδεύσει την Λιβική ακτοφυλακή και πολλές ζωές έτσι έχουν σωθεί ως τώρα. Δυστυχώς όμως η κατάσταση παραμένει άσχημη. Αυτό πιστεύω εγώ. Ξέρετε ότι είμαι μεταξύ εκείνων που επισκέφθηκα την Τυρίπολη. Ευρωβουλευτή δεν είδα εκεί. Πηγαίνετε να δείτε πώς έχει κατάσταση στην Τρίπολη. Εκεί εστιάζουμε την προσοχή μας. Πώς να σώζουμε ζωές και πώς να ενθαρρύνουμε αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους να επιστρέφουν με τη δική μας ε, συνεργασία με γειτονικές χώρες. Ο Νίγηρας, για παράδειγμα, είναι μια πολύ καλή χώρα με την οποία συνεργαζόμαστε, αλλά ως Ιταλίδα εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα αυτά. Γιατί πάντα γνωρίζατε την κατάσταση στη Λιβύη τις τελευταίους τέσσερις αιώνες. Η δική μας προτεραιότητα είναι να σώσουμε ζωές και να προστατεύουμε εκείνους που ε, θέλουν προστασία, κυρίως οι πιο ευάλωτοι επιτόπου και να τους δίνουμε την απαραίτητη ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό το κάνουμε συνεργαζόμενοι με διεθνείς οργανισμούς. Είμαστε παρόντες, ξέρουμε πώς έχει η κατάσταση. Ας ε, ελπίσουμε να επανέλθει η ασφάλεια στη χώρα, γιατί όσο είναι ρευστή η κατάσταση, όπως είναι τώρα, και αυτό ξέρετε είναι ευθύνη της διεθνούς κοινότητας. Ε, αν ήταν δικό μας καθήκον ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα το είχαμε κάνει. Ε, αλλά η διεθνής κοινότητα φέρει μεγάλη ευθύνη απέναντι στη Λιβύη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέτρα που έχει στη θέση και τα μέσα. Κάτι λέει η κυρία Βερζιά. Κοιτάξτε, δεν θα το λύσουμε τώρα το Λιβικό, ε, αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μας όταν συζητούμε. Ο Πρόεδρος. Καλά, δεν θα ήταν σωστό τώρα να ε, τελειώσουμε με αυτό το τόσο επίμαχο και τόσο διχαστικό θέμα. Ωστόσο πρέπει να πω ότι η Μπάρμπαρα Σπινέλη που ε, μπορεί να έχει κάνει πολλά κακά, αλλά δεν φταίει και για 400 χρόνια ε, κατάσταση στη Λιβύη. Με φτάσουμε μέχρι τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχει κάνει και καλά. Λοιπόν, ε, ε ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα η Λιβύη. Όπως σας είπα προηγουμένως, σε προσωπικό επίπεδο και το ξέρετε πολύ καλύτερα. Ήταν μια πενταετία απίστευτη. Και να το πω ξεκάθαρα. Τα χειρότερα έρχονται. Ε, ξέρουμε μέσα μας όλοι προς τα που το πάνε τα κράτη-μέλη. Ε, το επενηχθήκατε. Επανέρχομαι σε προσωπικό επίπεδο θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτή τη συνεργασία. Ήταν μεγάλο το πολιτικό φάσμα ε, και ε, πολλά τα θέματα που αντιμετωπίσαμε. Και εσείς ως βασικός επίτροπος ε, ήσασταν πάντα εδώ πολύ συχνά. Τώρα φτάσαμε στο τέλος πέρα από τις πολιτικές συζητήσεις προφανείς που είχαμε, καμιά φορά σας άρεσε και όλα το το, το χαιρόσασταν μέσα σας, το διασκεδάζατε κρυφά και αυτό το διαπίστωσα και αυτό με ανησυχεί κιόλα. εντάξει, εσείς να έχετε το τελευταίο λόγο. Ε, πριν έρθω τώρα, ε, σήμερα εδώ, έριξα μια ματιά ε, στις απαντήσεις που σας έδωσα τα τελευταία πέντε χρόνια, μάλλον πριν από πέντε χρόνια στην ακρόασή μου και μπορώ να σας πω ότι ανταποκρίθηκα σε όλες μου τις δεσμεύσεις ε, και ε, στις υποχρεώσεις που είχα αναλάβει από την αρχική μου ακρόαση και τη σχέση με την αρχική μου παρουσίαση ενώπιόν σας. Άρα έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Φυσικά και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στο μέλλον, αλλά προτεραιότητά μας είναι να διαφυλάσσουμε και να διατηρούμε τις αρχές τις οποίες έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και πάλι και ιδιαίτερα ε, την ομάδα σας και ιδιαίτερα τη Σοφία και τους άλλους συναδέλφους. Ήταν ε, παλιά εδώ σε εμά στην Επιτροπή μας η Σοφία, τη γνώρισμα από ε, τον παλιό καιρό. Και πάλι όλοι είμαστε λίγο τσιτωμένοι. Ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείτε για το μέλλον. Στο καλό. we have um, just one more point. Um, Έχουμε άλλο ένα θέμα να συζητήσουμε, έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε γιατί αυτό το ζήτησαν και οι συντονιστές μας. Και ε, πρόκειται για την ανταλλαγή απόψεων με τον εκπρόσωπο της ε, εκστρατείας Time for Truth που λέγεται Kieran as Kieran comes up, just to explain that coordinators uh, decided that we would hear. Οι συντονιστές αποφάσισαν ε, να ακούσουμε τον ε, εκπρόσωπο αυτής της εκστρατείας ε, που ξεκίνησε στη Βορειολανδία και έχει σχέση με το πώς εξετάζεται το παρελθόν θα μας παρουσιάσει τις δραστηριότητες και τους στόχους. Λυπάμαι που καθυστερήσαμε. Αλλά ε, σας καλωσορίζουμε θερμά και παρακαλώ σας δίνω το λόγο για να κάνετε την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο και την Επιτροπή που με προσκαλέσατε σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Το εκτιμώ ιδιαίτερα και πράγματι αυτή είναι η ε, περίπτωση, είναι η ευκαιρία για να ζητήσουμε υποστήριξη για την εκστρατεία μας. Ε, θα συστηθώ ε, και μετά θα σας δείξω τις οικογένειες οι οποίες έχουν υποφέρει στη, από τη σύγκρουση με την Βόρεια Ιρλανδία και θα ήθελα να σας παρουσιάσω ε, το τι ακριβώς έγινε ε, στο παρελθόν στη Βορειολανδία και θα ήθελα να παρουσιάσω ε, τελευταίες περιπτώσεις νομικής φύσεως. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί βεβαίως και έχουν στυλιτεύσει την έλλειψη δραστηριοποίησης των Βρετανικών αρχών και νομίζω ότι θα πρέπει να απαντηθούν κάποιες ερωτήσεις που τίθενται από πλευρά οικογενειών. Είμαι ο κ. Μακάουτς, Είμαι ο εγγονός της Κάτλιν, η οποία είναι μία από εκείνες που σφαγιάστηκαν το 1971. Ο παππούς μου, Τζον, και αυτός ε, τραυματίστηκε σοβαρά, αλλά κατόρθωσε να ζήσει. Αυτή η σφαγή ήταν η μεγαλύτερη επίθεση που είχε γίνει ποτέ ε, εξαιρουμένη της επίσκεψης, ε, της επίθεσης ε, από τους Ναζί. Έσκασε μία βόμβα στο μπαρ και οι δράστες διέφυγαν. Άρα δηλαδή αυτοί που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα προσπάθησαν να ποινικοποιήσουν τα πάντα εμείς λοιπόν ως οικογένειες θελήσαμε να επιδείξουμε μεγάλη αξιοπρέπεια, ε, θελήσαμε να καθαρίσουμε το όνομά τους. Επίσης, εγώ είμαι μάνατζερ της, ε, ενός ε, ιδρύματος το οποίο χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θύματα της σύγκρουσης ανεξάρτητα από το παρελθόν τους. Και είμαι και επίσης εκπρόσωπος της εκστρατείας για την αλήθεια. Η εκστρατεία αυτή για την αλήθεια συστήθηκε από οικογένειες ε, οι οποίες κατά τη διάρκεια της ε, σύγκρουσης ε, υπέφεραν, αποφάσισαν να ενώσουν τη φωνή τους για να ακουστεί και ε, μας ένωσε η κοινή εμπειρία από το γεγονός ότι και το ίδιο το κράτος δεν μπόρεσε να εξετάσει το παρελθόν της Ιρλανδίας. Αυτό ισχύει και για τη Μεγάλη Βρετανία. Εμείς ε, δεν πιστεύουμε ότι το θέμα είναι να αποδίδονται ευθύνε. Αυτό που έχει σημασία είναι το τι πρέπει να κάνουν οι Βρετανικές αρχές για να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι ε, στους πολίτες. Όλοι είμαστε ίσοι κατ' ουσίαν απέναντι στον νόμο. Ε, όλοι μαζί είμαστε πιο ισχυροί Θέλουμε να αγωνιστούμε για τρεις βασικούς στόχους που αφορούν όλες τις οικογένειες που υπέφεραν από την σύγκρουση. Πρώτον, ζητάμε να εφαρμοστεί η συμφωνία που έχει συναπτεί για την αντιμετώπιση του παρελθόντος. Αυτό το έχουν δεχτεί ε, οι ενδιαφερόμενοι και στο Βορρά ε, και στη Μεγάλη Βρετανία ήδη από το 2014. Εν τω μεταξύ ζητάμε δεύτερον την σωστή χρηματοδότηση των ε, δικαστικών ε, διαμαχών, όπως αναφέρεται και στο δικαστικό πρόγραμμα των 5 ετών. Και το τρίτο που ζητάμε είναι ε, το να υπάρξει ένας διαμεσολαβητής. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι οικογένειες να ελπίζουν ότι ε, θα εφαρμοστεί πραγματικά η συμφωνία που έχει συναυτεί. Χρειάζονται βέβαια άλλα δύο χρόνια ε, για να λειτουργήσουν όλα σωστά, ακόμα και αν συσταθούν σήμερα. Η τοπική κοινωνία μας στηρίζει ανεπιφύλακτα το ε, Φεβρουάριο πάρα πολλοί άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους του Μπέλφαστ και από τη Βόρεια και από για τη δική μας την παρέλαση και οι δικές μας οικογένειες μπόρεσαν να συγκεντρώσουν 15.000 περίπου αντιδράσεις που αφορούν ακριβώς στην ε, κληρονομιά του παρελθόντος. Από το Σεπτέμβριο έχουμε συγκεντρώσει πάρα πολλές ε, υπογραφές ε, για να επιτύχουμε τους τρεις στόχους μας. Εξάλλου, θα οργανώσουμε και άλλη μια μαζική εκδήλωση επειδή οι Βρετανικές αρχές ε, δεν ενδίδουν. Με τη βοήθεια της Μαρτίνα Άντερσον, της Ευρωβουλευτίνας, ε, μια αντιπροσωπεία δική μας επισκέφθηκε τόσο τις Βρυξέλλες όσο και το Στρασβούργο για να ενημερώσουμε τους Ευρωβουλευτές και συναντηθήκαμε και με τον Επίτροπο, Ευρωπαϊκό Επίτροπο Ανθρωπίων Δικαιωμάτων. Εν τω μεταξύ πρέπει να σας πω ότι δεν έχει δώσει καμία επίσημη απάντηση από τις Βρετανικές αρχές. Ε, μου έχουν πει ότι την απάντηση αυτή ε, θα την είχαμε τον Ιανουάριο, αλλά την, την προηγούμενη εβδομάδα μας είπαν θα περάσουν ακόμα ε, κάποιες εβδομάδες ε, χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτή η ε, καθυστέρηση ε, προκύπτει από το ότι ο Κάρν Μπράντλι και ο Υπουργό Άμυνα Γουίλιαμσον έδωσαν ιδιαίτερη σημασία ε, σε αυτό το θέμα. Ο πρώτος αναφέρθηκε σε αυτό στο Κοινοβούλιο, είπε ότι ο κάθε ένας από αυτούς που έχει υποφέρει πέστη ένα έγκλημα, περίπου το 10% όμως ήταν ε, ε, άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούσαν με βάση εντολές ε, που είχαν λάβει. Αυτά όλα είναι ιδιαίτερα προσβλητικά και προκάλεσαν την οργή των οικογενειών που έχασαν και παιδιά, αλλά και εκείνους που δολοφονήθηκαν από πράκτορες του κράτους. Ε, όλα αυτά ήταν λάθος δηλώσεις. Ε, βεβαίως ανακλήθηκαν μετά από 24 ώρες, αλλά η ζημιά είχε γίνει. Και ο ε, πρόεδρος είπε τότε ότι θα προβλέψει τη σχετική νομοθεσία για να προστατεύεται, προστατεύονται οι άνδρες του στρατού σε παρεμβάσεις και στην Βορειολανδία αλλά και στο Αφγανιστάν και αλλού. Όλα αυτά έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο για την ε, διεκδίκηση τη δική μας ε, για την αλήθεια. Από τότε που οι άνθρωποι μας δολοφονήθηκαν από τον ε, Βρετανικό στρατό. Ήταν μια αιματηρή Κυριακή, μια σφαγή. Θα έπρεπε οι στρατιώτες να αντιμετωπίσουν την κατηγορία της δολοφονίας και μόνο ένας από 17 ε, σύρθηκε στα δικαστήρια. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η αμνηστία θα υπονομεύσει την πολιτική που ακολουθείτε. Τις τελευταίες 24 ώρες η κυβέρνηση μοιάζει να έχει ενδώσει, αλλά και πάλι η ζημιά έχει γίνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Υπουργών έχει ασκήσει κριτική για το ότι η Βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να μην εκπληρεί τις βασικές υποχρεώσεις για θέματα κληρονομιάς, ε, ηθικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι έρευνες ε, θα ε, πρέπει να συνεχιστούν. Η Επιτροπή εισακούστηκε και συμφωνήθηκε ότι τελικά αυτή η συμφωνία που είχε υπογραφεί ακόμα δεν εφαρμόζεται και είναι απαράδεκτο ότι εκατοντάδες οικογένειες ε, αντιμετωπίζουν όλη αυτή την καθυστέρηση. Δεν έχουν πρόσβαση σε ένα σύστημα το οποίο κατ' ουσίαν ερευνά και τους θανάτους. Οι εξελίξεις στις τελευταίες εβδομάδες κατέδειξαν ότι υπάρχει ανικανότητα ή και έλλειψη βούλησης για να εξεταστεί το παρελθόν της Βόρειας Ιρλανδίας. Έχουμε δύο πρόσφατες περιπτώσεις που δείχνουν ότι έχουν παραβιαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, υπολείπεται ακόμα μία αποτελεσματική έρευνα ε, και οι ε, εκπρόσωποι του κράτους βλέπουμε ότι τελικά δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις με βάση το άρθρο 2 όπου βλέπετε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή έρευνα αυτής της δολοφονίας που έγινε πριν από 30 χρόνια η οικογένεια του Τζιν Σμιθ Κάμπελ αποφάσισε να στραφεί κατά της αστυνομία στη Βόρεια Ελλανδία και να ξεκινήσει ε, περίφημη περίπτωση LIB. Η Τζιν ήταν ε, μια γυναίκα η οποία το 1972 δολοφονήθηκε. Η αστυνομία είπε στην οικογένειά της ότι δολοφονήθηκε από τον Ήρα. Στα αρχεία μας όμως διαπιστώσαμε, στα εθνικά μας αρχεία στο Λονδίνο, ότι δολοφονήθηκε κατ' ουσίαν από το Βρετανικό στρατό. Και ε, μάλιστα από μια ειδική μυστική υπηρεσία, ένα παρακλάδι μυστικής υπηρεσίας ε, το οποίο δραστηριοποιείται στις αρχές δεκαετίας του 70 στη Βόρεια Ιρλανδία. Το εφετείο του Belfast θεώρησε ότι δεν είμαστε ε, αμερόληπτοι ε, για να γίνει έρευνα για το φόνο, τη δολοφονία της Τζιν και ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτα τη τετραετία που ε, ε, η οικογένεια είχε προσφύγει. Ο αρχηγός της αστυνομίας τώρα ε, ζητεί μια ανεξάρτητη ομάδα να κάνει την έρευνα. Αυτό έχει μεγάλες επιπτώσεις σε πολλές υποθέσεις μας, πολλές από τις οικογένειές μας ποτέ δεν θεωρούσε ότι ήταν ανεξάρτητη αυτή η ε, Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρξει μια μονάδα ε, ανεξάρτητη διερεύνησης των ιστορικών δεδομένων με βάση τη συμφωνία του Stormont House. Ε, το PSNI μέχρι σήμερα ακολουθούν τη στρατηγική άρνησης θανάτου ε, αρνούνται ε, οποιαδήποτε ε, αρνητική δράση. Κάνουν παρελκυστικές κινήσεις για να μην προσφεύγουμε στην δικαιοσύνη και να μην δικαιωθούμε ποτέ και να μην επερτανεύσει ποτέ η αλήθεια. Ακόμα και τα αγγλικά δικαστήρια και ο διαμεσολαβητής της αστυνομίας καταγγέλουν ότι δεν ε, διαβιβάζουν τις πληροφορίες ε, οι Βρετανικές ένοπλες δυνάμεις για τον τρόπο όπου ενέχονται σε δεκάδες δολοφονιών ε, κάποιες μυστικές υπηρεσίες ήδη από το 1982. Στο Βρετανικό Υπουργείο Αμήνης υπάρχουν στοιχεία τα οποία όμως δεν ε, δημοσιεύονται και στο Derbyshire. Πέρσι το Φλεβάρι έγινε μια περίεργη πυρκαγιά, πιάσαν φωτιά κάτι στρατόπεδα στη Βορειοελλανδία και καταστράφηκαν αρχεία. Και υποτίθεται ότι η αστυνομία θα μας βοηθούσε, ε, αλλά ε, δεν εμπιστεύονται οι οικογένειες, ούτε την αστυνομία, ούτε κανέναν επίσημο φορέα. Για το λόγο αυτό τι ζητούμε και χρειαζόμαστε να εφαρμοστεί η συμφωνία του Stormont House και να επανέλθει η έρευνα ε, και ε, ο διαμεσολαβητής της αστυνομίας στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι οικογένειές μας είναι οι πρώτες ε, που πλήττονται γιατί δεν μπορεί το Βρετανικό κράτος να διαχειριστεί την κληρονομιά του παρελθόντος. Και μάλιστα πεθαίνουν και πολλοί χωρίς να δικαιωθούν ποτέ. Και βολεύει και ο θάνατός τους και το Βρετανικό κράτος και την αντίστοιχη πολιτική.